Στο όνομα του Ευρωκοινοβουλίου θέλω να σε λυπηθώ την οικογένεια και τους φίλους του Τζόρτζ Φλόιντ. Ο θάνατός του προκάλεσε τόσο στην ΣΥΠΑ αλλά και στην Ευρώπη πολλές διαμαρτυρίες που δείχνουν σε όλους πως ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των, και ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα καθήκον καθημερινό, ε, απαραίτητο και επιτακτικό. Μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι το όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ θα γίνει κάποια ημέρα των ημερών πραγματικότητα, που, ώστε οι άνθρωποι να μην κρίνονται ποτέ από το χρώμα της επιδερμίδας του, αλλά μόνο από το ε, χαρακτήρα τους ε, και τη συμπεριφορά τους. Εμείς πάντοτε καταδικάζουμε ως Κοινοβούλιο οποιαδήποτε είδος βίας, ε, και δεσμευόμαστε πάντοτε για τη στήριξη του κράτους δικαίου. Θα το συζητήσουμε και εδώ στην Ολομέλεια. και θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του George Floyd αλλά και όλων των θυμάτων βίας, ρατσισμού και διακρίσεων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. E Συνάδελφοι, ήθελα να σας θυμίσω πως η αίθουσα SPAC 3C50 είναι συνδεδεμένη με το ημικύκλιο ώστε να μπορέσουν οι βουλευτές που δεν θα βρουν θέση εδώ σε αυτή την αίθουσα της Ολομέλειας να μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες μας. Είναι οι ε, βουλευτές οι οποίοι είναι στον κατάλογο μιλητών και όταν θα χρειαστεί να μιλήσουν θα μπορέσουν να έρθουν εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας και θα βρουν τη θέση τους που θα είναι ε, σημασμένη με το όνομά τους και το επίθετό τους. Σας ενημερώνω ότι ο κατάλογος των παρουσιών βρίσκεται ε, μπροστά στην είσοδο και των δύο αιθουσών. Να σας θυμίσω ότι η χρήση των μασκών που καλύπτουν ε, μύτη και στόμα είναι υποχρεωτικές. Οι ομιλητές που θέλουν να μιλήσουν χωρίς την μάσκα μπορούν να το κάνουν μόνο για τη διάρκεια της ομιλίας τους. Θα ήθελα επίσης να καλέσω τους συναδέλφους να εισάγουν την κάρτα ψηφοφορίας ε, ε, ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε ότι ζητούν το λόγο επανακοινά η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ρουσούλα Βαντελάιν. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ε, κάποιος έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Η κυρία Ομπρί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου να πάρω το λόγο στην έναρξη της Ολομέλειας για να αναφερθώ στο ψήφισμα της ακροδεξιάς που κατετέθη στη συζήτηση που θα κάνουμε για το θάνατο του Τζόρτζ Φρόιτ που χειραγωγεί αυτό το θάνατο για να, για να κατηγορήσει τη δική μας ομάδα και τη Φράνσα να... ότι ενθαρρύνει και, και διαπράττει βίαιες ενέργειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι η δυσφήμιση είναι το σήμα κατατεθέν του Θέλουμε όμως εδώ να καταδικάσουμε και να βασιστούμε στη στήριξη της καταδίκης αυτής της ε, της ε, χειραγώγησης από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Η υπεροχή των Λευκών είναι αυτή που ε, ε, αναδύεται από αυτές τις δηλώσεις. Είμαστε περήφανοι εδώ γιατί εκπροσωπούμε αντιστασιακούς κομμουνιστές που έδωσαν τη ζωή τους ε, στη διάρκεια του πολέμου ενάντια στους Ναζί, ενώ οι δικοί σας βοήθησαν τους Ναζί. Τη βία της δεξιάς, η βία η αστυνομική την οποία εσείς συγκαλύπτετε, αυτή τη βία που εσείς συγκαλύπτετε όσον αφορά τις, τα διάφορα φασιστικά γκρουπούσκουλα. Εκεί που δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν υπάρχει ούτε ειρήνη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε κατά του ρατσισμού και εναντίον σα με ορίζοντα τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Τζαμπάσκη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο με βάση το άρθρο 1.7 και 1.7.1 το ε, εσωτερικό κανονισμού του Κοινοβουλίου. Πρέπει να αντισταθώ, να, μάλλον να διαμαρτυρηθώ για την κατανομή του χρόνου αγόρευση. Σημαντικέ συζητήσει, όπω το Brexit, οι μεταφορέ και άλλα ε, αδικούνται. Έχουν δοθεί εδώ πολλά λεφτά ομιλία για αυτό εδώ το θέμα. Αν εγώ έπρεπε να κατανείμω στου συναδέλφου μου το χρόνο αγόρευση θα είχαν 17 δευτερόλεπτα έκαστο. Είναι δική σας ε, αρμοδιότητα και καθήκον να ορίσετε το χρόνο έτσι ώστε κάθε μέλος του Κοινοβουλίου να μπορέσει να πάρει το λόγο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξέρω πως υπάρχει κόσμος εδώ που δεν θέλει να ακούσει ορισμένους συναδέλφους που δεν συμφωνεί μαζί μας. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να πάρουμε το λόγο και οι αριστεροί συνάδελφοι, οι αριστεριστές συνάδελφοι να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να ε, παίρνουν τον λόγο περισσότερο. Αυτό γίνεται με βάση τη συνεργασία των προέδρων των ομάδων. Président, je tiens tout d'abord Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους στην Ευρώπη εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους. Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω, καθώς και τους συναδέλφους, ότι εγώ ήμουν θύμα αστυνομικής βίας εδώ στο Βέλγιο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό αποτελεί πράξη, πράξη διάκρισης, ρατσιστική. Χθες, βγαίνοντας από το σταθμό του Βορρά, Gare du Nord, είδα δύο αστυνομικούς να κακοποιούν δύο νεαρούς μου και άρχισα να του μαγνητοσκοπώ με το βίντεο μου, κάτι το οποίο είναι νόμιμο. Οι αστυνομικοί κατευθύνθηκαν προς τα μένα, μου πήραν το τηλέφωνο από τα χέρια, τέσσερις από τους εννέα αστυνομικού οι οποίοι ήταν πάνω πλημέ έσπρωξαν στον τοίχο, μου πήραν την τσάντα, με κόλλησαν στον τοίχο, μου άνοιξαν τα πόδια και ένα αστυνομικό ε, με ψαχούλευε και με έψαχνε. Ήταν πραγματικά ατιμωτικό. Όταν είπα στον αστυνομικό ότι ήμουν ευρωβουλευτή, δεν με πίστεψε ενώ είχε στα χέρια του τα δύο διαβατηριά μου καθώς και το πάσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το γερμανικό διαβατήριο. Μου ζήτησε τότε την άδεια παραμονής μου στο Βέργιο Του έδειξα την, άδεια παραμονής, πήρα το badge ε, του Κοινοβουλίου. Σήμερα υπέβαλα μήνυση, διότι δεν μπορούμε αυτή την αστυνομική βία να την αφήνουμε ατιμόρυτη αυτή η εμπειρία τη στιγμή που ο κόσμος όλος βλέπει ποιες είναι οι επιπτώσεις της αστυνομικής βίας ήταν τραυματική για μένα. Όμως είμαι εδώ, παρότι πέρασα όλη τη νύχτα εδώ στο κοινοβούλιο, δεν είχα το κουράγιο να βγω μέχρι τις 6 το πρωί. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε μέτρα συγκεκριμένα για πολλούς ανθρώπους που δεν βρίσκονται εδώ και που δεν μπόρεσαν αυτοί να ξεφύγουν από την αστυνομική βία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Sì, Grazie, ευχαριστώ πολύ για, τα, για την κατάθεσή σας και βεβαίως ε, σας ε, παραστεκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας καλώ να έρθετε στο γραφείο μου να μου πείτε με λεπτομέρειες τι συνέβη και να ζητήσουμε μαζί διευκρινήσεις από τις βελγικές αρχές. Ναι, πιστεύω πως ε, οφείλουν εξηγήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ω επικεφαλή τη ομάδα των Πρασίνων, στην οποία ανήκει η κυρία Χερτσμπέργκερ, αλλά και ω απλό πολίτη του Βελγικού κράτου, θέλω πραγματικά να σα πω ότι είμαι ε, πραγματικά έκπληκτο με αυτό που συνέβη. Δεν έχει κάνει. Δεν έχει, δεν κανένα αδίκημα η κυρία Χερτσμπέργκερ. Και απλά τη επιτέθηκαν επειδή έπαιρνε φωτογραφία δύο. Πήρε φωτογραφία δύο αστυνομικού που ε, ήταν βίαιη απέναντι σε δύο νέου. Αυτό λοιπόν ε, συμβαίνει με την αστυνομική βία και αυτό συνέβη επί, λόγω του χρώματο τη συναδέλφου και το ξέρουμε αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι η δουλειά του αστυνομικού είναι δύσκολη, ότι είναι ε, απαιτητική. Ακριβώ όμω επειδή η αστυνομία είναι ένα βραχίωνα του κράτου, για να μπορέσει το κράτο να ασκήσει την νόμιμη βία τη οποία έχει το μονοπόλιο, όλοι όσοι φορούν αυτή τη στολή τη αστυνομία πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί να είναι μετρημένοι, διότι μόνο έτσι θα έχουν σεβασμό από εμά. Πρέπει οπωσδήποτε οι κοινωνίε να ξεσηκωθούν απέναντι στην αστυνομική βία, η οποία είναι όλο και πιο διευρυμένη. Ιδιαίτερα όταν αυτή είναι κατά των, των, έχρωμων και οποιοδήποτε γενικά ε, αντίθετη άποψη. Αυτά που συνέβησαν χθε είναι πραγματικά απαράδεκτα. ζητώ λοιπόν στο όνομα όλων να απευθυνθείτε στι βελγικέ αρχέ, να διαμαρτυρηθείτε και να ζητήσετε να, να χυθεί άπλετο φω απέναντι γύρω από την υπόθεση αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και ναι, δέχομαι αυτή την πρόταση που κάνατε. Τα πρακτικά της Συνόδου της 27 η Μαΐου είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσει Όχι. Οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Κάποιε ανακοινώσει μετά από την παρέτηση του κυρίου Κλάους Μπούκνερ, το Κοινοβούλιο με βάση τον κανονισμό διαπιστώνει την κένωση της θέσης του από τον 1η Ιουλίου 2020 και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Η ομάδα των Πρασίνων μου ανακοίνωσε την απόφασή της να τροποποιήσει τον διορισμό στις αντιπροσωπείες. Αυτή η απόφαση θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της Συνόδου και θα αρχίσει να ισχύει από τη σημερινή ανακοίνωση και στο εξή. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη κατάσταση τη επιμονή του COVID-19 και για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να ασκήσει τι λειτουργίε του μαζί με του Προέδρου των πολιτικών ομάδων σε συνεδρίαση των Προέδρων, της 5ης 28 Μαΐου αποφάσισα να παρατείνω τη σημερινή σύνοδο μέχρι την Παρασκευή 19 η ώρα, 7 η ώρα το απόγευμα και του Ιουλίου τη Σύνοδο από την Δετάρτη 8 το πρωί μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου το απόγευμα και θα βρείτε αυτές τις αλλαγές στον ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Επίσης, μέσω μιας τροποποίησης του κειμένου που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο, ε, σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 4 του ιστορικού κανονισμού του Κοινοβουλίου, θεωρείται ε, ότι εγκρίνεται εκτός κι αν εντός 24 ωρών μια πολιτική ομάδα ή μια, ένας αριθμός βουλευτών συγκεκριμένο ζητήσουν να ε, ψηφιστεί. Ε, και θα δημοσιευθεί η έγκριση στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού, η Επιτροπή Ήτρε αποφάσισε να ξεκινήσει διάφορες διαπραγματεύσεις διαθεσμικά πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου. Οι πέντε θέσεις που έχει υιοθετήσει το Ευρωκοινοβούλιο πριν από την πρώτη ανάγνωση που αποτελούν την εντολή για αυτές τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα και θα δημοσιευθούν και στα πρακτικά της σημερινής συνόδου. Η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών με ενημέρωσε ότι δεν έλαβε καμία αντίρρηση όσον αφορά τις συστάσεις των Επιτροπών Άγκρη και ΕΚΟΝ να μην αντιταχθούν σε κατεξοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 του κανονισμού. Οι συστάσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας ε, αν εντός 24 ώρων δεν εκδηλωθεί καμία πολιτική ομάδα ή αριθμός ε, ε, ευρωβουλευτών που χρειάζεται θα θεωρηθεί πως εγκρίνονται. Διαφορετικά θα ψηφιστούν, θα τεθούν μάλλον σε ψηφοφορία. Να σας ενημερώσω ότι την Πέμπτη θα υπογράψω με βάση το άρθρο 79 του κανονισμού του Κοινοβουλίου μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου τέσσερις πράξεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της νομοθε... τακτικής νομοθετικής διαδικασίας. Λεπτομερείς τίτλοι δημοσιεύονται στα πρακτικά τα σημερινά. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη των εργασιών. Οριστικό και η ημερήσια διάταξη ορίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων της 5ης 11 Ιουνίου, 11 Ιουνίου. Σύμφωνα με το άρθρο 157 και έχουν διανεμηθεί μάλλον η ημερήσια διάταξη έχει διανεμηθεί, έχουμε κάποιες τροποποιήσεις. Έλαβα τρία αιτήματα για εφαρμογή της διαδικασίας κατεπήγοντος με βάση το άρθρο 163 του κανονισμού για να προσθεθούν τα εξής νομοθετικά κείμενα που σχετίζονται με το COVID-19 και θα πρέπει να εγκριθούν στη διάρκεια της Συνόδου της 17ης και με 19η Ιουνία. Το ένα αφορά την διοικητική συνεργασία στον φορολογικό τομέα που έχει ε, ε, καθυστερήσει λόγω της πανδημίας. Έπειτα, εξαιρετική ε, κατάσταση στο πλαίσιο της πάλι για, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η τρίτη αφορά την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών για τα προσωρινά μέτρα όσον αφορά τι φάσει συλλογή, επαλήθευση, εξέταση των στοιχείων με βάση το COVID-19. Σας ενημερώνω ότι με βάση το άρθρο 200 παράγραφος 4 ο κανονισμός προβλέπει την ενημέρωση με βάση την έκθεση της κυρίας Ντέλη σε σχέση με τη Ευρωμασιογειακή Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ για τις αεροπορικές μεταφορές. Αυτή η ε, συμφωνία θα υποβληθεί σε ψηφοφορία στην πρώτη σημερινή σύνοδο. Όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός πλαισίου που ευνοεί τις βιώσιμες επενδύσεις και το άλλο για τις κοινοτικές στατιστικές σε θέματα μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας, σας ενημερώνω πως δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση ε, που να στοχεύει στην απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου και δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες με βάση το άρθρο 67 και 68 του κανονισμού. Οι πράξεις λοιπόν που προτείνονται θα θεωρηθεί πως εγκρίνονται. Έπειτα, μετά από τις ε, διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες, θέλω να υποβάλω στη Σύνοδο την εξής πρόταση τροποποίησης του οριστικού σχεδίου μερίσης διάταξης Όσον αφορά την Τετάρτη, οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την προετοιμασία της ε, ε, Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 Ιουνίου και τις δηλώσεις της ε, κυρία Σπύρη και του κυρίου Χάνσεν για τις διαπραγματεύσεις για τη νέα εταιρική σχέση με το Ενωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία θα εξεταστούν σε μια συζήτηση κοινή που θα γίνει ως δεύτερο σημείο απόψε μετά από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά το θάνατο του George Φλόιντ. Όσον αφορά την πέμπτη, τρεις δηλώσεις ε, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής είπα του εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλεια για τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στην εξωτερική πολιτική. Δεύτερη, για το νόμο τη Λαϊκή Δημοκρατία τη Κίνα για την εθνική ασφάλεια για το Χονγκ Κόνγκ και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπιστεί τον υψηλό βαθμό αυτονομία του Χονγκ Κόνγκ. Τρίτο σημείο αφορά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενδεχόμενη στην ε, προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας στο Ισραήλ. Θα γίνει συζήτηση ε, ως πρώτο σημείο αύριο. Στη συνέχεια θα γίνουν δύο σύντομε παρουσιάσει. Πρώτον, έκθεση του κυρίου Αστρεβίσιου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι συστάσει του για την Ανατολική Εταιρική Σχέση εν ώψη τη διάσκεψη κορυφή του Ιουνίου 2020 και έκθεση Πίκουλα για τι συστάσει του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια μετά από τη διάσκεψη του 2020, κορυφής του 2020. Θα εξεταστούν λοιπόν με μια δήλωση, μάλλον συγγνώμη, διορθώνει ο Πρόεδρος σε μια σκηνή συζήτηση ω τρίτο σημείο αύριο το πρωί μετά από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την αγώνα κατά των εξατιών παραπληροφόρηση στη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και ε, σε σχέση με την ελευθερία έκφρασης. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ε, τροπολογιών που υποβλήθηκαν και των ε, χωριστών και κατά τμήματα ψηφοφοριών θα γίνουν διάφορες σύνοδοι ψηφοφοριών και θα ψηφίσουμε για τα έγγραφα προτεραιότητες πρώτα. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Οπότε εγκρίνονται οι τροποποίησεις αυτές. Τώρα, Όσον αφορά το διαδικαστικό για ενημέρωση της ψηφοφορίας για την έκθεση τέλη που έχει να κάνει με την σύναψη Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 196 του κανονισμού εκτός από το συντάκτη του ψηφίσματος θα μπορέσουν να παρέμβουν μόνο ένας ομιλητής κατά και ο πρόεδρος και η της αρμόδιας επιτροπής επί της Θέλει κανείς το λόγο εδώ. Το λόγο έχει η κυρία Κλέρ που θα υποβάλει το σχέδιο ψηφίσματος. Κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα να συμφωνήσω με το αίτημα να αναβληθεί η ψηφοφορία σχετικά με την υποκήρυξη της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας με το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει άμεσες πρακτικές συνέπειες η συμφωνία αυτή, διότι εφαρμόζεται προσωρινά από το 2013 και μετά. Το να υιοθετηθεί τώρα όμως ε, στο πλαίσιο της ανακοίνωση ε, της νέας Ισραηλινής κυβέρνησης ε, σχετικά με του στόχους της να προσαρτήσει το 1 τρίτο τη, δυτική όχθη παραβιάζοντα παραβιάζοντας το εθνικό δίκαιο, το, το διεθνές δίκαιο, θα ήταν ένα μήνυμα ασυνεπές από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θεωρείται ότι ενισχύει τις διμερείς συμφωνίες με το Ισραήλ ε, και θα αποτελούσε και ε, αλλαγή της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά το Ισραήλ και την επίλυση των διαφορών. Κάτι τέτοιο θα επιταχύνει τις συγκρούσεις με τον Παλαιστινιακό λαό. Δεν θα πρέπει να ομαλοποιούμε τις παραβιάσεις του διεθνούς και από πλευρά του Ισραήλ και παρακαλώ του συναδέλφου ε, να υποστηρίξουν την αναβολή αυτή τη απόφαση. Σα ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιο ομιλητή ε, που να είναι κατά. Όχι, ο εισηγητή. Πρόεδρε, ε, ως εισηγητής πρέπει να πω ότι η συμφωνία αυτή περιμένει ήδη υπερβολικά πολύ καιρό για την επικύρωσή της και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση στον τομέα αερομεταφορών. Τέτοιες συμφωνίες επιφέρουν νομική ε, βεβαιότητα, ασφάλεια δικαίου και για τους εργαζόμενους και προστατεύουν και τους ε, επιβάτες, τους οποίους επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ήδη επικυρώσει τη συμφωνία αυτή. Δεν μπορώ λοιπόν να δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο από το ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει τη συμφωνία. Αυτό λοιπόν είναι απλά το τελευταίο στάδιο και πρέπει να πω ότι δεν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει εμπόδιο. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης, όχι μέρος του ε, προβλήματος. Σας παρακαλώ λοιπόν να διατηρήσουμε στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή. Υπάρχει κάποιος ε, ε, κατά όχι. Προχωράμε με βάση τα τρία αιτήματα που θα ζητήθηκε να εξεταστούν ως κατεπήγοντα και θα ψηφιστούν στην πρώτη σύνοδο ψηφοφοριών. Μπορούμε να ακούσουμε μόνο του συντάκτες των αιτημάτων ε, και έναν ομιλητή κατά, καθώς και τους προέδρους ε, των αρμοδίων τη ουσία επιτροπών. Υπάρχει κάποιος που θέλει να παρέμβει για το αίτημα τη Επιτροπής ΕΚΟΝ. Κύριε Πρόεδρε, ζητήθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής ΙΚΟΝ ε, να διαβάσω το εξή κείμενο σχετικά με την επίγουσα διαδικασία. Στις 8 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε πρόταση που τροποποιεί την οδηγία διοικητικής συνεργασίας ε, τροποποιώντας ε, τις προθεσμίες για τους σωματοπιστωτικούς οργανισμούς ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας. 1η Ιουλίου προβλέπεται η υιοθέτηση αυτή τη οδηγία και ακολουθείται η διαδικασία διαβούλευση. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να υιοθετήσει ομόφωνα την θέση του αν δεν έχει λάβει πρώτα την θέση του Κοινοβουλίου. Ε, το Συμβούλιο προχώρησε πολύ γρήγορα με γενική προσέγγιση που συμφωνήθηκε στην Κορεπέρα αρχέ ε, Ιουνίου. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ε, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλεί το Κοινοβούλιο να υποβάλει τη γνωμοδότησή του μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι συντονιστές της ΕΚΟΝ λοιπόν αποφάσισαν να ακολουθήσουν την επίγουσα διαδικασία σύμφωνα με τον, το άρθρο 163 του κανονισμού. Ευχαριστώ κυρία Πίνγκ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μανών Ομπρί για παρέμβαση ε, κατά του αιτήματο τη Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπό την πίεση του λόμπι των τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζητάει να ψηφίσουμε κατεπηγόντως τα μέτρα φορολογικής διαφάνειας ε, τα οποία χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή. Ε, Μα ζητάτε λοιπόν να αποφασίσουμε κατεπηγόντω για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Περιφρονείται δηλαδή το Κοινοβούλιο. Είναι απαράδεκτο. Η ομάδα μα θα ψηφίσει κατά αυτή τη έκτακτη διαδικασία, τη επίγουσα διαδικασία και απευθυνόμαστε σε όλε τι πολιτικέ ομάδε. Αυτή η μέθοδο, αυτή η διαδικασία είναι ενδεικτική τη σημασία τελικά που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην, στη φοροδιαφυγή. Ε, για άλλη μια φορά καθυστερούμε την θέσπιση εργαλείων που θα μα επέτρεπαν να προχωρήσουμε. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, πρέπει να συμπεράνουμε ότι επίγει να περιμένουμε. Επήγει να περιμένουμε και να μην κάνουμε τίποτα για τη φοροδιαφυγή. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη πρέπει να δαπανίσουν τώρα άμεσα δισεκατομμύρια ευρώ για να σώσουν τι οικονομίε του, να σώσουν θέσει απασχόληση, να σώσουν επιχειρήσει. Και είναι η στιγμή τώρα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή, να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα δισεκατομμύρια χρήματα που έχουν χα, χαθεί από τη φοροδιαφυγή. Πάντα θα υπάρχουν λόγοι έτσι ώστε οποιαδήποτε ρύθμιση να παραπέμπεται στον αιώνα του άπαντα. Εμεί δεν θέλουμε να διευκολύνουμε όμω τα τραπεζικά λόμπι. Εμεί νομοθετούμε, όχι τα λόμπι. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να αρχίσουμε να αντιστεκόμαστε στα λόμπι και να δρούμε προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να παρέμβει για το αίτημα της Επιτροπής Άγκρη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπάιτς για να παρέμβει κατά του αιτήματο Επιτροπής Άγκρη. Παρακαλώ. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν ε, υπάρχει αντίρρηση ότι ε, είναι ώρα να υποστηρίξουμε τους αγρότες της Ευρώπης ε, στην κρίση αυτή που περνάμε. Ωστόσο, στην κοινή γεωργική πολιτική μας υπάρχουν αποθέματα για κρίσεις. Ε, και το Συμβούλιο και η χώρα μου, η Αυστρία, ε, έλαβαν απόφαση κατά της ε, καταβολής επιδοτήσεων από το απόθεμα για τις κρίσεις. Μπορώ μόνο να μαντέψω ποιοι είναι οι λόγοι για αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του δεύτερου πυλώνα για την προστασία του κλίματος ε, για την ε, βελτίωση του περιβάλλοντος και γι' αυτό εμείς ε, οι πράσινοι θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά. Ως ευρωβουλευτές εδώ στο Κοινοβούλιο υποβάλλουμε τροπολογίες και θέλουμε να αν ανακληθεί αυτή η πρόταση, οι γεωργοί μας δεν θα λάβουν καμία βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την ε, ομάδα μου να μην καταψηφίσει την πρόταση. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιο να παρέμβει για το αίτημα της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Ο κύριος Βίντσι, παρακαλώ. Υπέρ ή κατά είστε. Υπέρ. Είμαι εισηγητής. Κύριε Πρόεδρε, η πανδημία είχε η σημαντικό αντίκτυπο στις πρωτοβουλίες πολιτών που δεν πόρεσαν να, να οργανώσουν καμπάνιες συλλογής υπογραφών. Πρέπει να τους υποστηρίξουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι η συμμετοχική δημοκρατία που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να λειτουργήσει. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό για την Ένωσή μας. Θέλω να ζητήσω λοιπόν να δεχτείτε να αποδεχθούμε τον κανόνα 163 για κατεπίγουσα διαδικασία για να αντιμετωπίσουμε την πρόταση της Κομισιόν για ένα κανονισμό σχετικά με τα προσωρινά μέτρα, σχετικά με τα χρονικά όρια για τη συλλογή επαλήθευση ε, που προβλέπεται στο, στο κανονισμό 877 του 2019 για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στα πλαίσια του COVID-19 όλα αυτά ε, όπως άλλωστε αποφασίστηκε με ευρία πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που θέλει να παρέμβει κατά? Όχι. Ε, Οπότε έτσι ορίζεται πλέον η ημερησία διάταξη. Και τώρα περνάμε στις συζητήσεις. Η πρώτη αφορά τις αντιρατζιστικές διαμαρτυρίες μετά από το θάνατο του George Floyd. Θυμίζω ότι δεν προβλέπεται η διαδικασία Catch the Eye. Ε, ούτε θα γίνουν ερωτήσει με γαλάζια κάρτα. Παρακαλώ, Υπουργό Μπρινιάτ. Εξ ονόματο του Συμβουλίου. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστούμε που καλέσατε την Προεδρία να ε, μοιραστεί μαζί σας ε, τις θέσει τη πάνω ε, στο πολύ επίκαιρο καυτό θέμα του ρατσισμού. Ήταν συγκλονιστικό ο θάνατο του George Floyd και οδήγησε σε διαμαρτυρίες όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, εκφράζοντας ε, στο όνομα της Κροατικής Προεδρίας ε, και του Συμβουλίου να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους, στην οικογένεια του George Floyd. Ε, αλλά ε, πρέπει ε, να επιδείξουμε αλληλεγγύη για όλα τα θύματα ρατσισμού σε όλο τον κόσμο. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός δεν έχουν θέσεις στις κοινωνίες μας. Οι διαμαρτυρίες θίγουν το θέμα της συμπεριφοράς της αστυνομίας απέναντι στους Αφροαμερικανούς και την θέση τους στην κοινωνία. Και λόγω της ε, ιστορία ε, της κάθε χώρας ε, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί ένα προς ένα στην Ευρώπη. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η απαγόρευση διακρίσεων είναι οι ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας ε, για να καταπολεμήσουμε τον ε, ρατσισμό. Το βασικό είναι ο Ευρωπαϊκός ε, Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση λόγω χρώματος φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας. Η ίση μεταχείριση σημαίνει ότι παρέχεται νομική προστασία και αυτό είναι το βασικό εργαλείο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όχι μόνο επέκτηνε την προστασία, αλλά άλλαξε και την υποδομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι έπρεπε ε, τα κράτη-μέλη να ορίσουν ε, εθνικούς φορείς ε, για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης. Η Προεδρία είναι προσιλωμένη στο στόχο της καταπολέμησης του ρατσισμού και γι' αυτό θα ήθελα να σας ανακοινώσω τον εορτασμό της 20ης επαιτίου αυτού του σημαντικού εργαλείου που έχει οργανωθεί από την Κροατική Προεδρία, ε, τους Εθνικούς Φορείς Ισότητας ε, και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα έχει θεσπίσει ένα στιβαρό νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της μυσαλλοδοξίας και του μίσους, όπως είναι η απόφαση πλαίσιο του 2008 για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Τον Ιούνιο του 2016 το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την σωστή εφαρμογή αυτής της απόφασης πλαίσιο καθώς και άλλων σχετικών ε, νόμων σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον ζητείται από όλα τα κράτη-μέλη να ε, αναπτύξουν μεθόδους για την σωστή καταγραφή ε, των εγκληματών μίσους. Τον Οκτώβριο του 2017 το Συμβούλιο επίσης χαιρέτησε τα μέτρα τη επιτροπή Υψηλού Επιπέδου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση τη ξενοφοβία του ρασισμού και άλλων μορφών μυσαλλοδοξίας. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να συνοδεύονται από αντιρατσιστική εκπαίδευση, ε, δουλειά με τους νέους και πιο συγκεκριμένα την ε, ανάγκη ανάπτυξης δημοκρατικής ανθεκτικότητας ε, στην εκπαίδευση. Συνοψίζοντας, ε, έχουμε εργαλεία, έχουμε νομοθεσία, γνώσεις, εκπαίδευση, έχουμε ε, σωστά αφηγήματα, ε, αλλά και ποινές για τα απαγόρευση των διακρίσεων του, της δωρικής μίσους κλπ. Πρέπει όμως να επαγρυπνούμε όταν βλέπουμε τέτοια δείγματα ρητορικής μίσους ε, εις βάρος μειονοτήτων. Ε, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, τον Νοέμβριο του 2018 σε έκθεση αποκάλυψε τις απίστευτες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι, οι μαύροι στις κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν διακρίσεις ε, κατά την αναζήτηση εργασίας, ε, στην εκπαίδευση, ε, στις δουλειές που έχουν και στην εξέβριση στέγασης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα θέματα αυτά. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στην καταπολέμηση του ρατσισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιλωμένη στην καταπολέμηση κάθε μορφής ε, Διάκριση ε, και εντός των συνόρων της ε, και σε όλο τον κόσμο. Τον Μάρτιο του 2019 το Συμβούλιο υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για τις μη διακρίσεις στις εξωτερικές δράσεις. Ε, παρέχεται έτσι προσανατολισμός ε, για να ε, βελτιωθεί η εφαρμογή της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αυξήσει την ορατότητα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση του ρατσισμού στις εξωτερικές της δράσεις. Η κατάχρηση εξουσίας θα πρέπει να καταδικάζεται παντού. Οι κοινωνίες που περηφανεύονται ότι αντιπροσωπεύουν το κράτος δικαίου, τι θεμελιώδει ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να θέτουν το καλό παράδειγμα. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε κατά της ε, υπερβολικής ε, χρήσης ε, εξουσίας και θα πρέπει να φροντίσουμε περιστατικά όπως ήταν η δολοφονία του George Floyd να αντιμετωπίζονται άμεσα και να εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, πιστεύουμε ότι ο Αμερικανικός λαός ε, θα μπορέσει να συσπηρωθεί ε, ως έθνος και να αντιμετωπίσει αυτά τα σημαντικά προβλήματα. Ο ρατσισμός όμως δεν είναι πρόβλημα μόνο, στην μόνο στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπως έχουμε δει. Η ευθύνη για την καταπολέμηση του ρατσισμού ανήκει σε όλους μας. Πολιτικούς, δασκάλους, σπουδαστές, πολίτες. Όλων μα είναι αυτή η ευθύνη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Και τώρα το λόγο έχει η Πρόεδρος Φοντερ Λάγιαν. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Mr. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, δεν ξέρω τι σημαίνει να είναι κανείς μαύρος. Δεν ξέρω τι σημαίνει να είναι κανείς ε, μαύρος ή μέλος κάποιας μειονότητας ε, εθνοτικής, ε, σεξουαλικής, θρησκευτικής, εκεί που έχω ζήσει. Δεν είχα ποτέ την εμπειρία του να μου φερθούν διαφορετικά μόνο και μόνο λόγω της εμφάνισής μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει να με κοιτάζουν καχύποπτα, να μου συμπεριφέρονται καχύποπτα καθημερινά στον δρόμο, όταν κάνω τα ψώνια μου, όταν ψάχνω ένα σπίτι για να στεγαστώ, όταν ψάχνω μια θέση εργασίας. Μετά από αυτήν την απίστευτη ιστορία που διηγήθηκε η συνάδελφός. Οι περισσότεροι από εμάς δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ξέρουμε όμως κάτι. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν ζήσει αυτά και μας το λένε ότι ανεχόμαστε το ρατσισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτό πρέπει να λάβει τέλος κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτοί που διαδηλώνουν στους δρόμους μας, στις χώρες μας και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, τον κόσμο ολόκληρο, υψώνουν τις φωνές τους και θέλουν οι φωνές τους να ακουστούν. Ήρθε η στιγμή όμως να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να ακούσουμε, κάτι περισσότερο από το να καταδικάσουμε. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για το ρατσισμό. Ανοιχτά και ειλικρινά. Γι' αυτό λοιπόν Θέλω να σας ευχαριστήσω που συμπεριλάβατε το θέμα αυτό στην τη διάταξη της Ολομέλειας και που το βάλατε ως πρώτο θέμα στην σύνοδο αυτή. Αξιότιμα μέλη. Ως κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Εμείς αδιάκοπα θα πρέπει να καταπολεμούμε το ρατσισμό και τις διακρίσεις. Τις ορατές διακρίσεις αλλά και τις πιο υποχθόνιες διότι υπάρχουν και προκαταλήψεις ασυνείδητες και στον τομέα της δικαιοσύνης, στον τομέα της επιβολής του νόμου, στον τομέα της στέγασης, στον τομέα της αγοράς εργασίας, στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της υγείας, στον τομέα της πολιτικής, στον τομέα της μετανάστευσης. Πρέπει λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, δημόσιο, ιδιωτικό, σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Ο κάθε ένας από εμά ατομικά, ο κάθε πολίτης, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη πιο ίση, πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη και θέλω να είμαι σαφής, στην, ένωση, στην ένωσή μας δεν υπάρχει θέση για τον ρατσισμό ή για καμία, κανένας είδους διάκριση και αυτό είναι βέβαιο. Αξιότιμα μέλη, θα πρέπει από κοινού να απαντήσουμε σε δύσκολα ερωτήματα. Γιατί ο ρατσισμός και οι διακρίσεις επιβιώνουν, αντέχουν στις κοινωνίες μας. Γιατί υπάρχουν πολιτικά κόμματα που υποστηρίζουν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και που κερδίζουν εκλογές. Γιατί οι μέλη εθνικών μειονοτήτων, προσθετικών μειονοτήτων υποεκπροσωπούνται σε πολιτικό, κοινωνικό, ακαδημαϊκό επίπεδο και υπερακροσπροσωπούνται σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τι ασθένειε, τη φτώχεια, την επιβολή του νόμου. Τι μπορούμε να κάνουμε στην τομέα τη εκπαίδευση, τη απασχόληση, τη στέγαση, τη υγεία, να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη, πιο ανοιχτή κοινωνία, πιο ενσυνείδητη, έτσι ώστε και στους θεσμού μας να, εκπροσωπούν είτε πιο ορθά, πιο πιστά η ποικιλομορφία της κοινωνίας μας. Αυτό δεν είναι θέμα μίας μόνο πολιτικής ή ενός ανθρώπου ή ενός επιτρόπου. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ σήμερα ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω πραγματικά αυτό το, αυτά τα θέματα να τα δούμε σε βάθος. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει μια δομημένη συζήτηση για τον ρατσισμό στο Κολέγιο των Επιτρόπων και θα πρέπει και εδώ, σε αυτό το ημικύκλιο, να δούμε εκπροσωπείται η ποικιλομορφία της κοινωνίας μας. Όχι. Και δεν είναι βεβαίως καλύτερα τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τον ρατσισμό και θα πρέπει και να δράσουμε. Πάντα μπορούμε να αλλάξουμε κατεύθυνση εφόσον υπάρχει βούληση για κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να πάρω ένα μικρό παράδειγμα, να σας αναφερθώ σε ένα μικρό παράδειγμα το οποίο έζησα όταν ήμουν υπουργό Άμυνα στη χώρα μου. Τότε είχαμε ένα σύστημα στρατολόγησης της ενόπλης δυνάμεις που πάντα ήταν υπέρ των ίδιων. Είχαμε εξαιρετικού υποψηφίους που είχαν πολλά να προσφέρουν στις ενόπλες δυνάμεις μας. Ορισμένοι μιλούσαν αραβικά, φαρσί, πολύ σημαντικά πνευματικές δεξιότητες, αλλά αυτά δεν τα αξιολογούσαμε. Καθόλου. Ενώ τέτοιες δεξιότητες σε μια αποστολή μπορεί να σώσουν ζωές. Και τότε μας έλεγαν το σύστημα δεν μας το επιτρέπει. Αυτό δεν το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Όμως τότε, μετά από ανάλυση, μετά από σκέψη, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις άλλαξαν το σύστημα στρατολόγησής τους και αυτό ήταν καλό για τις ίδιε ενόπλε δυνάμεις και για την ίδια την κοινωνία. Έχουμε τώρα ένα πιο δίκαιο σύστημα για αυτού τους στρατιώτες. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, υπάρχει τρόπος. Αξιότιμα μέλη θα πρέπει να μιλήσουμε για τον ρατσισμό με ανοιχτό πνεύμα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν ξεκινάμε βεβαίω από το μηδέν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι διακρίσεις απαγορεύονται στο υψηλότερο νομικό επίπεδο. Αναφέρομαι στη συνθήκη μας, στην Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων. Υπάρχουν και ευρωπαϊκοί νόμοι κατά του ρατσισμού, κατά των εθνικών διακρίσεων, του λόγου μίσους, της ισότητας. Υπάρχουν νομοθεσίες για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, Έχουμε εργαλεία με ομάδε ψηλού επίπεδου, με εμπειρογνώμονε από όλα τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση τη ξενοφοβία, άλλε μορφέ ε, μη ανεκτικότητα. Και βεβαίω ε, υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για αυτά. Όμω θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Χαίρομαι που ζω σε μια κοινωνία που καταδικάζει το ρατσισμό. Δεν φτάνει όμως αυτό. Όταν διαπιστώνουμε τέτοια φαινόμενα πρέπει να κρούμε τον κόδωνα το, το του κινδύνου και να αντιδρούμε άμεσα. Διότι ξεκινάει σε πολύ μικρή κλίμακα αυτή η ευαισθητοποίηση στο επίπεδο του καθενό από εμά. Η ευαισθητοποίηση έχει να κάνει και με το να εξετάσουμε τον ίδιο μα τον εαυτό. Να αντιδρούμε και να παρεμβαίνουμε όταν βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα διακρίσει. Να αμφισβητούμε προνόμια τα οποία θεωρούνται δεδομένα. αξιότιμα μέλη. Λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε ενωμένοι στη διαφορετικότητά μας. Αυτό όμως θα πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Θα πρέπει να πάρουμε σάρκα και ωστά αυτές οι λέξεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη Ευρώπη ενωμένη, ενωμένη στη διαφορετικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie. Grazie Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για την παρουσία σας και για τα λόγια σας. Και τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες εξ του ε, Λαϊκού Κόμματος, κυρία Λίμα. Παρακαλώ, Ιζαμπέλα. η επανάσταση, η άρνηση με όλες τις δυνάμεις μας, με το πνεύμα μας αλλά και με τα σωθικά μας κάθε μορφή ρατσισμού. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό είναι το καθήκον μας εδώ των βουλευτών στο πλαίσιο, μέσα σε αυτή την αίθουσα. Γι' αυτό ήταν σημαντικό να έχουμε ένα κείμενο κοινό για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ε, δυνατή φωνή ε, για την άρνησή μας και την απόλυτη καταδίκη του ρατσισμού. Την αλληλεγγύη μας να εκφράσουμε με όλους όσους ε, υποφέρουν από τις διακρίσεις. Ένα ισχυρό μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου. Ο βίος θάνατος του George Floyd ε, ε, αναζωγόνησε την ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο να εκφραστεί η άρνηση του ρατσισμού και της αστυνομική βίας. Αυτό το κίνημα που συγκέντρωσε τόσους πολλούς νέους δίνει ελπίδα για το μέλλον. Θέλω όμως να εκφράσω και την θαυμασμό μου για τους υπόλοιπους αστυνομικούς που κάνουν τη δουλειά τους με υποδειγματικό τρόπο και για τους οποίους το να είναι αστυνομικοί δεν είναι απλά ένα επάγγελμα, αλλά είναι πραγματικά ε, ε, μια ε, ένα καθήκον και ένα λειτουργήμα. Να μπορέσουμε λοιπόν να πούμε πως όχι δεν μπορούμε να, να μην ντρεπόμαστε για τα όσα συμβαίνουν. Είναι προφανές όταν σκεφτεί κανείς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Πρέπει να είναι προφανή όταν μιλάμε, για, όταν βλέπουμε ε, βάρκες γεμάτες με σκλάβους. Οι κανόνες που εμείς φτιάχνουμε σήμερα και αύριο για ένα καλύτερο μέλλον θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την καθημερινότητα, να μπορέσουμε να στήσουμε μια πολιτική που θα μπορέσει να δώσει σε όλους άνευ διακρίσεων τις ίδιες ευκαιρίες και θα μπορέσει να εκριζώσει το ρατσισμό. Σας ευχαριστώ. Γκαρσία Πέρες, εξ των Δημοκρατών και Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τα λόγια του George Floyd μετά από μια αγωνία 8 λεπτών και 45 δευτερολέπτων δεν είναι μόνο η κραυγή μια στιγμής. Είναι η αδικία και η πραγματικότητα μια εποχή ολόκληρη. Γιατί λοιπόν αυτή η πραγματικότητα οδηγεί σε ασφυξία του μαύρους και του λευκού, λευκούς. Γιατί και η κρίση του COVID πνίγει περισσότερο τους μαύρους από ό,τι τους λευκούς. Η Ρόζα Πάρξ βρέθηκε στη φυλακή διότι δεν θέλησε να σηκωθεί από τη θέση της για ένα λευκό και να πάει να κάτσει πίσω στο λεωφορείο. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ πλήρωσε με τη ζωή του μετά από μια προσπάθεια για να βάλει τέλος στις διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, παρόλα αυτά, δεκαετίες μετά, τα όνειρά του παραμένουν ζωντανά. Αυτή η κραυγή για τη δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα που ακούγεται σε όλους τους δρόμους του κόσμου μας έχουν επιστρέψει την ελπίδα και η ελπίδα βεβαίως σημαίνει δέσμευση και εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρω... των... της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας πρέπει να εκριζώσουμε τον θεσμικό ρατσισμό που υπάρχει στις χώρες μας. Είναι απαράδεκτο από το 2008 να έχουν μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο η οδηγία κατά των διακρίσεων. Και βλέπω εδώ την Επίτροπο, την κυρία Ντάλη. Ελπίζω πραγματικά να έχουμε εδώ μία σύμμαχο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απεμπλέξουμε αυτό το φάκελο. Χρειαζόμαστε και νομοθετικά εργαλεία για να μπορέσουμε να βάλουμε τέλο στο ρατσισμό στην Ευρώπη. Τη στιγμή που αναγεννώνται εδώ πολιτικές δυνάμεις που ανοιχτά μας λένε ότι είναι ρατσιστές. Οι λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους, αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όταν κάποιος υπόκειται ε, σε διακρίσεις ε, λόγω της φίλου του, λόγω του χρώματός του, ε, τότε αυτό το ξαναβρούμε μπροστά μας. Πρέπει να εγγυηθούμε ότι όλα τα ανθρώπινα όντα θα είναι ελεύθερα και ίσα. Χάρη στις φωνές των εκατομμυρίων συμπολιτών μας, θυμηθήκαμε ότι οι μαύρες ζωές μετράνε. Πρέπει να το πούμε λοιπόν σοβαρά. Πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε άσπρα γόνατα πάνω σε μαύρους λαιμούς. Ε, Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Τσόλος, εξ ονόματο του Ρινιού. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ζωές των ε, μαύρων έχουν σημασία. Όλες οι ζωές έχουν σημασία. Όμως ε, βλέπουμε πως στην κοινωνία μας ακόμα δεν υπάρχει σεβασμός ε, για την ανθρώπινη ζωή. Όμως ε, ο ρατσισμός δεν είναι αποκλειστικά αμερικάνικο πρόβλημα, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτό που συμβαίνει στη ΣΥΠΑ με τον Τζόρτζ Φλόιντ, η επιθετικότητα που φάνηκε στην θάνατό του και η έλλειψη σεβασμού για την ανθρώπινη ζωή και όλα όσα αυτό σημαίνει θα πρέπει να μας επιτρέψουν να δούμε τι συμβαίνει εδώ στο δικό μας χωριό, το ευρωπαϊκό. Να να δούμε ότι ο ρατσισμός και οι διακρίσεις υπάρχουν δεξιά, μάλλον δυτικά και ανατολικά. Πολύ συχνά ο φόβος του άλλου συνοδεύεται από βαθιές διακρίσεις που είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, θεσμικού, κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες που τελικά βλάπτουν το σύνολο της ε, κοινωνίας μας και δυστυχώς συμπεριλαμβανομένων κάποιοι πολιτικοί ε, παίζουν με αυτό το αίσθημα φόβου για να το χειραγωγήσουν υπέρ του σε εκλογικέ αναμετρήσεις. Είναι διαφορετικό το να έχουμε μια κοινωνία που επιτρέπει να, έχει, να φοβάται κάποιο επειδή είναι διαφορετικό από του υπόλοιπου δεν είναι κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει την πολυμορφία ατού τη και δεν αρκεί να νομοθετούμε υπέρ της ποικιλομορφίας και της ε, κατάρρησης των διακρίσεων. Πρέπει να το καλλιεργούμε, όχι να το επιβάλλουμε με τη βία, αλλά να το καλλιεργούμε με τη καλή θέληση. Πρέπει να αρχίσουμε ο καθένα από τον εαυτό του. Και θέλω εξ ονόματο τη πολιτική μου ομάδα να προτείνω να συνεργαστούμε οι τρει θεσμοί. Το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, το Συμβούλιο, να κάτσουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι και να διερωτηθούμε αν οι θεσμοί μας στο εσωτερικό τους αντικατοπτρίζουν πραγματικά την πολυμορφία της Ένωσης. Ζητώ συμβουλή και από εσά Συμβητώ από το Συμβούλιο να στηρίξει τη δημιουργία μια task force σε αυτό το θέμα και από εσά το ζητώ, κυρία Πρόεδρο, για να ξεκινήσουμε από εμά του ίδιου, εμεί οι ίδιοι να είμαστε πιο ανοιχτοί. Και όταν θα δώσουμε εμεί το καλό παράδειγμα, θα ζητήσουμε και από του υπόλοιπου να σεβαστούν αυτό το παράδειγμα. Οι και οι διακρίσει, ο ρατσισμό και οι διακρίσει είναι μια ντροπιαστική πτυχή του παρελθόντος μας αλλά και δυστυχώς του παρόντος μας. Γι' αυτό θα ήθελα να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν θα αποτελέσουν και τμήμα του μέλλοντός μας. Ευχαριστώ. Τσεκάρτη, ID. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο θάνατος ενός ανθρώπου ε, μετά από την άσκηση της βίας πρέπει να δικαιωθεί και έτσι και δίκαια ολόκληρος ο κόσμος έχει εκφράσει την οργή του ε, μετά από το θάνατο του George Φλόιντ. Αλλά για το διεθνή τύπο ε, του σειρμού ορισμένες ζωές έχουν περισσότερη αξία από άλλες και αυτό ισχύει για τον David Dorn που θέλω να θυμίσω ένας νεαρός Αμερικανός μαύρος που που πέθανε τον Ιούνιο το, απευθείας στο facebook ενώ προσπαθούσε να υπερασπιστεί στο Σεν Λουί έναν φίλο του που δέχτηκε επιθέσεις και εκείνος ήταν μαύρος και αθώος 25 μόλις ετών όμως για εκείνον καμία απορία δεν έγινε καμία διαμαρτυρία οι διαμαρτυρίες στην Αμερική γίνονται όλο και πιο βίες και έχουν ξεχυθεί και στην Ευρώπη. Στην οργή κατά των αστυνομικών ε, ε, υπάρχει και η οργή των ε, οικονομάχων κατά των ε, αγαλμάτων διαφόρων ε, ανθρώπων του παρελθόντος, όπως του Χριστόφορου Κολόμβου και τα Αυτό όμως δεν θα λύσει τα προβλήματα του ρατσισμού. Πέρα από το ρατσισμό υπάρχει μια ανοιχτή πληγή που επίσης υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Είναι η άγνοια και η, και η βλακεία των όσων θέλουν να κυρώσουν την ιστορία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκούνκερ από τους Πρασίνους. Η κυρία Κούνκερ, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, κύρια Πρόεδρε Φόντερ Λάιεν, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, λίγες μέρες ε, μετά ε, την δολοφονία του George Floyd, ε, έβαζα για ύπνο την μικρότερη μου κόρη. κάποια στιγμή σώπασε και με ρώτησε, θα σκοτώσουν και μένα. Η απεικιοκρατία έχει καθορίσει τις ε, κοινωνίες της Αμερικής ε, και της Ευρώπης εδώ και ε, αιώνες έχει δημιουργήσει ε, βαθιές ε, προκαταλήψεις ε, που ακόμη επηρεάζουν και όπως βλέπουμε σκοτώνουν ανθρώπους. Φυσικά η δομή του ρατσισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετική από ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν έχουμε την ίδια ιστορία σκλαβιάς και λιντσαρισμάτων. Έχουμε όμως καταγεγραμμένες θηριωδίες στη δική μας απεικιοκρατική ιστορία που ε, ακόμη φαίνεται σήμερα στις διακρίσεις ε, και τη βία συμπεριφορά της αστυνομίας. Επίσης έχουμε πρόσφατη ιστορία συστηματικής δίωξης μειονοτήτων ε, τον ΛΟΑΤΚΙ, τον Ρώμα. Κανείς δεν είναι ελεύθερος εάν δεν είναι όλοι ελεύθεροι. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στο δικό μας σπίτι. Ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσουν ε, το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καταφέρει να δημιουργήσει μια δίκαιη κοινωνία που να μην αφήνει κανέναν πίσω. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν να ξεμπλοκάρει η οδηγία κατά των διακρίσεων που έχει κολλήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το 2008. Κυρία Πρόεδρε, καλώ εσά και την επικείμενη Γερμανική Προεδρία να αδράξουν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να αναλάβουν δράση. Απόψε, θέλω ε, όταν θα βάζω για ύπνο την κόρη μου να την ε, διασφαλίσω ότι θα είναι καλά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρνούμαστε να ε, σοπάσουμε λόγω του μίσους και της άγνοιας. Και ρωτώ στο όνομα της κόρης μου, αν όχι τώρα, τότε πότε. παρακαλώ, Χέρμαν από το e Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά εδώ η Ευρώπη ε, δείχνει αυτή την υπεροψία, τη γνωστή πόσο καλοί είμαστε εμείς Ευρωπαίοι και, και πώς μας αρέσει να μιλάμε άσχημα με τους Αμερικανούς. Θα διαβάσω κάτι που το έχει γράψει και το έχει πει ένας Ευρωπαίος τώρα που έχει σύμμαχους εδώ στην Ευρωκοινοβούλιο και που ένα μέλος του κόμματός του βρίσκεται εδώ τα ζώα αυτά, οι ίενες, τα σαρκοβόρα αυτά ζώα είναι αυτά που μοιράζουν, σπέρνουν το μίσος απέναντι στην Καταλωνία και στην καταλανική γλώσσα. Ο Τωρά το είπε αυτό, που είναι επικεφαλής Τη αυτόνομη περιφέρεια τη Καταλωνία και είναι το κόμμα του εδώ, ο κ. Πουτζεμόν είναι εδώ, ο κ. Τώρα είναι σύμμαχος του Πρωθυπουργού του κ. Σάντσεθ αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Είναι σύμμαχος με του κομμουνιστές, με τους σοσιαλιστές, ένας ρατσιστής λοιπόν, ο οποίο κυβερνάει μέρο τη Ισπανία, κατά των Ισπανών. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται κανεί λοιπόν να πάει στην Αμερική. Στην Αμερική είχαμε ένα τραγικό κεφάλαιο με ένα τραγικό περιστατικό από ένα έγκλημα ενός αστυνομικού σκοτώθηκε ένας μαύρος ο οποίος ήταν, είχε παρελθόν στη φυλακή, ο άνθρωπος αυτός σκοτώθηκε και αυτό οδήγησε σε ένα κύμα ρατσισμού κατά του Αμερικανικού συστήματος. Ένα κύμα μίσους κατά του Αμερικανικού έθνους που χρησιμοποιείται, χειραγωγείται πολιτικά κατά των Αμερικανών και κατά του Προέδρου της. Και τώρα έχουμε άλλη μια χειραγώγηση λοιπόν. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Ομαρζέ από την ε, Γκούε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά τιμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινάει αυτή η ολομέλεια με αυτή τη συζήτηση και στο όνομα όλη τη ομάδας μας θέλω να σα ευχαριστήσω γι' αυτό. Συνέβη λοιπόν αυτό το περιστατικό, το τραγικό, το οποίο έγινε μια σημαντική πολιτική στιγμή. Αυτές οι οκτώ, τα αυτά τα οκτώ λεπτά στα οποία πάγωσε η ζωή του, του, του George Floyd ε, έβαλαν μπροστά ένα ολόκληρο κίνημα. Και η αγανάκτησή μας σήμερα το απόγευμα δείχνει πώς αυτές οι πράξεις προσβάλλουν τις αξίες που μεριζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε στο πλάι αυτού του κινήματος Είμαστε στο πλάι των θυμάτων του ρατσισμού και τη αστυνομική βία έτσι ώστε να δοθεί μια συγκεκριμένη απτή απάντηση στο αίτημα για σεβασμό και για ισότητα. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το γεγονός θα πρέπει να δούμε με καθαρό μυαλό την ιστορία μας και θα πρέπει να δούμε ότι αυτό το γεγονός παραπέμπει σε αιώνες επιβολής των λευκών επί των μαύρων στις ΗΠΑ και ανισοτήτων στην Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε ότι η ιστορία μας, η ευρωπαϊκή μας ιστορία, πάντα ήταν σαν το εκρεμές ανάμεσα στη βαρβαρότητα και τον πολιτισμό. Στην Ευρώπη, παρά τον ορθολόγο, παρά την, ε, το διαφωτισμό, έχουν γεννηθεί οι χειρότερες θεωρίες περί φυλών, περί ράτσας, για να μπορέσει αυτό να δικαιολογήσει από το ολοκαύτωμα μέχρι την απεικιοκρατία. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να εκριζώσουμε αυτό το κακό. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα βίας και οικονομικής βίας που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Διότι το διαπιστώνουμε. Οι ανισότητες, οι κοινωνικές ανισότητες εξακολουθούν να συνδέονται και με ρατσιστικές ανισότητες. Κύριε Πρόεδρε, τα σύμβολα όπως η μνήμη έχουν τη σημασία τους. Γι' αυτό λοιπόν στον αγώνα αυτό που δίνουμε θα πρέπει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως το ζητεί το ψήφισμά μας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η δουλεία είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ας δείξουμε λοιπόν όλοι πολιτισμό σήμερα. Ευχαριστώ. Από τους πήγε γραμμένους Φεράρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η βία δολοφονία του George Floyd προκάλεσε σε ολόκληρο το κόσμο δίκαιη η και προκάλεσε διαμαρτυρία. Μόνο δεν είναι μεμονωμένο επεισόδιο και απέναντι στη βία και το ρατσισμό δεν μπορεί κανεί να μείνει αδιάφορο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο με ειλικρίνεια, χωρί υποκρισία. Και πρέπει να αναχαιτήσουμε όλε τι μορφέ ρατσισμού, τι πιο προφανεί, τι βίε, αλλά και εκείνε που είναι λιγότερο εμφανεί και γι' αυτό πιο ύπουλε. Η αναφορά μου είναι σε αυτό το ρατσισμό που κρύβεται πίσω από την συμπάθεια ή κρύβεται από την φιλάνθρωπη προσέγγιση ή από την την ηθική υπεροχή που προδίδεται μετά από μια χρηστική χειραγώγηση ε, των όσων έχουν ε, μαύρο δέρμα. Ναι, στην Ευρώπη αυτό το φαινόμενο, ε, ε, έχουμε ακόμα πολλούς αγώνες να δώσουμε κατά αυτό το φαινομένο, ε, πολιτιστικές προκαταλήψεις, για να μπορέσουμε να εγκριθούμε σε όλους τα ίδια δικαιώματα, σε θέματα εργασίας, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, συμμετοχής πολιτικής και κοινωνικής. Και αυτό για κάθε μορφή και ε, διακρίσεων που μας απομακρύνουν εδώ και στα κρατημέλη. Ευχαριστώ. Γκονσάλες Πόνς, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι οι αντιρατσιστές είμαστε εδώ, από ό,τι φαίνεται, και ε, χαίρομαι γι' αυτό. Οι ρατσιστές είναι πάντα άλλοι. Όμως το πρόσωπο του George Floyd είναι ένας καθρέφτης όπου μπορεί να κοιταχθεί ο καθένα μα και τα, τα στρατόπεδα συγκέντρωση όπου εκατομμύρια Εβραίοι εξολοθρεύτηκαν έγιναν στην Ευρώπη. Δεν λύνεται το θέμα του ρατσισμού μόνο με νόμου, ούτε μόνο με προπαγάνδα, ούτε λύνεται ρίχνοντα αγάλματα, ούτε ε, προσβάλλοντα του αστυνομικού, ούτε κλείνοντα τα μάτια. Ο ρατσισμό δεν λύνεται με άλλο ρατσισμό. Θα πρέπει η κάθε συναγωγή, η κάθε η εκκλησία, η, το, ο κάθε μιναρές να είναι όλων μας Αυτά επιλύονται με κουλτούρα και με εκπαίδευση. Είναι η πιο παλιά πανδημία της ανθρωπότητας ο ρατσισμός εδώ και αιώνες και δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή τελικά να βάλουμε σε καραντίνα όσους έχουν πληγεί από τον ρατσισμό και να επενδύσουμε ό,τι χρειαστεί για να βρεθεί το σωστό εμβόλιο. Ευχαριστώ συνάδελφοι. κυρία Ινσίρε, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, το χρώμα, ε, η χώρα καταγωγής ε, ενός ανθρώπου ε, στους ρατσιστές προκαλούν φόβο και βλέπουμε τέτοια φαινόμενα ακόμα και στη δική μας Ήπειρο. Θέλουμε λοιπόν να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας ε, απέναντι σε όλους τους μαύρους που κάθε μέρα αντιμετωπίζουν ε, ρατσισμό ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αλλά μετανάστες και άλλες ομάδες αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αυτός ο δομικός ρατσισμός είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε καθημερινά σε συζητήσεις ε, με τους ε, συμπολίτες μας ε, το βλέπουμε αυτό. Τους αξίζει όμως κάτι καλύτερο θα πρέπει όχι μόνο να μιλάμε για κοινωνική πολυμορφία, αλλά θα πρέπει να καλύπτουμε όλους τους ανθρώπους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει μόνο να μιλάμε αντιρασιστικά, θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε αντιρατσιστικά ε, υπερψηφίζοντας το ψήφισμα αλλά και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει αντίστοιχα να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ραφαέλα, ένα λεπτό παρακαλώ. ο Τζορτζ Φλόιντ, η Ριάννα Τέιλορ, η Αντάμα Τροϊόρα ε, είναι όλοι θύματα και πολλά θύματα θα ακολουθήσουν εάν δεν ενεργήσουμε. Ε, ε, Συμπαρίσταμε σε οποιονδήποτε διαμαρτύρεται κατά της αστυνομικής βίας και, της, και των θεσμικών διακρίσεων. Δεν έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία. Θα πρέπει να προοδεύσουμε. Εάν ε, όμως οι πρόγονοί μου βλέπαν τη σημερινή κοινωνία, θα έβλεπαν ε, πράγματι ισότητα και ε, σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενωμένη στην πολυμορφία λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας κάνουμε λοιπόν αυτά που λέμε. Χρειαζόμαστε θεμελιώδεις αλλαγές στους θεσμούς μας, ώστε να εκπροσωπούν όλους τους πολίτες της Ευρώπης νέα γενιά Ευρωπαίων θέλουν και αυτοί μια θέση στο τραπέζι. Θα ε, φωνάξουν και θα ε, περάσουν τις θέσεις τους. Έχουν σημασία οι ζωές των μαύρων. Ευχαριστώ. Ριβιέρα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Φόντερ Λάιεν, το να χρησιμοποιούμε το θάνατο ενό ανθρώπου, ακόμα και τραγικό, για να μπορέσουμε ε, να μιλάμε για συστημικό ρατσισμό στην Ευρώπη είναι ανήθικο. Το να μιλάμε για αυτή τη δραματικό θάνατο του George Floyd εδώ είναι να φέρνουμε, να εισάγουμε στην ήπειρό μα ζητήματα τα οποία δεν μα αφορούν. Ο ρατσισμό και οι διακρίσει ε, οι ρατσιστικέ δεν είναι στι συνήθειέ μα. Εκατό μέτρα από εδώ ε, κάποιοι σπάγανε βιτρίνες. Εγώ προτιμώ αντί να ε, καταδικάζουμε του ε, προγόνου προγόνους μας να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, οι Ευρωπαϊκέ χώρε είναι αυτέ οι οποίε κατήργησαν τη δουλεία Γιατί να κατηγορούμε τι γαλλικέ ε, αστυνομικέ αρχέ για ρατσισμό θέλω να του υποστηρίξω ότι δέχονται όλο και πιο βάραβε επιθέσει. αντί να βάζω του ανθρώπου σε κατηγορίε ανάλογα με τη ράτσα του θέλω να μιλάω για την ε, ηθαγένεια και μόνο το να κλαίμε για κάποιον επειδή είναι μαύρο, αλλά δεν είμαστε ποτέ κατά του ρατσισμού, κατά των λευκών αυτό δεν είναι σωστό. Όλοι οι ρατσισμοί πρέπει να καταδικάζονται. Η κυρία Ετσπέργκερ Φοφανά για ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, εγώ ως μαύρη γυναίκα στην Ευρώπη ε, δεν έχω απλά συνειδητοποιήσει τη ρατσιστική πραγματικότητα στην Ευρώπη. Ε, την έζησα εδώ και 40 χρόνια. Αυτό που συμβαίνει στον κόσμο σήμερα είναι το αποτέλεσμα δομών Καταστολή απεικιοκρατικέ που υπάρχουν εδώ και εκατοντάδε χρόνια. Δεν πρόκειται για άτομα. Πρόκειται για ένα ρατσισμό συστημικό, θεσμοθετημένο, κατά των μαύρων και όλων των εθνοτικών μειονοτήτων. Δεν θέλω να μιλούμε μόνο για του αστυνομικού και την κατάρτισή του. Θέλουμε να, θέλουμε να υπάρξουν επιπτώσεις. Θέλουμε να υπάρξει δικαιοσύνη για όλου όσου έχασαν τη ζωή του, για όσου έχασαν του κοντινού του ανθρώπου και όσου έχουν ε, τραυματιστεί ψυχικά από την αστυνομία. Δεν αφορά μόνο τους Αμερικανούς μαύρους, όλους τους μαύρους ε, και αυτούς οι οποίοι πνίγονται στη Μεσόγειο λόγω μιας πολιτικής μετανάστευσης η οποία είναι ρατσιστική. Θέλω να είμαι σαφής. Όλες οι ζωές των μαύρων μετράνε, είτε είναι Ευρωπαίοι πολίτες είτε όχι. Των γυναικών, των τρανς, όλων. Ως καθηγήτρια είδα πως η ψυχή των παιδιών έχει καταστραφεί από την, το ρατσισμό είτε αυτός είναι ανοιχτό είτε υποχθόνιος. Μπαίνει στη ψυχή του παιδιού αυτό και οδηγεί σε μεγάλες αποτυχίες. Ήρθε η στιγμή να ξανανοίξουμε το διάλογο έτσι ώστε κανείς να μην μείνει εκτός και όπως είπε ο Μάρτιν Λουθερ Κίνγκ θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί σαν αδέρφια. Ιδάλλως θα πεθάνουμε όλοι σαν ηλίθιοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαμπάσκη για ένα λεπτό. Αξιότιμη πρόεδρε του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, όλε οι ζωέ έχουν σημασία. Αν αυτό το αρνηθούμε και αν πιστέψουμε πω μόνο οι ζωέ των ε, εκπροσώπων μία φυλή μόνο έχει σημασία, αυτό είναι ρατσισμό ήδη. Είναι επίση ρατσιστικό το να ισχυριζόμαστε ότι μόνο μία φυλή είναι αυτή που έχει σημασία. Παρακαλώ, επιλέξτε την πορεία σας. Είτε θα σέβεστε όλων τις ζωές, είτε θα είστε και θα υποστηρίζετε ρατσιστικές προσπάθειες. Όταν κανείς χρησιμοποιεί την προσωπική τραγωδία κάποιου για δικό του πολιτικό όφελος, αυτό είναι υποκρισία. Αυτή είναι η προσέγγιση των αριστερών, των κομμουνιστών, των ρατσιστών. Να θυμίσω τους συναδέλφους που φοράνε αυτά τα πλουζάκια σήμερα, πόσες ζωές καταστράφηκαν από τους Μπολσεβίκους και τους κομμουνιστές. Όταν ε, πιστεύεις ότι ο βανδαλισμός είναι το σωστό, αυτό είναι ήδη ε, επίση ρατισμός. Οι δικοί μου πρόγονοι ε, πολέμησαν ενάντια στους ε, Τουρκούς που υποδούλωσαν τους Βούλγαρους. Όμως δεν έσπαγαν μαγαζιά για να κλέψουν Το να κάνουμε κάποιον να αισθάνεται ένοχος λόγω της φυλής του είναι ύπουλο. Το να κάνεις κάποιον να αισθάνεται ε, ένοχος μόνο και μόνο της πρέλευσής του, αυτό είναι απαράδεκτο. Όχι μόνο δεν τρέπομαι για την πρέλευσή μου και το έθνος μου, αλλά αντίθετα είμαι περήφανος για το αρχαίο και ένδοξο κράτος το οποίο εκπροσωπώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ο Τζορτζ Φλόιντ πέθανε ενώ ε, τον κρατούσαν τρεις αστυνομικοί ε, στη ΣΥΠΑ και μεταξύ όλη η Ευρώπη κατηγορείται για ρατσιστική και καταστρέφονται αγάλματα διαφόρων πολιτικών ανδρών. Δεν καταπολεμούμε την αδικία με μια άλλη αδικία. Δεν δικαιώνουμε τον Τζορτ Φλόιτ βάζοντας στην θέση του ενόχου όλους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς. Κάθε χρόνο οι αστυνομικοί δίνουν τη ζωή τους για τη δική μας ασφάλεια και τη δική μας ειρήνη και εδώ δεν αναφέρονται καθόλου. Η δική του ζωή δεν ε, μετράει. Δεν καταπολεμάμε το ρατσισμό ρίχνοντας λάδι στη φωτιά των αμαλγαμάτων. Πώς ε, Λέει ότι η Ευρώπη αρχιασκεί ρατσιστικέ πολιτικέ σε όλους του τομεί. Εγώ δεν επιτρέπω να προσβάλλονται οι πολίτε που παντού στην Ευρώπη συμβάλλουν σε μεταναστευτικέ, οικονομικές, ε, υγειονομικέ πολιτικέ που είναι από τι λιγότερο ε, ρατσιστικέ και για όλου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα καταπολεμήσουμε το ρατσισμό μόνο μέσω διχασμών ρατσιστικών. Ε, η ιστορία της Ευρώπης εδώ και 24 χρόνια ότι εμείς δημιουργήσαμε την ιδέα του καθολικού. Το ξεχάσαμε αυτό και θα ψηφίσουμε ένα ψήφισμα που ξεχωρίζει τις μαύρες ζωές από τις υπόλοιπες. Κάθε ζωή έχει σημασία. For one minute, Madam Piri. President. Η κυρία Πύρη, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, χιλιάδες ανθρώπους είδαμε ε, στους δρόμους ε, που ζητούν ε, δικαιοσύνη για τον θάνατο του George Floyd. Επί 8 λεπτά αστυνομικός είχε καθυλώσει τον George Floyd στο έδαφος με το γόνατό του, παρότι φορούσε ήδη χειροπέδες. Και αυτή η πράξη δεν αποτελεί εξαίρεση και άλλοι μαύροι έχουν πεθάνει στα χέρια αστυνομικών. Και πολύ σωστά ο κόσμος ζητά δικαιοσύνη, όχι μόνο για τον George Floyd, αλλά και για όλες τις άλλες ε, αθώες ζωές που χάθηκαν. Και η έκκληση για δικαιοσύνη δεν είναι νέα, αλλά ε, το κίνημα είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Νέοι, γέροι, ε, μαύροι, λευκοί, όλοι ζητούν συστημική αλλαγή. Το αίτημα για φυλετική δικαιοσύνη έχει μεταφερθεί και στην Ευρώπη. Δεν αποτελεί αποκλειστικά ε, αμερικανικό πρόβλημα. Και στην Ευρώπη βλέπουμε στους ε, θεσμούς και στις κοινωνίες μας ε, τέτοιες διακρίσεις. Ε, έχουν μεγάλη σημασία και οι μαύρες ζωές ε, και γι' αυτό έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και ε, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τη συμφιλίωση εάν δεν αναγνωρίσουμε τις θηριωδίες του απεικιοκρατικού μας παρελθόντος. Μαζί θα καταφέρουμε να πετύχουμε την αλλαγή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Βάουτμανς. Εκτός μικροφώνου η κυρία Βάουτμανς. Εκτός μικροφώνου. Κακή αρχή έκανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, φανταστείτε την, ε, μια μητέρα της οποίας η κόρη Τη λέει κάθε βράδυ ε, «Δεν θέλω να έχω το χρώμα που έχω, θέλω να είμαι λευκή, μπορεί να με κάνεις λευκή». Φανταστείτε το, μπορείτε, εγώ μπορώ, διότι μου συμβαίνει. Έχω ε, έναν ε, πολύ όμορφο μαύρο σύζυγο και δύο πανέμορφα μαύρα παιδιά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή για μένα. Ο θάνατος ε, του George Floyd ας αλλάξει το παιχνίδι, ας ε, καταπολεμήσουμε την ε, ρητορική μίσους της διακρίσεις όλοι μαζί και περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Η Ευρώπη είναι η πιο προοδευτική ήπειρος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες. Αλλά κυρία Φόντερ Λάιεν τις τελευταίες μέρες είχα απογοητευτεί. Σήμερα ήταν πολύ ισχυρό το μήνυμά σα, αλλά τις τελευταίες μέρες ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πολύ ε, σιώπησαν. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα με δυνατή φωνή ε, και δεν πρέπει μόνο να μιλάμε, πρέπει να ενεργήσουμε κιόλα. Κάθε παιδί, οποιοδήποτε χρώματο θα πρέπει να μπορεί να μεγαλώνει με ασφάλεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Φέστ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο θεσμικός ρατσισμός στην Ευρώπη είναι κάτι περίεργο, διότι βλέπουμε ε, παράνομους μετανάστες ε, στην Ευρώπη και βλέπουμε να διαμαρτύρονται για δικαίωμα παραμονής. Ε, αυτό δεν έχει να κάνει με θεσμικό ε, ρατσισμό και βλέπουμε ε, και τις επιθέσεις, ε, βλέπουμε την επιθέσεις κατά της αστυνομίας από Τσετσένους. Βλέπουμε τι συμβαίνει σε διάφορες γειτονιές μεταναστών. Όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει τέτοιος ρατσισμός θέλουν να φέρουν εκατοντάδες χιλιάδες Αφρικανούς στην Ευρώπη. Αλλά αν ε, πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, σταματήστε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση επί 10 χρόνια και θα δείτε ότι θα εξαφανιστεί ο ε, υποτιθέμενος αυτός θεσμικός ρατσισμός ε, από τους θεσμούς της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ε, η κυρία Ντελπό Ο θάνατος του George Floyd ε, μας εξαγριώνει και αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι ένας μακρύς κατάλογος μαύρων νεκρών στα χέρια των Αμερικανών αστυνομικών εδώ και πολύ καιρό χωρίς να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη τις περισσότερες φορές. Σε πολλά επίπεδα λοιπόν υπάρχει ένας διαρθρωτικός ρατσισμός στο αμερικανικό σύστημα. Αλλά συστηματικός ρατσισμός υπάρχει στις δικές μας δημοκρατίες, στις ευρωπαϊκές, στις δικές μας κοινωνίες. Ευρωπαίοι πολίτες υποφέρουν καθημερινά για να έχουν πρόσβαση στην στέγαση, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση λόγω του χρώματος του δέρματός τους, λόγω της ενδεχόμενης, της υποτιθέμενης καταγωγής τους ή των γονέων τους. Δεν υπάρχει αρκετή διαφορετικότητα στους θεσμούς μας, εδώ στο Κοινοβούλιο, στις διοικήσεις μας, αλλά κυρίως κάποιοι από τους συμπολίτε μας έχουν να υποστούν καθημερινά ελέγχους από την αστυνομία αστυνομική βία ορισμένε φορές, έλεγχο ανάλογα με το χρώμα και εξακολουθούν οι κυβερνήσεις μας να αγνοούν το συστηματικό χαρακτήρα αυτών των ε, περιστατικών. Στη Γαλλία, στη Γερμανία και αλλού είχαμε νεκρούς σαν τον George Floyd και θα έχουμε και άλλους εάν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και αν δεν θέσουμε το ζήτημα αυτών των καθημερινών ελέγχων. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κυρία Ζόφτκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εξότιμοι συνάδελφοι. Ένας Αμερικανολιβανέζος συγγραφέας αναφέρεται στον ρατσισμό στην καθημερινότητά μας και λέει ότι ε, βίες ε, ε, επαναστάσεις με καλές προθέσεις έχουν οδηγήσει τελικά σε σκλαβοπάζαρα όπως το Τάτι Λιβύης ή την καταπολέμηση των Γεζίντιων στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να όλες οι χώρες οι οποίες δεν έχουν ένα σύστημα, ένα κράτος, μια αστυνομία να διαστρώσει την βία, ε, εκεί οδηγούνται. Είχαμε τέτοια παραδείγματα ε, μετά από επαναστάσεις που έριχναν ένα πρωταρχικό καθεστώς και έφεραν ένα άλλο και βεβαίως υπήρχαν, υπήρχε δίωξη για όσους ε, δεν συμφωνούσαν μαζί τους. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έτσι. Ο, η, η θανάτωση του George Floyd βεβαίως χάλα το αμερικανικό όνειρο στο οποίο έχουμε κατά νου. Μας ξύπνησε αυτό, αντιληφθήκαμε ότι παρεμφερείς ε, περιπτώσεις μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε μειονότητα, έτσι ώστε όλοι ε, να μπορέσουν να νιώσουν ίση και όχι πολύ του δεύτερης ε, διαλογής. Έχουμε, προσπαθούμε να εξηγήσουμε εδώ και πολύ καιρό ότι θα πρέπει να εξάγουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καλύτερο μοντέλο, ένα σχέδιο ειρήνης εδώ και 70 χρόνια. Οπότε πραγματικά ας εξάγουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο ανά τον κόσμο και όχι να και να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα, ε, διότι το μόνο σύστημα που λειτουργεί μέχρι τώρα είναι το δικό μα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριο Πιτσιόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να καταδικάσω κάθετα την υπερβολική βία που ασκήθηκε ενάντια στον Τζόρτζο Φλόιντ και το τραγικό της αποτέλεσμα δεν είναι το μόνο θύμα αυτού του θεσμικού ρατσισμού που δεν έχει εξαφανιστεί ενάμιση αιώνα μετά την κατάργηση της δουλείας και ε, ε, μετά από την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν τα πάμε καλά. Η οδηγία για την μη διάκριση είναι μπλοκαρισμένη εδώ και 12 χρόνια ε, στο Συμβούλιο και τα ε, ε, μαθήματα των παιδιών στα σχολεία πολύ συχνά ε, ε, παραβλέπουν πολλά από τα γεγονότα του παρελθόντος. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσιλωθεί στο να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη ΣΥΠΑ και να βασίζεται αυτή στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και, και την κοινή κατανόηση περί δημοκρατίας. Είναι ανάγκη να καταδικαστούν όλοι όσοι στην κοινωνία μας δουλεύουν υπέρ του διχασμού και του πολιτικού τυχοδιοκτισμού, αλλά ε, να ε, αγωνιστούμε αντίθετα για την ισότητα για όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, να μοιραστώ μαζί σας μια έκθεση που έγραψα όταν ήμουν 8 χρονών. Μόνικα Σεμέδο λέγομαι. Έχω όμορφο μαύρο δέρμα. Ε, η οικογένειά μου ήρθε από το Πράσινο Ακροτήρι στο Λουξεμβούργο. Σχεδόν έπρεπε να επιστρέψουμε στη... στο νησί μας, ε, διότι επρόκειτο να μας ε, απελάσουν από τη χώρα. Στην αρχή ήμουν στο Ινστιτούτο Σανφρόσα. Τώρα η μητέρα μας βρήκε ένα ωραίο μεγάλο διαμέρισμα. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με όλους. Στη δασκάλα μου άρεσε όταν είπα ότι είμαστε όλοι Λουξεμβούριανοι και προσέθεσε εκείνη ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Ωστόσο, το χρώμα δεν είναι αόρατο. Ε, έχω ε, ε, εμπειρίες ρατσισμού. 40 νεοναζί είχα γύρω μου κάποια στιγμή που μου φώναζαν συχνά με σταματάνε στο αεροδρόμιο. Κάποια φορά μάλιστα με είχαν ξεχωρίσει από τους φίλους μου επί ώρες. Ακούω συνέχεια παρατηρήσεις για τους μαύρους και μετά μου λένε «Ναι, αλλά εσύ είσαι εξαίρεση». Ε, αλλά τους λέω όχι, δεν είμαι. Και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα και να καλέσουμε το Συμβούλιο να ξεμπλοκάρει την οδηγία ε, κατά των διακρίσεων. Έχει σταματήσει η εποχή της σιωπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριος Φαντεντρίσε. Συνάδελφοι, η κάθε ε, ζωή έχει σημασία. Αυτό έχει γίνει ταμπού. Οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί και οι καθηγητές ε, προσπαθούν να μας ε, μεταφέρουν στην Ευρώπη ένα αμερικανικό πρόβλημα και να το χρησιμοποιήσουν για το δικό τους αριστερό θεματολόγιο. Ε, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν έχουμε εμεί κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε εδώ στην Ευρώπη πρόβλημα ε, βίασης βάρος ε, μαύρων. Δεν υπάρχει θεσμικός ρατσισμός πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν τόσε ευκαιρίε για του ανθρώπου αυτού. Δεν έχουμε εμεί προνόμια επειδή έχουμε λευκό δέρμα. Ε, Αντιθέτω, οι κοινωνίε μα είναι αποτέλεσμα σκληρή δουλειά. Τη σκληρή δουλειά των προγόνων μας και θέλουν να τα καταστρέψουν όλα αυτά και τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας θέλουν να παραποιήσουν. Δεν φταίμε εμείς που είμαστε αυτοί που είμαστε. Ε, ούτε λέμε σε κανέναν ότι πρέπει να αγωνατίσει επειδή έχει άλλο χρώμα. Ε, αυτός είναι ρατσισμός ει βάρο των λευκών. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για το ποιοι είμαστε. Συνάδελφοι, προτού προχωρήσουμε πρέπει να κάνω μια ανακοίνωση θα πρέπει να ξεκινήσει η πρώτη ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ε, τα έγγραφα που ανακοινώθηκαν ε, στην αρχή της σημερινής ε, συνόδου. 4.30 μέχρι τις 6 παρατέταρτο θα γίνουν οι ψηφοφορίες και θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδος με την, με την πρώτη μερική σύνοδο. Οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν με το συνηθισμένο τρόπο, αλλά δεν θα φαίνεται το πώς ψήφισαν, θα φαίνεται μόνο ότι ψήφισαν. Όλες οι ε, ψηφοφορίες θα είναι ονομαστικές, ε, αιτιολογήσεις ψήφου μπορούν να υποβληθούν γραπτός κατ' εξαίρεση. Ε, θα επιτραπούν μόνο εάν έχουν μέχρι 400 λέξεις. Κηρύττω λοιπόν την έναρξη της πρώτης ψηφοφορίας μέχρι τις 6 παρατέταρτο και στις 20 και 4, 8 και 4 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Ένα λεπτό έχει ο κύριος κύριος Καράς, Η, η εικόνα του, ε, ρατσιστικού, της, ε, του ρατσιστικού φόνου του ε, George Floyd ε, είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Και εδώ έχουμε ρατσισμό, έχουμε κοινωνική ανισότητα, φτώχεια, διακρίσεις, βία. Ε, στην αγορά στέγασης, ε, στους ε, χώρους εργασίας, στην εκπαίδευση. Έχουμε πολλή δουλειά. Εάν θέλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το, τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ε, η απαγόρευση των διακρίσεων, η φιλελεύθερη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, προστασία των ε, μειονοτήτων, ε, ο κορονοϊός. Όλα αυτά ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και κατά των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη, διότι μόνο έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε την δημοκρατία και τον αγώνα κατά του ρατσισμού και της ε, κοινωνικής ανισότητας. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, η κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν πολλοί συνάδελφοι για την αηδία του απέναντι στο ρατσισμό και τις διακρίσεις που εδώ και υπερβολικά πολλά χρόνια ε, μας απασχολεί. Έχουμε μάλιστα αύξηση των αριθμών των θανάτων κατά τη διάρκεια των συλλήψεων ή κατά τη διάρκεια ερευνών και αύξηση των ερευνών για τις ε, διακρίσεις. Υπάρχει βεβαίως η οδηγία κατά των διακρίσεων η οποία εδώ και 11 χρόνια δεν μπορεί να προχωρήσει διότι το Συμβούλιο δεν θέλει να προχωρήσει. Λέει ότι είναι πολύ ακριβό να αντιμετωπίσουμε όλε τι διακρίσει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Είτε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλάβουν τι διακυβεύεται εδώ, είτε θα πρέπει να υποβληθεί μια νέα νομοθετική πρόταση. Δεύτερον, το, το κείμενο του ψηφίσματό μα, κατά τη γνώμη μου, λείπει εδώ μία αναφορά στι μη κυβερνητικέ οργανώσει πολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων. Πρέπει να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε αυτέ τι ε, ε οργανώσει για να μην οδηγούμαστε στα άκρα. Επίση, θέλει ε, προσοχή όταν μιλάμε για στατιστικά στοιχεία εθνοτικά. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει πρόβλημα με το ε, συνταγματικό. Επίση, είναι κάποιε φωτογραφίε στι στιγμέ από τα στατιστικά στοιχεία και δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υποκατηστήσουν συγκεκριμένε προτάσει οικονομικέ και κοινωνικέ για να μειωθούν οι ανισότητε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Τόλερε έχει το λόγο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πολύ συχνά νεοφασιστικά, νεοναζιστικά κόμματα, εξαιρετικά μειονοτικά, εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε συζήτηση για να μπορέσουν να διαδώσουν τη ρητορική μίσου του. η σημερινή συζήτηση λοιπόν είναι πολύ σημαντική για να, για να θυμίσουμε κάτι κεφαλαιώδε για του συμπολίτε μα οι οποίοι υποφέρουν από το ρατσισμό στην Ευρώπη. Εμεί, οι Ευρωβουλευτέ, είμαστε εδώ για αυτού. Είμαστε εδώ για να σταματήσει αυτό ο λόγο ε, ο διχαστικός να μην, μιλάμε ε, σαν τον Τραπ, τον Μπολσονάρο ή τη Λεπέν και τον Σαλβίνη. Συζήτηση με τη συζήτηση, ψήφισμα με το ψήφισμα, δεν πρόκειται να κάνουμε τα, ένα βήμα πίσω απέναντι στις ρατσιστικέ και ξενοφοβικέ αυτές ιδεολογίε. Το ευρωπαϊκό σχέδιο βασίστηκε στη συμφιλίωση. Είναι η καλύτερη ασπίδα απέναντι στα άκρα. Ε, στο κέντρο ε, της Ευρώπης μας ε, βλέπουμε πόσο ενωμένοι είμαστε, όσο, όσο είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε πιο όμορφοι ή είμαστε πιο δυνατοί. Thank you. I now give the floor to the Commission. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει, παρακαλώ κυρία Γιούροβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Ήταν προφανές νομίζω από αυτά που είπε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, νωρίτερα δεν υπάρχει θέση για τον ρατσισμό στην Ένωσή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει όλα τα περιστατικά ρατσισμού, ξενοφοβίας, αλλά καταδικάζουμε τη βία γενικά, από όπου και αν προέρχεται. Και η αστυνομία βεβαίως θα πρέπει και αυτή να κάνει την απαιτητική δουλειά της. Πάντα εντός συγκεκριμένων και σαφών ορίων η επιλεκτική ε, προσέγγιση ανάλογα με το χρώμα κάποιου δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ανεκτό. Το παρατηρητήριο το ευρωπαϊκό έχει εκδώσει πολύ χρήσιμε κριτικέ γραμμέ που μπορούν να αποτελέσουν ε, αποτελέσει υλικό κατάρτιση για τι αστυνομικέ αρχέ αλλά και για τι άνοπλε δυνάμει. Για να αποφεύγουμε ακριβώ αυτού του είδου την κακομεταχείριση. Ναι, βεβαίω και έχουν σημασία οι ζωέ των μαύρων. Όλε οι ζωέ έχουν σημασία όλοι, μαύροι, λευκοί, οποιοδήποτε άλλο άλλης εθνικότητας ή φυλής και χρώματος πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν ε, στην κοινωνία μας και να αναζητούν την ευτυχία στις κοινωνίες μας. Πρέπει όλοι να μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας μην ανησυχείς, κανείς δεν πρόκειται να σε σκοτώσει λόγω του χρώματος του δέρματός σου. Όμως αυτή η συζήτηση έχει να κάνει και με το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Έχουμε πολλά δεδομένα από την Υπηρεσία Θεμελών Δικαιωμάτων στην τελευταία έκθεσή της που δείχνει σαφώς ότι τα άτομα που έρχονται από μειονότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν βία, εθνική, ρατσιστική διάκριση σε διάφορους τομείς της ζωής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως υπάρχει νομοθεσία, όμως η νομοθεσία δεν φτάνει. Έχουμε την νομοθεσία σε ψηλότερο επίπεδο. Η πρόεδρος Φόντε Λάιεν το ανέφερε. Η Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων. Έχουμε, εδώ και 20 χρόνια έχει ε, εγκριθεί η οδηγία για την ισότητα μεταξύ των φυλών και υπάρχει και απόφαση πλαίσιο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Έχουμε λοιπόν νομοθεσία. Τα πράγματα όμως εξακολουθούν να είναι ανησυχητικά. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε, να εγκρίνουμε την οδηγία ίσης μεταχείρισης. Έγινε αναφορά σε αυτήν εδώ και είναι κρίμα που και είναι ντροπή που περιμένουμε 12 χρόνια για να εγκρίνουμε αυτή την οδηγία και βασίζομαι στη συνάδελφο την Έλενα Ντάλη ε, να, δείξει, να επιδείξει αποφασιστικότητα για να πείσει τα κράτη-μέλη να πάρουν μια ομόφωνη απόφαση διότι αυτή η οδηγία απαιτεί ομοφωνία. Είναι τόσο σημαντική, δεν είναι τόσο σημαντική βέβαια η διαρρύθμιση αλλά η εφαρμογή της. Διότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με στερεότυπα, έχει να κάνει με προκαταλήψεις, χρειάζεται λοιπόν και ευαισθητοποίηση, χρειάζεται εκπαίδευση, παιδεία, κουλτούρα, χρειάζεται και χρειάζονται και κάποια σώματα ισότητας τα οποία έχουν ενισχυθεί ήδη το περασμένο χρονικό διάστημα. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη ε, έτσι ώστε όσοι υπόκεινται σε διακρίσεις να έρθουν να το καταγγείλουν, διότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Πολλές φορές δεν γίνονται αυτές οι αναφορές. Την ερχόμενη εβδομάδα θα επικαιροποιήσουμε και τη στρατηγική μας για την εφαρμογή της οδηγίας ε, των δικαιωμάτων των θυμάτων. Δεν θα είναι δηλαδή τα θύματα να ε, βγουν μπροστά, αλλά είναι αργά βέβαια ε, να επιλύνουν για να επιληθεί το πρόβλημα των θυμάτων όταν πια έχει γίνει το κακό. Έχουμε προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και ειδικέ ε, καταστάσεις σε διάφορες χώρες. 15 ε, χώρες της Ένωσης έχουν αυτή τη στιγμή ε, στρατηγική του ρατσισμού. Θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Επίσης, ε, εργαστήκαμε πολύ περισσότερο σε ψηφιακό επίπεδο είδαμε μεγάλη αύξηση του μίσους ε, διαδικτυακά. Έχουμε κάποια εργαλεία για την αντιμετώπιση του, της ρητορικής μίσους, όμως πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα προς την κατεύθυνση αυτή. Φέτος, ε, εφόσον γνωρίζετε το πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν, θέλουμε να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Μελών Δικαιωμάτων, να εγκρίνουμε μια στρατηγική για την εφαρμογή της χάρτας αυτής. Θα επικαιροποιήσουμε και τις στρατηγικές για την ε, ένταξη των Ρωμά και των, ε, της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και θα ξέρετε επίσης ότι στην πρόταση για τον προπολογισμό για την ε, νέα γενιά, New Generation, ξέρουμε ότι πρέπει να έχει μια διάσταση κοινωνική που να μην αφήνει κανέναν απ' έξω έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια. θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο είναι και αυτό ε, εδώ για να βοηθήσει τις μειονότητες. Ε, δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα, δεν είναι θέμα πολιτικών χρώματων. Μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα. Το να μπορεί κάποιο να την χάνει ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από το σεξουαλικό του προσανατολισμό, από τη θρησκεία του, το χρώμα του. Εμεί οι πολιτικοί θυνοντέ πρέπει να δεχτούμε μεγαλύτερη πίεση. Ε, πρέπει όσοι μπορούν να επηρεάσουν ε, το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, ε, πώς προσεγγίζουν οι άνθρωποι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν στις μειονότητες, να βρεθούν πίεση και πρέπει ε, να μην διαδίδουμε ε, έναν λόγο ρατσιστικό ε, για να έχουμε κάποιο πρόσκαιρο πολιτικό όφελος. Όπως είπε ο Σλαβόντερ Λάιεν, επιβεβαιώνω κι εγώ ότι δεν ξέρω πώς είναι να νιώθει κανείς ότι είναι μαύρος. Δεν έχω υποστεί διακρίσεις. Κανενός τύπου. Γι' αυτό λοιπόν όταν πάω στα κράτη-μέλη και μιλάω στους νέους Ρωμά, πάντα ρωτάω αυτούς που μπόρεσαν να τελειώσουν το σχολείο, το γυμνάσιο και τους ρωτάω πώς τα καταφέρατε. Διότι ξέρω ότι το σημείο αφετηρίας για αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό των δικών μου παιδιών και πολλών από εδώ. Και όλοι πάντα μου λένε ότι υπήρξαν τρεις στιγμές. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να ζήσω όπως ζούσαν οι γονείς μου, θέλω να κάνω κάτι περισσότερο, θέλω να βγω από αυτή την παγίδα της φτώχειας και το δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι ότι μας λένε ότι έπρεπε να βρω κάποιον να με βοηθήσει. Όσοι τα κατάφεραν πάντα βρήκαν κάποιον να τους βοηθήσει, είτε στην τοπική τους κοινότητα, ο δήμαρχος, μια μη κυβερνητική οργάνωση, κάποιο διευθυντή σχολείου, χωρίς αυτούς δεν θα τα είχαν καταφέρει. Μηδενική λοιπόν ανοχή απέναντι στι διακρίσει, μηδενική ανοχή απέναντι στο ρατσισμό, αλλά αυτό δεν αρκεί πρέπει να έχουμε και ενεργή δράση για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να βγουν από την παγίδα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο Υπουργός Μπερνέτς για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, χρήσιμη και πολύ ε, συγκινησιακή συζήτηση, συγκινητική. Ε, ναι, Σα ευχαριστώ όλους. Πιστεύω πως οι θεσμοί μας είναι στην ίδια γραμμή όσον αφορά αυτά τα βασικά θέματα. Σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, ισότητα, κράτο δικαίου. Αυτά είναι τα θεμέλια τα ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο δεσμεύεται στη στήριξη αυτών των αξιών ε, και στη στήριξη των εξωτερικών μα σχέσεων με με τους εταίρους μας όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες. Σας διαβεβαιώ για ακόμη φορά ότι το Προεδρείο και το Συμβούλιο γενικά απορρίπτουν κάθε είδος ρατσισμού, ρατσιστικής διάκρισης και στηρίζει τον αγώνα για την δικαιοσύνη. Έχουμε ε, νομοθεσία που πρέπει να συμπληρωθεί από την υλοποίηση, την εκτέλεση, την εφαρμογή και με σημαντικά μέτρα στην παιδεία, στη δημόσια συζήτηση ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση πολύ στενά, να άκουσα προσεκτικά τις απόψεις σας. Πρέπει να ακούσουμε τις φωνές των νέων ανθρώπων που ειρηνικά ζητούν καλύτερη, καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ συνάδελφοι πέρα στη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει την Παρασκευή. Ehm, e Σας Σα ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη, τώρα έχουμε κοινή συζήτηση για την προετοιμασία τη συναντρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για τι συστάσει για τι διαπραγματεύσει για τη νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και τη Βόρεια Ιρλανδία. Ε, θα υπάρξουν δηλώσεις Συμβουλίου και Επιτροπής όσον αφορά την προπαρασκευή της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Μετά θα ακούσουμε τον Πύρη Γιάνσεν ε, για τα θέματα Brexit. Να θυμίσω ότι αυτή η συζήτηση δεν σε αυτή τη συζήτηση προβλέπεται το ΚΑΤΣΔΙΑ και δίνω το λόγο στην Υπουργό Μπερνίτσε. Παρακαλώ, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, ο κορονοϊός συνεχίζει να ε, δημιουργεί ε, περίεργες προκλήσεις για τις κοινωνίες μας. Τώρα αντιμετωπίζουμε το εξή επίγον έργο, την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Πρέπει να στηρίξουμε τις περιφέρειες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ε, για βιώσιμη ανάκαμψη σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ε, θα πρέπει να φροντίσουμε και άλλες προτεραιότητες ε, της Ένωσής μας όπως είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Και γι' αυτό το σχέδιο ανάκαμψης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που παρουσιάστηκε τέλη Μαΐου είναι τόσο σημαντικό και γι' αυτό θα είναι και το βασικό επίκεντρο των προσπαθειών μας τις επόμενες εβδομάδες. Καλούμαστε να συμφωνήσουμε όχι μόνο πάνω στα εργαλεία για την ανάκαμψη, αλλά και το συνολικό πολιετές ε, πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό ε, δεν είναι λίγο. Ε, το Συμβούλιο έχει κινητοποιηθεί για να πετύχει αυτή την κοινωνική προσπάθεια το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο ε, θα έχει βιντεοδιάσκεψη την Παρασκευή και ο πρόεδρος του Συμβουλίου θέλει να δώσει στους ηγέτες τη δυνατότητα να συζητήσουν ε, διάφορες πτυχές και να προετοιμάσουν τη διάσκεψη κορυφής που ελπίζουμε ότι θα γίνει διαζώσεις. Ενώ ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησε τις πολιτικές συζητήσει σε υψηλό επίπεδο ε, μετά από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ξεκινήσαμε αμέσω ε, και τι εργασίε εντό του Συμβουλίου. Η Κροατική Προεδρία έχει οργανώσει μια σειρά συναντήσεων και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο, ώστε οι αντιπρόσωποι να μπορέσουν να εξετάσουν ε, και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ε, πάνω στα διάφορα τμήματα της δέσμης μέτρων. Αυτή η τεχνική και πολιτική δουλειά είναι απαραίτητη για να ανοίξει το δρόμο για τη συζήτηση των ηγετών. Αυτές οι συζητήσεις στο Συμβούλιο έγιναν με θετικό κλίμα και ήδη έχουν γίνει πολλές απαραίτητες διευκρινήσεις και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχέδιο ανάκαμψης ε, είναι μία δέσμη μέτρων ε, και ε, η συνεχής συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι, συνεχίσει να είναι ζωτική σημασίας εάν θέλουμε να τεθεί σε ισχύ η δέσμη μέτρων ήδη τον Ιανουάριο του 2021. Φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λοιπόν είναι να παράσχει τον πολιτικό προσανατολισμό πριν το καλοκαίρι και να ζητήσει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας είμαστε ειλικρινεί, ε, είναι πολύ φιλόδοξη η προσέγγιση αυτή. Μαζί όμως ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο και το ε, σχέδιο ανάκαμψης να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας ενώ το σχέδιο ανάκαμψης θα είναι ε, το επίκεντρο των συζητήσεων των ε, ηγετών την Παρασκευή, θα ασχοληθούν και με άλλα θέματα. Ο πρόεδρος Μισελ θα ενημερώσει τους ηγέτες ε, σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε πετύχει τόσα όσα ελπίζαμε. Αυτό ισχύει σε όλους τους ζωτικούς τομείς. Συνθήκες ίσου ανταγωνισμού, διακυβέρνηση, εσωτερική ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εξωτερική ασφάλεια ε, είναι επίσης σημαντικά θέματα και πολύ σωστά στις συστάσεις σας ε, έχετε αφιερώσει χώρες αυτά. Εφόσον ε, η ε, κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ε, θέλει να δεχτεί παράταση της μεταβατικής περίοδου, μας περιμένουν τέσσερις μήνες έσπληρων διαπραγματεύσεων. Το γεγονός ότι έχουμε μείνει ότι έχουμε τελικά τόσο λίγο χρόνο μπροστά μας δεν αποτελεί επιλογή ούτε του Συμβουλίου ούτε του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να το σεβαστούμε όμως η ε, πολιτική δήλωση που ε, καθοδηγεί τον διαπραγματευτή μας ε, αποτελούν τις προϋποθέσεις, αλλά όλα εξαρτώνται και από τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διαλέξει είτε να συμμορφωθεί με τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχει πρόσβαση στην εσωτερική αγορά ή να διαλέξει το δικό του δρόμο ε, κάτι που θα ε, περιορίσει το πεδίο εφαρμογή ε, τη εταιρική σχέση. Πιστεύουμε ότι η διαπραγματευτική εντολή που υιοθετήθηκε πέρσι το Φεβρουάριο από το Συμβούλιο και που αντικατοπτρίζεται και στο ψήφισμά σα παρέχει επαρκή ευελιξία ώστε να βρεθεί μια λύση στον λίγο χρόνο που έχουμε μπροστά μα. Γι' αυτό στηρίζουμε και τη θέση των διαπραγματευτών να ε, εντείνουν ε, το ρυθμό των ε, διαπραγματεύσεων το καλοκαίρι, ώστε τον Οκτώβριο να έχουμε ένα σχέδιο συμφωνία εταιρικής σχέσης. Πριν κλείσω, να πω, όπως λέτε και εσείς στο σχέδιο σύστασή σας, ότι υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης. Περιτεύει να πούμε ότι η πρόοδος θα ε, πρέπει να συνοδεύονται, να ακολουθούν και την πρόοδο στην ε, Συμφωνία Αποχώρησης. Σας ευχαριστώ. Να χαιρετήσω και τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτ ε, ε, και να δώσω το λόγο μέσα στην Πρόεδρο της Επιτροπής που ακόμα μια φορά θα ευχαριστήσω που είναι σήμερα παρούσα. Οι διαπραγματεύσεις με τον Ηνωμένο... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι διαπραγματεύσεις με τον Ηνωμένο Βασίλειο ανέκαθεν ήταν δύσκολε και δεν μα απογοήτευσαν ούτε αυτή τη φορά. Ε, τη Δευτέρα ο πρόεδρος όλοι, ο κύριος Μισελ και εγώ το συζητήσαμε και είδαμε ότι ο Πρωθυπουργό της Βρετανίας δεν επιθυμεί να παρατείνει την περίοδο πέρα από αυτό το φέτος. Ε, εμείς ε, ήμασταν διαθέσιμοι, αλλά χρειάζονται δύο για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα είμαστε στο ίμιση των διαπραγματεύσεων και πέντε μήνες μόνο στη διάθεσή μας. Αλλά Σίγουρα δεν έχουμε φτάσει το ίμιση της συμφωνίας, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε σε συμφωνία, θα είμαστε επικοδομητικοί όπως ήμασταν ανέκαθεν και είμαστε έτοιμοι να είμαστε και δημιουργικοί για να βρούμε κοινό έδαφος εκεί που φαίνεται πως δεν υπάρχει. Αυτό που δεν είμαστε έτοιμοι όμως να κάνουμε είναι να βάλουμε και να αφισβητήσουμε τις αρχές μας και την ακεραιότητα της Ένωσης, γιατί είναι δικό μας καθήκον να προστατέψουμε το συμφέροντα των πολιτών μας. Ο Μισελ Μπαρνιέ έκανε εξαιρετικό έργο το τελευταίο μήνα. Έχει πολλές φορές προσπαθήσει καταρχάς ισότιμο πεδίο έχουμε τέσσερα ζητήματα το βασικό θέμα εδώ είναι, είναι δίκαιος ανταγωνισμός μπορούμε να ανταγωνιστούμε με τις βρετανικές εταιρείες και οι δικές μας εταιρείες είναι εξαιρετικέ, αλλά όχι ο διαταγωνισμός προς τα κάτω. Ας πούμε η περιβαλλοντική προστασία και τα πρότυπα αυτής θα ήταν κάτι το αρνητικό το να οπισθοδρομήσουμε ενώ μπορούμε να προχωράμε προς τα υψηλότερα πρότυπα. Δεύτερον, αλληλεία. Δεν αφιερωθεί κανείς την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου στα υδατά του. Φυσικά, αλλά ζητάμε προβλεψιμότητα και εγγυήσει ε, για τους αλληλείς μας που αλλιεύουν εδώ και δεκαετίες σε αυτά τα ύδατα. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνολική εμπορική συμφωνία χωρίς την αλληλεία, χωρίς ισότιμο πεδίο ή χωρίς ισχυρούς μηχανισμούς διακυβέρνησης. Διακυβέρνηση μπορεί να ακούγεται κάτι το πολύ γραφειοκρατικό, αλλά δεν είναι. Είναι... Ε, είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε ότι αυτά που έχουν συμφωνηθεί θα γίνουν και στην πράξη. Και έπειτα, ε, αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Θέλουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δεδομένα των πολιτών μας να είναι προστατευμένα σε κάθε περίπτωση και γι' αυτό και περιμένουμε να υπάρχει ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και που αυτό έχει σημασία. Αυτή είναι στόχη όχι μόνο στι συζητήσει μα με τον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε οποιαδήποτε σχέση με οποιονδήποτε εταίρο γιατί ακριβώς ε, ε, αυτά είναι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δίκαιος ανταγωνισμός, αυξανόμενες κοινωνικές προδιαγραφές, προστασία κράτους δικαίου. Αυτό είμαστε και αυτό δεν θα το αλλάξουμε, ούτε πρόκειται να αλλάξει. Ε, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την ενότητα που έχουν δείξει όλοι οι θεσμοί και για την πλήρη στήριξη αυτή, σε αυτή τη διαδικασία. Θα είναι ακόμα πιο σημαντικό στην επόμενη φάση. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πού θα βρίσκονται αυτές οι διαπραγματεύσεις στο τέλος του έτους, αλλά είμαι βεβαία ότι εμείς θα έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να φτάσουμε σε καλή συμφωνία και να ξεκινήσουμε καλά με το Ηνωμένο Βασίλειο ως εταίρο μας. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, δυστυχώς οι Βρετανοί φίλοι μας ε, είναι διατεθειμένοι να πάνε ένα βήμα πίσω. Θέλουν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή αγορά. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες ε, ώστε να περιορίσουμε τις συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη έχουμε και την οικονομική και, και κοινωνική κρίση που αποτελούν σημαντική πρόκληση. Με ε, το Next Generation EU έχουμε μια ε, πολύ τολμηρή ε, πρόταση. Είναι μια ισορροπημένη πρόταση. Βοηθάει τις χώρες που είχαν πολλούς ασθενείς και νεκρούς αλλά και τις χώρες που εμέσως πλήγησαν λόγω της, λόγω των αλυσίδων τροφοδότησης της παραγωγής κλπ. Ε, είναι ένα πρόγραμμα που θα επιταχύνει την οικονομία, θα ενθαρρύνει την ε, έρευνα και την ανάπτυξη. Και αν ε, τα κάνουμε όλα σωστά, τότε θα έχουμε όχι μόνο αναβίωση της εσωτερικής αγοράς, αλλά θα έχουμε και αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας εδώ και καιρό χρειαζόμασταν εξυγχρονισμό. Δεν θέλουμε λοιπόν να επανέλθουμε στην κατάσταση πριν την κρίση. Θέλουμε να έχουμε μια σύγχρονη οικονομία ε, και καινοτόμα οικονομία. Ε, το πρόγραμμα Next Generation EU είναι και μια σύμβαση ανάμεσα στις γενιές θα πρέπει να κάνουμε μια τεράστια επένδυση για να ξεφύγουμε από την κρίση. Θα δημιουργήσουμε όμως μια πιο βιώσιμη, ε, μια καλύτερη, μια πιο ψηφιακή Ευρώπη. Ε, άλλα μέρη του κόσμου παρακολουθούν ε, στενά τι γίνεται εδώ στην Ευρώπη και ακριβώς γι' αυτό το πρόγραμμα αυτό στόχο έχει ε, να ενισχύσει τη θέση της ε, Ευρώπης ε, και στην περιοχή άμεσης γειτονίας μας αλλά και στην ευρύτερη διεθνή σκηνή. Θέλουμε μια Ευρώπη που να είναι πιο ανθεκτική σε παγκόσμιες κρίσεις και να αποτελεί ασφαλή πατρίδα για τις επόμενες γενιές. Κυρίες και κύριοι, επανειλημμένα είχα τη δυνατότητα να εξηγήσω σε εσά και το πολιτες πλαίσιο και το Next Generation EU. Αυτό θα το κάνουμε και την την Παρασκευή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, το σχέδιο αυτό γενικά έγινε θετικά αποδεκτό. Ε, αντιδράσεις ε, πολύ θετικές είδαμε και από τις αγορές. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό δεδομένου του μεγέθους του εγχειρήματος και εδώ στο Κοινοβούλιο θα το συζητήσουμε αναλυτικά για μένα είναι σημαντικά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η σωστή σχέση με τις εθνικές προσπάθειες μεταρρυθμίσεων και οι ευρωπαϊκές μας προτεραιότητες, ιδιαίτερα η Πράσινη Συμφωνία, η ψηφιοποίηση και η ανθεκτικότητα και τρίτον η σημασία των νέων ίδιων πόρων ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρόθεσή μου να έχω αναλυτικές συζητήσεις μαζί σας. Ε, δεν ε, μπορούμε να καθυστερήσουμε. Ας ε, καταβάλουμε λοιπόν μαζί μια προσπάθεια για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και τώρα το λόγο έχει η συγκεκριμένη κυρία Κάτι Πύρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την κυρία, τον κυρία Φόντερ μας πήρε τόσο καιρό να φτάσουμε σε μια συμφωνία με τους Βρετανούς. Τώρα έχουμε, έχουμε τη μεταβατική περίοδο, τέσσερις γύρους διαπραγμάτευσης και πάλι σε διέξοδο έχουμε βρεθεί. Τι χρειαζόμαστε τώρα λοιπόν. Χρειαζόμαστε νέα ενέργεια, έναν νέο δυναμισμό, να αλλάξει η προσέγγιση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, την περσμένη Δευτέρα δεν μάθαμε και πολλά πράγματα ε, ελπίζουμε παρόλα αυτά ότι η ομάδα υψηλού επίπεδου αυτό δημιούργησε. Ε, δημιούργησε ένα νέο δυναμισμό. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο μια συνολική συμφωνία σημαίνει εγγυήσει για δίκαιο ανταγωνισμό με σαφεί κοινωνικέ. ε, στοιχεία κοινωνική προστασία, περιβαλλοντική προστασία, και αυτό συμφώνησαν στην πολιτική δήλωση με τον κύριο Τζόνσον ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρελθόν και αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα. Μηδενικέ ποσοστώσει. ε, ε, μηδενικές, ε, ε μηδενική δασμή, οπότε μηδενικό ντάμπινγκ. Αυτό είναι προς, όφελ, προς ε, συμφέρον και των Ευρωπαίων πολιτών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμείς καλωσορίζουμε τον ενθουσιασμό και την εφορία του κυρίου Τζόνσον πρόσφατα ε, σε μια προσπάθεια να φτάσει μια συμφωνία εντός έξι εβδομάδων. Όμως ο Πρωθυπουργός δεν μας εξήγησε πώς θα γίνει αυτό και περιμένουμε ανυπομονησία να ακούσουμε τις λεπτομέρειες. Τους τελευταίους μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιδείξει τη δέσμευσή του, έχει αναλάβει τι ευθύνε του, τις ευθύνες του για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Με την ομάδα των Ισμού του Μενού Βασιλείου, δύο επιτροπέ, 17 επιτροπέ που γνωμοδοτούν, έχουμε μια ε, μοναδική ε, διαδικασία με την έκθεση του Κρίστοφ Χάνσεν και εμού, όπου και αυτό δείχνει πόσο σοβαρά παίρνουμε το ρόλο, παίρνουμε το ρόλο μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην ομάδα υψηλού επίπεδου ε, θα παρουσιαστεί και η θέση μα στην ομάδα υψηλού επίπεδου από τον Πρόεδρο. Και χαίρομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενωμένο ε, με ένα ισχυρό κίνημα, κίνημα και κείμενο, ένα σαφέ πολιτικό μήνυμα, ένα απλό μήνυμα. Ναι, θέλουμε συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να δεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία. Υπάρχουν προποθέσει. Θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να σεβαστεί τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να σεβαστεί την πολιτική δήλωση και να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή τη συμφωνία. Ε, ε, αποχώρησης. Το γεγονός ότι θέλει να κρατήσει τα δικαιώματα και τα ωφέλη του κράτους μέλους χωρίς να έχει πλέον καμία υποχρέωση το βασίλειο δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι λογικό λοιπόν, εάν θέλει κανείς να έχει πρόσβαση στην, σε μια αγορά 450 εκατομμυρίων πολίτων, αυτό συνεπάγεται κάποιες προϋποθέσεις. Το η κυβέρνηση του μένου Βασιλείου πήρε μια συνειδητή απόφαση να φύγει από την ενία αγορά. Εμεί το σεβόμαστε αυτό. Αλλά πρέπει να το σεβαστεί και το ίδιο το Μένο Βασίλειο. Και χωρί ε, ίσο επίπεδο ε, ευκαιριών στον τομέα τη αλληλεία, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια, κάποιο δικασμό μεταξύ των πολιτών του ΕΒ Βασιλείου και τη Ευρώπη. Ο δικασμό που υπάρχει μεταξύ, είναι μεταξύ αυτών που έχουν ένα όραμα, θέλουν να φτάσουν σε μια συμφωνία και ενό Βρετανικού, μια Βρετανική κυβέρνηση που ουσιαστικά υπαναχωρεί σε σχέση με τι δεσμεύσει του και εξακολουθεί να βάζει την ιδεολογία πάνω από το συμφέρον των συμπολιτών του. Ο δρόμο μπροστά μα είναι σαφή. Εμεί είμαστε ενωμένοι στο αίτημά μα για μια φιλόδοξη συνολική εταιρική σχέση με σαφεί προποθέσει, κόκκινε γραμμέ, όπω μόλι αναφέραμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και εξακολουθεί να είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί καλόπιστα, επικοδομητικά σε ένα πνεύμα εμπιστοσύνη. Και ο κύριος Μπαρνιέ βεβαίω έχει την πλήρη υποστήριξή μα. Και ελπίζουμε τελικά να έχει έρθει η ώρα ο κύριος Τζόνσον και το, η κυβέρνηση του ΕΒ να έρθει και να τα βρούμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ την κυρία Πύρη. Τώρα ο κύριος Άνσε Χάνσεν έχει το λόγο, συνεισηγητής. Ευχαριστώ ε, κύριε Φοντερ Λάιεν, κύριε Μπερνία, αγαπητοί συνάδελφοι, τέσσερα χρόνια πριν, στις 23 Ιουνίου του 2016, έλαβε χώρα το δημοψήφισμα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Έκτοτε είχαμε τέσσερα χρόνια δραματικά, ε, όπου οι Βρετανοί άρχισαν να καταλαβαίνουν σιγά σιγά τι σημαίνει ε, το να αποχωρούν από τη μεγαλύτερη ενία αγορά ε, στον κόσμο μετά από 40, μετά δεκαετίες και το, και το καλύτερος χώρος που υπάρχει ε, με όλες τις ατελείες του. Ε, δεν είναι πλέον βιώσιμο το σχέδιο των Βρετανών. Ε, δεν ξέρουμε και αν ήταν ποτέ. σε ένα κόσμο που είναι εκ νέου πολλωμένο και οι οργανώσεις οι οποίες είναι υπέρ της πολυμερής προσέγγισης βρίσκονται υποπίεση και με τον κορονοϊό ε, το πολιτικό Brexit έλαβε χώρα το περσμένο Ιανουάριο, το οικονομικό Brexit όμως ε, εξακολουθεί ε, να είναι αβέβαιο στο τέλος του έτους. Μετά την ιδεολογική απόσταση του Βασιλείου να μην παρατείνει τη μεταβατική περίοδο. Το μήνυμά μας στις διπραγματεύσεις αυτές είναι σαφέστατο. Το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τον διαπραγματευτή, τον κύριο Μπαρνιέ. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να φτάσει σε μια συμφωνία που θα φασίζεται μόνο στο προηγούμενο. Στα προηγούμενα. Όμω οι τομεί όπω οι οικονομικέ υπηρεσίε, ή επαγγελματικέ δεξιότητες. Εδώ πάμε πολύ πέρα από αυτά που έχει παραχωρήσει ε, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Δημόσιες προμήθειες, ε, δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί στην πολιτική δήλωση. Ε, δεν μιλάει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Μένο Βασίλειο. Όταν διαπραγματεύεται όμως με άλλους εταίρους το κάνει, όπως παραδείγματος χάρη στις ε, διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Ε, και εκεί περιλαμβάνονται και δημοσίες προμήθειες, εκεί περιλαμβάνονται και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ περίεργο αυτό, μεγάλη έκπληξη για μας. Χρειάζεται λοιπόν ένα ίσο πεδίο ευκαιριών, χρειάζεται συμφωνία για την αλληλεία, ιδάλω δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, να είμαστε σαφεί. Όταν λέμε ένα πεδίο, ε, ένα ίσο πεδίο ευκαιριών, δεν λέμε να αντιγράψουμε του κανόνε μα απλώς να έχουμε ένα κοινό σημείο αφετηρίας το οποίο δεν θα, πάμε, δεν θα επαναχωρήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν ισοδύναμα, όχι οι ίδιοι κανόνες για όλους. Εμείς υποστηρίζουμε την προσέγγιση της Κομισιόν έτσι να έχουμε μια συνολική συμφωνία. Δεν δεχόμαστε την τομεακή προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι η σαλαμοποίηση οδηγεί συνήθως σε μια κακή μακαρονάδα. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βεβαίω θα πρέπει να είναι το, το σημείο αναφορά μέσω του κοινωνικού δικαίου. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όσο κυρία και το Βασίλειο στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να ευχαριστήσω την συνεισηγήτρια, την Κέιτι Πέρι. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία ε, στην προσπάθεια αυτή και θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και τι 17 ε, επιτροπές για την γνωμοδότησή του που ήταν όλε πολύτιμε. Ε, Ελπίζω να υπάρξει μια τελευταία συμφωνία πριν τον Νοέμβριο φέτος. Προσωπικά εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι ο παρομοιώδης ε, ε, ε, βρετανικός ρεαλισμός θα επικρατήσει και θα βρεθεί μια λύση προς όφελος και των Βρετανών και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, τα, ο έλεγχος σύνορα σε ό,τι αφορά τα αγαθά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βασίλειο που ανακοινώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή για να έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν οι επιχειρήσει, δείχνει ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο momentum λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα ακούμε στο όνομα της Επιτροπής ε, ε υπολογισμού, Προϋπολογισμού τον κύριο Στεφανούτζα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύρια Πρόεδρε. Μισή φρατζόλα φαινόταν να είναι καλή αρκετοί ε, παρά να, έχουμε, παρά να έχουμε ολόκληρο το ψωμί. Εσύ, παλιότερα ίσχυε το αντίθετο. Εσείς είπατε περισσότερη όθηση, πως θέλετε, περισσότερη ε, ορμή. Ε, αυτό είναι μια απλή μεταφορά για το έλλειψη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου στου τελευταίου τέσσερου γύρου, την έλλειψη διαφάνεια και έλλειψη δέσμευση για τι πολιτικέ ε, δηλώσει που υπέγραψαν. Ο Πρωθυπουργέ Τζόνσον, ε, όποιο καβαλάει την τίγρη, φοβάται να, να ξεκαβαλικέψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τα συμφέροντα των πολιτών τη. Η συμμετοχή τη Βρετανία δεν μπορεί να είναι μπουφέ, να διαλέγεται και να παίρνετε δηλαδή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε με τέτοια προσέγγιση γιατί τέτοιες αποφάσεις έχουν συνέπειες αλλά κανείς δεν θα αφαιρέσει από το ρόλο ε, του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την ενοποίηση αυτής της φυπήρου. Όλοι ξέρουμε πως το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι φτωχότερο χωρίς τους Βρετανούς του συνάδελφους ε, και πριν από τέσσερα χρόνια σφαγιάστηκε η Τζο Κόξ που μας έλεγε τότε ότι αυτά μας ενώνουν είναι περισσότερο από αυτά μας διχάζουν. Ευχαριστώ. Και τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής ε, ε, ΕΚΟΝ ο κύριος Σίλβα Περέιρα για ένα λεπτό, ένα λεπτό Πέτρο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από πολλούς μήνες οι διαπραγματεύσει ανάμεσα στον Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να παραμένουν στάσιμε στα πιο λεπτά ζητήματα και αναδείται και πάλι το σενάριο έλλειψης συμφωνίας. Αυτές με αυτές τις προϋποθέσεις δεν είναι αποδεκτό ούτε υπεύθυνο το Ηνωμένο Βασίλειο να αρνείται οποιαδήποτε ε, παράταση της περίοδου του διαπραγματεύσεων και ενώ ταυτόχρονα κρατά αδιάλακτη θέση ε, και επιμένει να μην, επιμένει να μην τηρεί τις ε, υποσχέσεις τις οποίες έδωσε ε, στη Συμφωνία Εξόδου όσον αφορά την θέσπιση συνολικών ελέγχων στη Βόρεια Ιρλανδία. Άρα λοιπόν, εφόσον πραγματικά δεν θέλει ε, μάλλον αν ο Μπόρις θέλει πραγματικά μια ε, συμφωνία θα πρέπει να αλλάξει την πραγματευτική του στάση. Ο Μισελ Μπαρνιέ έχει κάνει το αδύνατο δυνατό για να πετύχει καλή συμφωνία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κακή συμφωνία που θα βλάψει την νέα αγορά και θα μειώσει τα δικά μας περιβαλλοντικά, κοινωνικά κλπ. πρότυπα. Είναι πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής Ιστορικού Εμπορίου, ο κ. Πίτερς, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, ο χρόνος ε, τρέχει και τα θέματα επίγουν όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το τι βούληση υπάρχει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι ευρωπαϊκοί πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν μια συμφωνία ε, πόσο μάλλον τώρα με ε, τον οικονομικό τυφώνα που έζησε η Ευρώπη με την κρίση του κορονοϊού. 42.000 θέσεις εργασίες διακυβεύονται ε, στη δική μου χώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,2 ε, εκατομμύρια θέσεις ε, διακυβεύονται με το Brexit. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να διευκολύνουμε την επίτευξη συμφωνίας. Θέλουμε μια νέα εταιρική σχέση. Η συμφωνία αποχώρησης είπαμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό τη, ε, να υπάρχει ασφάλεια για τις ε, μικρέ επιχειρήσεις. Ε, μια νέα συμφωνία εταιρική σχέσης θα πρέπει να φροντίσει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες τη εσωτερική αγορά και θα πρέπει να είναι βιώσιμη. Λίγους μήνες έχουμε μπροστά μα συνάδελφοι. Ελπίζω όμως η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορέσει να συναυθεί. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντάνιελσον από την Επιτροπή Μεταφορών. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Μισελ Μπαρνιέ ε, για όλη τη του δουλειά που είναι παρόν σήμερα. Ε, Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με βάση ε, την εντολή, τη διαπραγματευτική εντολή που συμφωνήσαμε νωρίτερα. Εγώ ήμουν αρμόδιο για το θέμα αυτό ε, στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν και στο μέλλον ε, καλέ και ομαλές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. 45, πάνω από 45 εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Ταυτόχρονα το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να διατηρήσει τα ίδια δικαιώματα χωρίς να διατηρήσει τις ίδιες υποχωρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συμφωνία που να διασφαλίζει τις ε, καλές συνδέσεις, ε, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε και ε, τις συνθήκες εργασίες, τα περιβαλλοντικά πρότυπα κλπ, ώστε να μην είναι χειρότερα από αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αρημό για ένα λεπτό από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπαρνιέ, αγαπητοί Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μην αυταπατώμεθα. Ε, το Brexit είναι τεράστιο ιστορικό λάθος. Μόνο χαμένοι θα βγουν από αυτή την υπόθεση. Ε, ο διχασμός μόνο σε απώλειες οδηγεί και η συνεργασία ε, πέρα από τα σύνορα οδηγεί στην πρόοδο, κάτι που έχουν δείξει τα τελευταία 50 χρόνια. αλλά θα ήθελα ε, να δω να προστατεύονται οι μικρομεσαίες μας ε, επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι τους ε, δεν φταίνε για την παρούσα κατάσταση και δεν έχουν την ίδια ευελιξία που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν πόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περίπτωση ενός σκληρού Brexit, κάτι που απευχόμαστε φυσικά. Ε, προτείναμε να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης για όλα αυτά. Ε, θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περίπτωση σκληρού Brexit. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Κύριε Πρόεδρε, το ψήσιμο που μας προτείνεται εδώ περιλαμβάνει το κείμενο που το σύνολο των κοινοβουλευτικών ομάδων υποστήριξαν στην Επιτροπή Αλίας για να επαναλάβουμε αυτή τη βασική αρχή που αναφέρει ο κ. Μπαρνιέ στη διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν θα περιλαμβάνει μια συμφωνία μακροπρόθεσμη, ισορροπημένη, βιώσιμη για το θέμα της αλίας που να επιτρέπει δηλαδή αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα ε, και στους υδάτινους και στους ε, πόρους και για τις δύο πλευρές είναι πολύ σημαντικό ε, οικονομικό ζήτημα δεκάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης ε, επηρεάζονται και μία έξοδο χωρίς συμφωνία θα ήταν ε, καταστροφική για αυτούς Και είναι και οικολογικό το ζήτημα, διότι η κοινή πολιτική αλληλεία μας έχει επιτρέψει εδώ και χρόνια να εφαρμόσουμε μαζί με του Βρετανού μία αλληλεία που σέβεται τη βιοπικιλότητα. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε αυτού του κοινού κανόνε σε αυτό το πνεύμα λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και θέλω να ευχαριστήσω όλη την διαπραγματευτική ομάδα, όλους τους βουλευτές που, που ε, ενέταξαν αυτή τη θέση στο κείμενο. Ευχαριστώ για τη Λίμπε. Ο κύριος Βίντσε έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ενωμένο Βασίλειο ε, θα πρέπει να γίνει ένα σημαντικός σύμμαχος της Ένωσης ε, αυτή είναι η φιλοδοξία μα. Ξέρουμε αν θα είναι η πραγματικότητα. Συμφωνούμε από αυτού. Είναι δίπλα το βασίλειο. Έχουμε κοινέ αξίε, έχουμε κοινέ προκλήσει, κινητικότητα, δικαιοσύνη, ασφάλεια, συνεργασία στον τομέα τη εσωτερική ε, των εσωτερικών υποθέσεων. Η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών είναι σημαντική για μας. Το ίδιο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το μήνυμα λοιπόν του Κοινοβουλίου είναι σαφέ. Δεν μπορούμε ε, να ε, κάνουμε παραχωρήσει ό,τι αφορά τις η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν διαπραγματεύονται. Η καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του κυβερνού εγκλήματο, του διασυνοριακού εγκλήματο, είναι μία, ένα από τα success stories των σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Να μην ξεχνούμε όμω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο με δική του απόφαση θα, ξεκινήσει, θα συνεχίσει αυτή τη συνεργασία ως τρίτη χώρα. Ελπίζουμε από την άλλη πλευρά της μάχης να επικρατήσει ο ρεαλισμός και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια στενή σχέση υπέρ των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Η Ντανούτα Χούμπνερ έχει το λόγο τώρα με την ε, Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε, αγαπητέ Μισελ, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Να πω ότι του τελευταίου τρει μήνε νομίζω πω απογοητευτήκαμε όπω και εσεί από το επίπεδο των διαπραγματεύσεων και από την συνεχιζόμενη και τελική άρνηση για παράταση τη μεταβατική περίοδου ώστε να αποφευθεί τον Ιάριο ο κίνδυνο άταχτου Brexit. Ε, σεβόμαστε αυτή την επιτυχία. Η ιδιωτικοποίηση των διαπραγματεύσεων είναι καλά νέα. Υπάρχει κάπως περισσότερος χώρος και ελπίζω και να υπάρχει και, πιστεύω να υπάρχει πολιτικός χώρος για να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Θα τονίσω όμως ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η ποιότητα της μελλοντική μας σχέσης. Τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς δεν μπορούν να σταθούν ακόμα και με τις πιο ε, γενναιόδορες ε, συμφωνίες. Να τελειώσω λέγοντας ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να είναι το παγκόσμιο διεθνές οικονομικό κέντρο, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να συνεργαστεί με τις αυξανόμενες, με τις ε, ε αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για για την Επιτροπή Ανάπτυξης Φάλτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζουμε πως αυτή η συμφωνία θα μπορέσει να καλύψει κάποια από τα προβλήματα και να παρέχει λύσεις. Περιμένουμε κάποιες λύσεις και από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναζητούμε συμβιβαστικέ λύσεις στα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχουμε εγγυηθεί τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προσπαθούμε λοιπόν να στηρίξουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όλοι και το Συμβούλιο και το Κομισιόν και το Κοινοβούλιο αυτό είναι ήδη μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, πριν από 4,5 μήνε το Μένο Βασίλειο αποφάσισε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευθύ εξ αρχή, εμεί στην ομάδα συντονισμού παρακολουθήσαμε τι συζητήσει στενά για μια νέα εταιρική σχέση έτσι ώστε να υπάρξει μια ευρεία πολιτική συνένεση. Είμαστε σε στενή επαφή με τον επικεφαλή στην πραγμάτευση, τον κύριο Μπαρνιέ, τον οποίο πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Θέλω επίση να ευχαριστήσω τον Μάρο Σεύκοβιτ και θα, θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε κανένα μισάωρο στην επόμενη συνεδρίαση συντονισμού. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει τις νομοδοτήσεις 17 επιτροπών. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο θέλουμε ένα σαφέ ηχηρό μήνυμα ενότητα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τον, την εισηγήτρια, του εισηγητέ γενικά, την κυρία Πύρη, τον κύριο Χάντσαν, αλλά και του προέδρου και εισηγητέ όλων των γνωμοδοτήσεων των επιτροπών που γνωμοδότησαν. Αποφασίσαμε ότι χρειάζεται ένα νέο momentum για αυτήν τη διαπραγμάτευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να εντατικοποιήσει τη συζήτηση, να φτάσουμε σε μια επικοδομητική ε, λύση σύντομα. Νομίζω πω είναι προ συμφέρον και των δύο πλευρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος Γαρσία Πέρες, για μισή λεπτά. Νομίζω ότι ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπανέ για την προσπάθεια που έχει κάνει, να τον συγχαρώ για το έργο του και τον υποστηρίζουμε τι διαπραγματεύσει αυτέ. Ε, γνωρίζουμε ότι είναι σε μια κρίσιμη στιγμή. Όμω θέλω να αναφερθώ επίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κυρίε και κύριοι. Ο χρόνο πιέζει. Στον δρόμο ο κόσμο ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει και το Κοινοβούλιο. Ελπίζω οι λίγε κυβερνήσει οι οποίε διστάζουν στο Συμβούλιο να το καταλαβαίνουν αυτό και να φτάσουν σε μια συμφωνία τον Ιούλιο. Δεν μπορούμε να φύγουμε διακοπέ χωρί να ε, ενεργοποιήσουμε το σχέδιο ε, ανάκτηση για να μπορέσουμε ήδη να το εφαρμόζουμε από τον Ιανουάριο τα 750 δις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα μίνιμουμ, όπως και τα 500 δις των επιδοτήσεων. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί μας λένε ότι δεν είναι η στιγμή να διστάσουμε να κάνουμε προσπάθεια οικονομική. Πρέπει να επενδύσουμε για να επανεργοποιήσουμε την οικονομία. Ω τώρα οι φιλελεύθεροι εξωτερικοί που το 2008 μιλούσαν για λιτότητα, ακόμα και αυτοί αναγνωρίζουν ότι ήταν λάθο κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό να, να αναγνωρίζει κανεί τα λάθη του. Όμω τώρα όλοι πρέπει όλοι να κινηθούν προ την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την όθηση για να αλλάξουν οι οικονομίε μα, να τι προσαρμόσουμε στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, στα περιβαλλοντικά ζητήματα, να εγγυηθούμε μια πιο δίκαιη κοινωνία με πιο ισχυρές δημόσιες πολιτικές, οικολογική μετάβαση, ψηφιοποίηση για να αλλάξει η οικονομία μας και η κοινωνία μας. Θα πρέπει και το Συμβούλιο να έχει το ίδιο όραμα καθώς και την ίδια, το ίδιο θάρρος. Όταν δεν υπάρχει όραμα τότε ο λαό υποφέρει. Εμείς έχουμε όραμα ως Κοινοβούλιο και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε δεν θα το επιτρέψουν οι συμπολίτε μα. Δεν θα δεχτούμε λοιπόν μια κακή συμφωνία στο Συμβούλιο. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιμείνουμε λοιπόν στην, στο ρόλο που παίζει το Κοινοβούλιο στι αποφάσει αυτέ. Μιλάμε για θεμελιώδη ζητήματα εδώ, όπω ε, το πώ ε, θα ε, διαχειριστούμε αυτό το, το, το μέσο ανάκτηση, το, το NEST, το Next Generation. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη δημοκρατία και μεγαλύτερη λογοδοσία και η μόνη προϋπόθεση που θα πρέπει να επιβάλλουμε σε αυτό το σχέδιο ανάκτησης είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Κυρίε και κύριοι, είναι η στιγμή να συνδυάσουμε τους στόχους μας, τις αρχές μας με την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε αγαθοί σε έναν κόσμο όλο και πιο περίπλοκο όπου πρώην εταίροι φαίνεται να έχουν χάσει ε, την πίστη στην, στην πολυμερή προσέγγιση και τη συνεργασία. Πρέπει να είμαστε λοιπόν στεναροί, αλλά να έχουμε αρχέ και όραμα. Θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη που να μπορεί να δείξει το δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Σόλτ. Τζάνι, πρέγω, μινούτο. Πρόεδρος Τζάνι, λεπτό. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για πρώτη φορά νομίζω πως ε, αυτή την εβδομάδα θα γίνει ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, για το οποίο γνωρίζουμε ε, ήδη την έκβαση, δεν θα υπάρξει συμφωνία για το σχέδιο ανάκαμψη και θα υπάρξει και μάλιστα σύγκρουση ανάμεσα στα κράτη-μέλη που ήδη είδαμε πήραμε μια γεύση αυτές τις μέρες. Και αυτό αποδεικνύει ακόμα άλλη μια φορά ότι είναι ανεπαρκής ενυπαρκεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά ε, ε, ε, όργανα όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. Πρόταση της Κομισιόν που ήδη ήταν πολύ ανεπαρκής. Μιλάμε για 400 δις ευρώ για καθαρών επιδοτήσεων και 3 τέταρτα αυτών των χρημάτων θα φτάσουν μόνο το 2023, δηλαδή τρία χρόνια μετά από την κρίση, μετά από το ξέσπασμα της πανδημίας, όταν ήδη δηλαδή οι εταιρείε εργαζόμενοι θα έχουν χάσει τη θέση τους. Δείχνει ακόμα μια φορά πως η διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της Ένωσης δεν είναι προσαρμοσμένη για να δίνει απαντήσεις ε, στους πολίτες και στις εταιρείες. Και αυτά τα χρήματα Ακόμα μια φορά θα δοθούν ε, σε με αντάλλαγμα νέους φόρους που θα επιβαρύνουν τις εταιρείες, περίπου 70.000 εταιρείες εντός της Ένωσης, δηλαδή όχι μόνο τις πολυεθνικές και θα βαρύνουν βέβαια και τους καταναλωτές, γιατί φυσικά οι εταιρείε θα τα μετακυλήσουν στους καταναλωτές. Και αφήστε με να τελειώσω ε, με Το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο για να μετατραπούν οι με βιομηχανίες ορισμένων χωρών με τα χρήματα κάποιων άλλων χωρών. Τράπεζα της Γαλλίας και της Γερμανίας και αυτό συνέβη αυτό μάλλον και τώρα ε, αυτό μπορεί να συμβεί εις βάρος ε, κάποιων ε, βιομηχανιών κάποιων χωρών. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ας είμαστε ειλικρινείς. Κανεί δεν περιμένει να συμβεί κάτι πραγματικά στο Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο όσον αφορά το σχέδιο ανάκαμψη Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν ε, παζαρέματα ε, και τελικά όλοι θα ε, επιστρέψουν στις πατρίδε του και θα πούνε πόσο καλά υπερασπίστηκαν τα εθνικά συμφέροντα. Ακόμα και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εγκατέλειψε κάθε ελπίδα αποτελέσματο πριν καν ξεκινήσει. Και αυτό είναι απογοητευτικό όταν συνέρχονται οι ηγέτες μα να μην περιμένει κανεί πολλά. Δεν θα ήταν ωραία ε, αν έστω και μία φορά ε, καταφέρναμε να υπερπληρώσουμε τις προσδοκίες των πολιτών μας. Ε, Έχουμε μία κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν τελείως απρόβλεπτη και όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα για να μετριάσουμε ε, τον οικονομικό αντίκτυπο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει πόρου γι' αυτό και θα πρέπει να διοχετευτούν στην οικονομία που θέλουμε αύριο, όχι αυτήν ε, που βάζει το κέρδο πάνω από τον πλανήτη και του ανθρώπου προσπάθειες αλλά και τα ωφέλη ε, θα είναι καλά διότι ε, αντιμετωπίζουμε την απώλεια βιοπικιλότητας, ε, την κλιματική κρίση, την ψηφιοποίηση. Φανταστείτε μία φορά οι κυβερνήσεις να μην επιδιώξουν δραματικές σκηνές ε, αλλά να επιλέξουν τολμηρές λύσεις ε, και αυτό άλλωστε είναι εθνικό συμφέρον κάθε κράτους μέλους το να υπάρχει μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες της και για την οικονομία. Ε, δεν είναι παιχνίδι μηδενικού υπολείπου, μηδενικού αθροίσματος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας εργαστούμε λοιπόν όλοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ πολύ. Ένα μισή λεπτό, κύριο Έπινγκ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο αγώνα για το σχέδιο ανάκαμψη. μοιάζει με παρτίδα πόκερ και ε, μοιάζει πιο πολύ με ε, παιχνίδι δωροδοκιών ε, και εκβιασμού. Ε, εκβιασμός εις βάρος των βορειοευρωπαϊκών χωρών ε, και δεν ε, έχει να κάνει αυτό το θέμα με τον ε, κορονοϊό. Φαίνεται ότι το, ο στόχο του σχεδίου ανάκαμψη είναι ο μεγαλύτερο προπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλύτερη φορολογία δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε πώ θα, πώς θα πάνε τα πράγματα. Νομίζω ότι οι Βρετανοί θα είναι πολύ ικανοποιημένοι που δεν συμμετέχουν σε όλα αυτά. Εμένα με εκπλήσει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το Brexit. Ε, εμένα μου φαίνεται ότι απλά είναι επανάληψη κάποιων απαιτήσεων απέναντι σε μια χώρα που τα τελευταία 100 χρόνια ηγείτο ε, ε, στην Ευρώπη. Δεν θα βρισκόμασταν εδώ χωρίς τους Βρετανούς. Ε, στο ψήφισμα αυτό ε, εγώ βλέπω χερεκακία και διάθεση εκδίκησης, αλλά πρόκειτο για δημοκρατική απόφαση. Ε, Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά όμως ε, είναι απλά ένας μικρός παίχτης ανάμεσα στους πραγματικά μεγάλους ε, οι Βρετανοί. Ε, θα υποστούν ψυχρολουσία τώρα αντί για ευγενή χαιρετισμό. Ε, φοβάμαι ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε πολιτική χωρίς σε πρόπτικες για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά. Ε, ο κύριος ε, Σίρδεβαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στο μεταξύ έχω την εντύπωση ότι ε, είναι μεγαλύτερες οι αντιφάσεις ε, παρά οι συμφωνίες ε, εδώ και ότι το καλό αποτέλεσμα όλο και απομακρύνεται πιο πολύ και δεν θέλω να επικρίνω τις εργασίες του Μισελ Μπαρνιέ τον οποίο εκτιμώ αλλά είναι πολύ κακή η θέση λόγω της βρετανικής θέσης και θέλω να το τονίσω αυτό. Στο τέλος της χρονιάς λοιπόν ή θα έχουμε κακό αποτέλεσμα ή σκληρό Brexit. Και στο όνομα της αριστεράς ε, θα ήθελα να πω ότι το κοινωνικό dumping, το περιβαλλοντικό dumping, το φορολογικό dumping, ε, το να μην έχουμε ασφαλή δεδομένα ε, είναι απαράδεκτα θέματα. Δεν θα αποτελούσε λύση για μας μια τέτοια συμφωνία. Και Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης ώστε να στηρίξουμε, να προστατεύσουμε τις περιφέρειες που θα πληγούν ιδιαίτερα από το Brexit. στο Συμβούλιο θέλω να πω ότι οι άνθρωποι περιμένουν ακόμα ένα μήνυμα αλληλεγγύης και συσπήρωσης. Ε, το Next Generation EU ε, είναι ένα σύμφωνο ε, ανάμεσα στις γενιές και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε απλά επιπλέον περικοπές ε, στη μελλοντική ε, κοινωνική προστασία. Πρέπει να κλείσουν ε, τα φορολογικά παραθυράκια και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει ε, τις εθνικές οικονομίες ε, και ε, οι κερδοσκόποι και οι μεγάλες εταιρείε θα πρέπει να καταβάλουν τους φόρους τους, θα πρέπει να έχουμε και ψηφιακό φόρο. Αυτή είναι η αλληλεγγύη που περιμένει η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα πάμε λίγο πίσω. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσόλο, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ενώ η υγειονομική κρίση φαίνεται σιγά σιγά να σταθεροποιείται, οι οικονομικέ προκλήσει είναι τεράστιε μπροστά μα, Για μένα δύο δυνατότητε υπάρχουν σήμερα για μα, Είτε θα διαπραγματευτούμε με βάση εθνικέ μα θέσει την έξοδο από την κρίση, ο καθένα να υπερασπίσει τα συμφέροντά του δηλαδή, είτε δεχόμαστε ότι η μόνη λύση είναι να οικοδομήσουμε κάτι μαζί. Αυτό είναι, αυτή είναι και η λογική του σχέδιου ανάκαμψης και του πολιτού δημοσιονομικού σχεδίου. Δεν θέλουμε εδώ απλάς, απλά να ε, μοιράσουμε χρήματα παντού. Θα πρέπει να είναι εστιασμένη ε, αυτή η ενίσχυση και θα πρέπει η αλληλεγγύη αυτή που θα δείξουμε να οδηγήσει σε πραγματική ανάκαμψη. Εγώ ε, είμαι ανήσυχος. Θα, θα, θα δανειστούμε 750 δισεκατομμύρια στις χρηματαχωρές χωρίς να ξέρουμε πώς θα τα επιστρέψουμε. Διότι όταν μιλάμε για μια εθνική συνεισφορά, μια μείωση των χρημάτων για τις επόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές, αυτό πραγματικά διακυβεύει το σύνολο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Για μας μόνο η θέσπιση μιας πραγματικών ιδιών πόρων θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε την αξιοπιστία αυτού του σχεδίου ανάκαμψη αλλά να και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η πρόταση για το πολιτές πλαίσιο είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξη από ό,τι περιμέναμε. Η, η ύπαρξη και μόνο ενός σχεδίου ανάκαμψη δεν αρκεί διότι ακόμα και αν μιλάμε για ένα πακέτο ε, είναι διαφορετική η στόχη. Το σχέδιο ανάκαμψη θα μα επιτρέψει να ξαναπάρουμε μπροστά. Ο νέο όμω προπολογισμό ευρωπαϊκό θα ορίσει τη δυνατότητα που θα έχουμε να φτάσουμε ω το τέρμα. Μόνο μια φιλόδοξη, ένα φιλόδοξο προπολογισμό μπορεί να δώσει διαθροτικέ απαντήσει στι πολλέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε και θα μα δώσει τη δυνατότητα να είμαστε ανεξάρτητοι και οικονομικά και στρατηγικά θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε μεγάλα ευρωπαϊκά σχέδια όπως ε, αυτό με τις μπαταρίε μπαταρίες ή το υδρογόνο κτλ. Ε, κάποια προγράμματα που χρηματοδοτούν τόσο σημαντικά ζητήματα στον τομέα της έρευνας, στον τομέα του ψηφιακού, στον τομέα της άμυνας, της νέας αγοράς, υποχρηματοδοτούνται. Το ίδιο ισχύει και για κοινωνικά σχέδια ή σχέδια που έχουν να κάνουν με τους νέους. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντα, θα ήθελα να θυμίσω ότι η δική μου πολιτική ομάδα δεν θα υποστηρίξει έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό εάν αυτό εξακολουθεί να χρηματοδοτεί ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που καθημερινά γυρίζουν τις πλάτες τους στις αξίες μας και ε, δεν σέβονται το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Πρέπει να σταματήσει αυτό και να σταματήσει τώρα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπέγκεν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, το Ταμείο Ανάκαμψη είναι ένα μέσο που άνευ προηγουμένου με πάνω από 700 δις ευρώ είναι η ίδια η έκορες μια νέα εποχή αλληλεγγύης στην Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την όθηση του Ιταλικής Κυβέρνησης στη Συμβολή των Άλλων Κρατών Ισπανίας, Γαλλίας και Γερμανίας. Τα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, εάν θα έχουν το θάρρος να το εκρίνουν, θα γράψουν την ιστορία της Ένωσης. Ξέρουμε ότι ορισμένε ε, κυβερνήσει διστάζουν, αλλά οποιαδήποτε συμβασμό προ τα κάτω είναι απαράδεκτο. Γιατί ε, αφαιρεί και τρώει ε, πολύτιμο χρόνο. Όπω είπα σήμερα μπροστά στι κάμερε ο Πρωθυπουργό μα Κόντε, η Ιταλία είναι προέτοιμη και ευχόμαστε και η Ευρώπη να είναι και να εγκριθεί το Next Generation EU όσο γίνεται πιο σύντομα. Οι πολίτε και οι ευρωπαϊκέ εταιρείε το αξίζουν αυτό, να διατεθούν τα χρήματα αμέσω το οφείλουμε σε όλους όσοι καθημερινά σημαίνουν τη διαφορά. Συνάδελφοι, η αλληλεγγύη έχει ρέει μάλλον στις φλέβες της Ευρώπης ξανά και τώρα ελπίζουμε και φροντίζουμε να φτάσει και στην καρδιά της. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ΕΛΚ ήταν στην πρώτη γραμμή στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν για ένα σχέδιο ανάκτηση με τι μεγαλύτερε ενισχύσει για την καταπολέμηση του COVID. Και το κάναμε αυτό ενωμένοι με λεγγύη και με ευθύνη, με έθιμη ευθύνη. Τώρα το Συμβούλιο πρέπει να σταθεί στο των περιστάσεων. Ο χρόνο πιέζει. Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι αυτοί οι οποίοι έκλεισαν τα μαγαζιά του να μπορέσουν να τα ξανανοίξουν. Γι' αυτό θα πρέπει οι κυβερνήσει των κρατών μελών να δράσουν γρήγορα και υπεύθυνα η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να συνοδεύεται από εθνικές μεταρρυθμίσεις, φιλόδοξες, έτσι ώστε η οικονομία μας να είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονη, πιο ανταγωνιστική, πιο βιώσιμη, τα, τα συστήματα υγείας να είναι πιο ανθεκτικά και να προστατεύσουμε όλες τις οικογένειες, να υπερασπιστούμε τους Ισπανούς, ε, και, πατρι, και να είμαστε πατριώτε σημαίνει ψηφιοποίηση, σημαίνει κοινή γεωρική πολιτική έτσι ώστε να υπάρχουν ευκαιρίες στην Ήπεθρο, να, να δώσουμε νέα ενέργεια στην, στον τουρισμό, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης που είναι η καλύτερη ε, κοινωνική πολιτική. Αυτή είναι η πραγματική Ευρώπη, αυτή που περασπίζεται το ΕΛΚ, η Ισπανία που θέλουμε. Thank you for minutes, Madam Για δύο λεπτά η κυρία Μποναφέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιτέλου, οι επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων θα πρέπει να εκφραστούν όσον αφορά το σχέδιο ανάκαμψη που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Θέλουμε να φτάσουμε σε συμφωνία γρήγορα, αλλά όχι οποιαδήποτε απόφαση. Απόφαση που να είναι στο ύψο τη κρίση που διανύουμε. Όπω ξέρετε, η πολιτική μα ομάδα εξ αρχή θετικά δέχτηκε το Next Generation EU. Για μα το σχέδιο τη Επιτροπή είναι το μήνυμο, δηλαδή ένα καλό σημείο εκκίνηση με στοιχεία που χρειάζεται να προσεχθούν και αναφέρω τα εξής δύο. 750 δις που θα χρησιμοποιηθούν για να ξανασταθούν στα πόδια τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι και να δοθεί προοπτική στους ανθρώπους που έχουν χάσει την δουλειά τους. Δύο, κοινό, η δυνατότητα κοινού ευρωπαϊκού δανείου που εγγυάται ε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ίδιους πόρους της ε, ε, δυνατότητα να πληρώσουν το κόστος της κρίσης αυτοί που δεν πλήρωσαν φόρους όταν έπρεπε ή όπως ας πούμε οι πολυεθνικές. Για να καταπολεμηθεί το περιβαλλοντικό dumping, οι πολίτες χρειάζονται βοήθεια σε κάθε μήκος και πλάτος Ευρώπης. Αυτή η κατάσταση χτύπησε παντός στην Ευρώπη. Ευρώπη με διαφορετικό τρόπο. Όμως ε, αυτά τα, τα, τα ε, λιτά κράτη ε, δεν πιστεύουν πως, δεν το πιστεύουν αυτό, δεν το σκέφτονται αυτό, ότι πρέπει να σωθούμε όλοι μαζί. Οι αλυσίδες παραγωγής είναι αλληλένδετες, οι οικονομίες μας επίσης και αν καταρρεύσει κάποιος θα καταρρεύσουμε όλοι. Και το ίδιο ισχύει και για τις χώρες που αισθάνονται λιγότερο ευάλωτες. Δεν είναι μόνο αλληλεγγύη, είναι ε, κοινό συμφέρον. Πρέπει να σκεφτούμε το δρόμο που έχουμε μπροστά μας για να υπάρξει ανάκαμψη ε, και θέλω να ανανεώσω την έκκληση προς το Συμβουλίο να μην αποδυναμώσει ούτε να καθυστερήσει το σχέδιο ανάκαμψης. Ε, με τους κατάλληλους πόρους και γρήγορα μπορούμε να αντιστρέψουμε την τάση και το Κοινοβούλιο μας είναι έτοιμο. Ευχαριστώ. Τέσσερις μήνες, που έχουμε στη διάθεσή μα να φτάσουμε σε μια εταιρική σχέση μεταξύ εξωμένο Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο χρόνο. Γίνεται όμω. Είμαι βέβαιη ότι όπω οι ευρωπαϊκοί λαοί που εκπροσωπούμε εδώ, έτσι και ο Βρετανικό λαό θέλει να διατηρήσουμε ισχυρού δεσμού με αμοιβαία ωφέλη και αύριο και σήμερα να μπορέσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, η υγεία, η διατροφική ασφάλεια όλων, να την χάνει προσοχής ο πλανήτης να προστατεύεται. Και είμαι βέβαιο ότι και ο Βρετανικό λαό θέλει να προστατεύονται τα προσωπικά του δικαιώματα και γνωρίζω πολύ καλά τα, τα προσωπικά του δεδομένα. Ε, και βεβαίω οι Βρετανικέ επιχειρήσει, όπω και οι ευρωπαϊκέ, θέλουν να συνεχίσουν τη βιομηχανική του συνεργασία και τι ανταλλαγέ του με του Ευρωπαίου. Είναι προ όφελο όλων αυτό. Αυτό που θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο είναι ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Το μήνυμα ότι περασπιζόμαστε τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων που μας ψήφισαν και που βασίζονται σε εμά. Οι γεωργοί μας, οι αλληλείς μας, οι επιχειρήσεις μας. Είναι ένα μήνυμα για το τι θεωρούμε εμείς ως δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία που θα πρέπει συνέχεια να επικυρώσουμε. Διότι από αυτή την πλευρά ε, της μάχης το δικό μας κοινοβούλιο θα έχει το τελευταίο λόγο. Κανείς δεν θέλει να προσθέσει τις αρνητικές επιπτώσεις Τη ύπαρξη συμφωνίας σε, αρνητικέ αρνητικές του COVID. Κανεί δεν είναι υπεύθυνο για την πανδημία αυτή βέβαια, αλλά έχουμε μια κοινή ευθύνη να αποφύγουμε να προσθέσουμε και άλλη κρίση στην κρίση. Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε όμω και ένα δρόμο μπροστά μας. Αυτό της πολιτική δήλωση ε, μεταξύ Ευρωπαίων και Βρετανών διαπραγματευτούν από κοινού, που υπέγραψαν από κοινού έτσι ώστε να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο, αύριο 18 Ιουνίου. Είναι η μέρα της έκκλησης, της ομιλίας του στρατηγού Ντεγκόλ από το Λονδίνο, όταν ήμασταν και τότε ενωμένοι για να πολεμήσουμε από κοινού. Ζητώ από Βρετανούς λοιπόν φίλους να είμαστε στο ύψος αυτής της κοινή ε, ιστορίας. Ας είμαστε φιλόδοξοι από κοινού, διότι αυτό είναι που κάνει το μεγαλείο μας. Για ένα λεπτό, κυρία Χωτοσάρη. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόλις εξοικονόμησαν 80 εκατομμύρια ευρώ, διότι ε, καθυστέρησαν ε, όσον αφορά τον κοροναϊό. Ε, σύντομα, κανένας ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ε, τολμάει να μιλήσει ε, ε, κατά του Brexit. Πρόκειται για άλλο ένα βήμα με κατεύθυνση μια μια κεντρική ένωση και αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με το άρθρο 205. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει και νομοθεσία για νέους ίδιους πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγάλο μέρος των οικονομικών προβλημάτων θα μειωνόταν εάν ε, καταργούσαμε το ευρώ. Σύμφωνα με μια μελέτη, οι φιλανδικές εξαγωγές ε, θα ε, ήταν αυξημένες κατά 40% εάν είχαμε το δικό μας νόμισμα. Θέλω τα λεφτά μου πίσω. Ένα λεπτό η κυρία Χάουταλα. Πρόεδρε, Βρίσκω θλιβερό όταν βλέπω να κολλάνε οι διαπραγματεύσεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ε, κάθε προϋπόθεση για να πετύχουν ε, μια καλή εμπορική συμφωνία. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε τέτοια ευθυγράμμιση συμφερόντων η συμφωνία πάνω στη νέα σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίζει την κοινή μας ιστορία, την γεωγραφική ε, ε, ε, το ότι βρισκόμαστε γεωγραφικά κοντά και κάθε συμφωνία που παρέχει συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα είναι απαραίτητο. Δεν ε, επιτρέπεται να αποτύχουμε. Χρειαζόμαστε την ε, δεύτερη καλύτερη συμφωνία στον κόσμο. Ε, δηλαδή μια συμφωνία που να είναι τόσο καλή που το μόνο καλύτερο από αυτή να είναι η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή. Ευχαριστώ κύριε Σκουσμίκ. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, εξετάζοντας ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχέδιο ανάκαμψη, ε, αυτό αποτελεί πολύ καλή βάση για τι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο. Προφανώς πρέπει να διαπραγματευτούμε γρήγορα προ όφελο και των κοινωνιών μας και ε, των κρατών μελών, διότι ήδη στο ε, δεύτερο τρίμηνο του έτους ε, θα έχουμε κατά 30% μείωση του ΑΕΠ. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι οι αγρότες ε, έχουν διασφαλίσει ε, την τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν με ευέλικτο τρόπο τα μέσα που έχουμε για στήριξη ώστε να λύσουμε τα πραγματικά οικονομικά προβλήματα στις χώρες μας και να μην λύσουμε μόνο το θέμα του κλίματος και της ψηφιοποίησης. Βιλανουέβα Ρουίς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τελειώνει ο χρόνο. Πέντε μήνε. Ε, η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Υπάρχουν ευκαιρίε για ισορροπία ανάμεσα στα καθήκοντα και τι υποχρεώσει ε, και τα δικαιώματα. Ε, εγώ δεν θέλω να διαλυθούν συμφωνίε ενώπιον τη απειλή για μη συμφωνία. Είναι σημαντικό να το επιτύχουμε. Οι πολίτε μα το περιμένουν. Ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. αναμένουν σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Ε, το σχέδιο ανάκαμψης το οποίο κάνουμε μαζί θα πρέπει να είναι ένας τρόπος για να μετατραπτοποιήσουμε πει αυτό σε ένα project ώστε οι πολίτες να μπορούν να το στηρίξουν ε, και να το δεχτούν. Υπάρχουν ε, θετικά στοιχεία στις συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου ε, κατά το dumping, περιβαλλοντικά στάνταρ, δικαιώματα, αλλά βλέπουμε και κάποιες ανεπάρκειες. Δεν μπορούμε να προχωράμε αν δεν είμαστε ένας ανεξάρτητος και διεθνής φορέας. Δεν μπορούμε εμείς να υποτάξουμε την διεθνή πολιτική μα στην διεθνή πολιτική του Τζόνσον, δηλαδή του Τραμπ. Ε, ε, θα πρέπει να είμαστε πιο ανεξάρτητοι εμείς και έτσι θα έχουμε και λαμπρό μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό η κυρία Ρουκμάκερ. Α είμαστε ρεαλιστέ και λογικοί. Το Βρετανικό Έθνο είναι ένα αγαπητό και αξιοσέβαστο μέλος τη ευρωπαϊκής οικογένεια. και αυτό ε, θα είναι για πάντα και για τι επόμενες γενίε δεν είναι πλέον μέλος της Ένωσης, γι' αυτό πρέπει να φτάσουμε σε συμφωνία με τον κοντινό μας γείτονα και παλιό φίλο. Μετά από τέσσερις γύρους ανεπιτυχών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να καταλήξουμε στο ότι η στρατηγική δεν έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής. Οι περιστάσεις έχουν αλλάξει. Είμαστε μια τεράστια οικονομική κρίση, τη κρίση COVID-19. Δεν μπορούμε να ε, περιμένουμε, να, να, μάλλον να αντέξουμε no deal. Το διαζύγιο είναι οδυνηρό για όλα τα μπλεκόμενα μέρη. Υπάρχει τίμημα και για τα δύο και τις δύο πλευρές. Πρέπει να σκεφτούμε ότι όμως τις επόμενες γενιές εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα ηθικό ζήτημα, αλλά με μια κατάσταση που χρειάζεται λογική προσέγγιση. Οι καταστάσεις, οι περιστάσεις αλλάζουν, αλλά οι στρατηγικές θα πρέπει και αυτές να αλλάξουν. Να μην στοχεύουμε στην ίστατη συμφωνία, αλλά στην καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή. σκεφτούμε τις επόμενες γενναίες στη Βρετανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε λογικοί. Ευχαριστώ. σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έξι μήνες ε, ε, πριν από άλλη ε, μία αγωνιώδη φάση του Brexit και πάλι δεν έχει δημιουργηθεί πρόοδος και αυτό το να κάνουμε το Brexit πραγματικότητα έχει γίνει το να μην κάνουμε τίποτα πραγματικότητα και ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται να ξέχασε την πολιτική δήλωση που ο ίδιος συμφώνησε και υπέγραψε πέρυσι. Ξέχασε την κοινή δήλωση που αναφέρεται σε μια βάση για μια φιλόδοξη εταιρική σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα ίσο πεδίο ευκαιριών. Το Brexit είναι κάτι όπου, όλοι χάνουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τουλάχιστον όμως με μια οργανωμένη έξοδο συντεταγμένη μπορούμε κάπως να μετριάσουμε αυτές, αυτή τη ζημιά. Πρέπει και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να έχουν κάποια ασφάλεια για το μέλλον τους. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε πια χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να φανούμε δημιουργικοί. Ίσως ε, κύριε Μπαρνίε μπορείτε να καλέσετε τον Μάρκους Ράσφορντ στον επόμενο κύριο διαπραγματεύσεων. Τουλάχιστον αυτός ε, κάτι κάνει στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Στην συζήτηση για τη συμφωνία με, την, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ακούγεται συχνά ας ε, κάνουμε το ίδιο που κάναμε με την ΣΕΤΑ, τη συμφωνία με τον Καναδά. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι ε, η χαρακτηριστική ψευδής ιδέα ότι τα πράγματα ε, μοιάζουν μεταξύ τους. Ε, Είδαμε ότι η συμφωνία με τον Καναδά ήταν μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσμα προσπάθειας όπου είχαμε προσέγγιση των θέσεων. Ε, με ε, το Ηνωμένο Βασίλειο όμως είχαμε μια κοινή αγορά και τώρα θέλουμε ε, διαζύγιο. Εάν λοιπόν κινηθούμε προς την κατεύθυνση της συμφωνίας με τον Καναδά θα είναι μια κακή συμφωνία. Δεν θέλουμε κακή συμφωνία, θέλουμε καλή συμφωνία προς όφελος των πολιτών των θέσεων απασχόλησης. Δεν θέλουμε λοιπόν κακή συμφωνία. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία. Κακή συμφωνία σημαίνει απώλεια οικονομικής ανάπτυξης. Ε, ακόμα και οι Βρετανοί είπαν ότι θα έχουμε απώλεια 4,6% εάν έχουμε συμφωνία παρόμοια με αυτήν ε, με τον Καναδά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πήρε την απόφαση να φύγει μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πλέον πραγματικό. Το Τζόνσον το είπε ξανά, θέλει να βρει μια συμφωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η επιλογή των Βρετανών απέδειξε ότι όταν, όταν ο λαός θέλει, μπορεί. Είχε τη, την, τη δυνατότητα να μπορέσει να είναι συνεπή στι επιλογέ του παρά τι πιέσει και ο κύριο Τζόνσον, ο οποίο έλεγε ε, μπόρεσε να φέρει σε πέρα αυτό το έργο διαψεύδοντας τους μάντες κακών και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία έχει το πρόβλημα τώρα. Ε, ε, Βεβαίω και χρειάζεται μια ισότιμη συμφωνία. Από την άλλη, φορά, από την άλλη στιγμή, πλευρά, καταλαβαίνουμε τον κύριο Τζόνσον, ο οποίο έχει αντιμετωπίσει και αυτό προβλήματα με τη μετανάστευση, ε, όπου έχουμε αυτή την ιδεολογικό φήμοτρο με τα 35.000 ευρώ που θα δίνονται σε ξένους μόνο. Ε, βεβαίως δεν λύνονται όλα τα τα προβλήματα με ένα Brexit και η Γαλλία δεν είναι ένα βασίλειο, όμως η κατεύθυνση είναι σωστή. Μια χώρα που δεν είναι πλέον υπόδουλος, είναι φίλος της Ευρώπης, ε, επιλέγει τους φίλους της, ε, επιλέγει τη συνεργασία και όχι την ε, υποτέλεια και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Τεχνοκρατών τόσο περιφρονητικών και κρύων όπως ο Μισελ Μπαρνιέ. Ο κύριος Λαγκουντίνσκι έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. They Μας ρωτούν γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί είμαστε ενωμένοι και παιδί με τόσο χρόνο να πραγματευόμαστε για κάτι που η Βρετανική κυβέρνηση έχει αγνοήσει και έχει απορρίψει. Και η απάντηση είναι το κάνουμε για το δικό μας κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, όχι το χρόνο, ίσως σε, σε δύο χρόνια, ίσως αργότερα, αλλά αυτό το μέλλον θα έρθει. Το κάνουμε για τις κοινέ αξίες μας, τα κοινά συμφέροντά μας. Αξίες που δεν εξαρτώνται από την υπογραφή ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλιματική αλλαγή, γυναίκες, δικαιώματα μειονοτήτων, είναι πράγματα τα οποία μοιραζόμαστε αναξάρτητα από να είναι κάποιο μέλο τη Ένωση Το κάνουμε για του Ευρωπαίου και από τι δύο πλευρέ τη μάχη. Και για αυτού που έχουν οικογένειε, ε, βιογραφίε, θέσει απασχόληση, ιστορίε αγάπη. Το κάνουμε για εσά, του Βρετανού φίλου, πολίτε που πιστεύουν στη σοφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο από ότι πιστεύουν ε, στην σοφία του Τη κυβέρνησή του, διότι εάν αυτοί πέφτουν χαμηλά, εμείς έχουμε στόχο ψηλά και το ψήφισμα αυτό είναι φιλόδοξο. Δεν θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτε να είναι πολίτε μια τρίτη χώρα. Δεν βλέπουμε τον Βασίλειο τρίτη χώρα. Όπω είπε ένα διάσημο Βρετανό, ένα Brexit με συμφωνία είναι το καλύτερο, η καλύτερη συμφωνία για το μέλλον, αλλά καλύτερη από οποιαδήποτε, η χειρότερη συμφωνία για το μέλλον ήταν καλύτερη από οποιαδήποτε όλη. Εσεί τώρα ε, να αποφασίσετε τον μπαλάκι τη δική πλευρά, κυρία Τζόνσον. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ο κύριο Φιντέντσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινάνε διαπραγματεύσει πολύ δύσκολε για μια απάντηση κρηματοοικονομική ε, που όσο και είναι σημαντική μπορεί να μείνει πολύ χαμηλότερα από τι προσδοκίε και μάλιστα να καλύπτεται από αιρεσιμότητα και είναι αργά μάλιστα ψίχουλα το 2020 και άλλα λίγα ψίχουλα το 2021. Όταν θα έρθουν τα χρήματα, πολλές εταιρείες σε πολλούς τομείς, στη βιομηχανία, στον τουρισμό, στις μικρομεσαίες θα έχουν κλείσει και πολλοί κόσμος θα έχει μείνει χωρίς δουλειά. Αυξάνονται οι ανισορροπίες της εσωτερική αγοράς και δεν απαντάμε πραγματικά στην κρίση. Θα αποφασίσει κάποιος ε, να δραστηριοποιήσει το, το, το Ταμείο Ανάκαμψης εσείς προχωράτε με το Green Deal, επιβάλλετε νέους φόρους ε, στις εταιρείες και στους πολίτες νέο ε, στυλ ζωής. Ανακαλύψατε την λέξη αλληλεγγύη, αλλά ξεχάσατε τη λέξη ε, υπευθυνότητα. Σόλτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να επηρεάσουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και επικροτώ τα ξεκάθαρα λόγια που ακούσαμε για την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των πολιτών ε, και την κατάσταση της Ιρλανδίας. Θα ήθελα να πω, ευχαριστώντας ε, και τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ότι η ε, συνθήκες μη ίσου ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται να υπάρξουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εισηγητές για τη δουλειά τους. Ε, θα ήθελα λοιπόν ε, να θέσω το ερώτημα. Ε, γιατί με την οικονομική κρίση και την κρίση του κοροναϊού δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε νέα μορφή στις διαπραγματεύσεις. Οι προτάσεις για συνεργασία, η η μείωση των ε, εξοπλισμών ε, ελπίζω να οδηγήσουν σε καλύτερο αποτέλεσμα και γι' αυτό ελπίζω ότι θα υπερψηφίσετε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πονσάτιο Πιόλ. Σε ένα λεπτό. Ε, η Σκοτία ήθελε να παραμείνει στην Ένωση, αλλά ε, φημώθηκε στις διαπραγματεύσεις και τώρα έχει ε, αποχωρήσει μαζί με το υπόλοιπο του Ηνωμένου Βασιλείου. Είδαμε να αλλάζουν τα σύνορα της Ευρώπης καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ε, αλλά η συνεργασία είναι ο δρόμος προς τη σταθερότητα. Το μόνο πράγμα που δεν έχει δοκιμάσει ακόμα η Ευρώπη είναι το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας και στον κόσμο. Ένα καλύτερο είδους ελευθερίας με βάση τη δημοκρατία και τη συνένεση. Για να έχουμε αξιοπιστία, για να επιστρέψουν οι Σκοτσέζοι, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει άμεσα το θέμα της εσωτερικής διεύρυνσης. Αλλιώς θα είναι καταδικασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ε, και όλες οι άλλες αυτοκρατορίες και μάλιστα για τον ίδιο λόγο επειδή καταπίεσε ε, την εσωτερική πολυμορφία. Ε, η ηθική πηξίδα θα μας σώσει από τα τυφλά σημεία μας και προς τους φίλους μας ε, στην Σκωτία. Θέλω να πω ότι πολύ ευχαρίστως θα σας ξανακαλωσορίσουμε στην Ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής ε, και ε, Επίτροπε. Ήδη πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για τις διαπραγματεύσεις ε, για το Brexit. Όμω εγώ θέλω να μιλήσω για το άλλο σημείο πολύ σημαντικό του Συμβουλίου, που είναι ακριβώς το σχέδιο ανάκαμψης. Είναι πολύ σημαντικό εμείς ως Κοινοβούλιο να στηρίξουμε όσο μπορούμε την Κομισιόν αυτή τη στιγμή, γιατί προβλέπεται για πρώτη φορά την έκδοση ευρωμολόγων. Προβλέπει ε, μεγάλη βοήθεια σε ενισχύσεις και δάνεια. Προβλέπει να δοθεί προτεραιότητα στους μεγάλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή τη δεκαετία όπως η ψηφιοποίηση και βεβαίως η πράσινη συμφωνία των Green Deal. Επίσης ε, λυπούμαστε γιατί το Συμβούλιο στο PDP ε, περιλαμβάνει πολύ σοβαρές περικοπές. Θέλω να κάνω έκκληση στο Συμβουλίο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη, στους λιτούς, στους ε, ε πιο γαλαντόμους και τα λοιπά. Ε, ε, όλους και είναι το εξής, η εξής η έκκληση. Εάν η ανησυχία σας, αν ανησυχείτε για τις μελλοντικές γενιές, στηρίξτε το σχέδιο της Κομισιόν όπως το παρουσίασε η Πρόεδρος Βαντερ Αυτό ε, περιμένουν οι μελλοντικέ γενιές από εμά. Thank you for one minute, Mr. Moreno Sanchez. Moreno-Sánchez. sanchez Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία μηνύματα σε ένα λεπτό. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν ε, έχουμε τηρήσει την υποχρέωσή μα για υποβολή φιλόδοξων προτάσεων. Τώρα το Συμβούλιο πρέπει να φτάσει σε συμφωνία για την οικοδόμηση τη Ευρώπη και για να υπάρχουν και να φτάσουν τα χρήματα όσο γίνεται πιο σύντομα στου πολίτε, στι εταιρείε, στι περιφέρειες που τα χρειάζονται. Επίση, εκεί η ώρα για την εισαγωγή νέων ε, ιδίων πόρων τη Ένωση για να αποπληρωθεί το χρέο. Ε, Μάνφρεντ Βέμπερ και Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μην ανησυχείτε, η Ισπανική κυβέρνηση θα υποβάλει ένα σχέδιο φιλόδοξο για την ανάκαμψη που δεν θα αφήσει κανέναν πίσω. Δεν δεχόμαστε τα σχέδια του παρελθόντος, ούτε ερεσιμότητα ούτε λιτότητα θέλουμε πια. Και τέλος, στους κυρίους του ΕΛΚ και στους συμμάχους τους, παρακαλώ μην κάνετε λάθος. Αυτό εδώ, αυτή εδώ η αίθουσα δεν είναι παράρτημα του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Μην το χρησιμοποιείτε ως χαρακόμματα για να επιτεθείτε κατά της κυβέρνησης του Πέντρου Σάντσες και μάθετε να είστε πατριώτες ακόμα και όταν είστε στην αντιπολίτευση. Ευχαριστώ. Ήμουν αρκετά ανεκτική, αλλά τώρα πρέπει να είμαι πιο αυστηρή με το χρόνο. Ζητώ συγγνώμη από αυτούς που πρέπει να σταματήσω. Δίνω το λόγο στην κυρία Στέιτμεν. Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε πάλι εδώ και ε, πρέπει να δώσουμε λογαριασμό στους ε, Σουηδούς φορολογούμενους, διότι μιλάμε για αλληλεγγύη, για κοινότητα, μιλάμε για το μέλλον των επόμενων γενεών, αλλά η αλληλεγγύη δεν μπορεί να βασίζεται στο ότι ο ένας κάνει οικονομία και ο άλλος σπαταλάει. Στη σκιά του κοροναϊού αυξάνουμε ε, το ε, βάρος του χρέους ε, και συγκεντρώνουμε ακόμη περισσότερη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι όμως δεν θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα ούτε θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη στο μέλλον. Αντιθέτως απλά αναβάλουμε το πρόγραμμα και το βάρος θα το φέρουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δεν είναι αλληλεγγύη αυτό, είναι ανευθυνότητα. Next Generation EU έχετε ονομάσει τη δέσμη. Εγώ την ονομάζω ότι δεν μας ενδιαφέρει η επόμενη γενιά. Ευχαριστώ. Very much Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, κύριο Σπασέσκου, Πασέσκου, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Το Brexit φαίνεται ναι, ε, να έχει φτάσει σε στάδιο κουβέντας, ενώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια καλή συμφωνία. Πρόσφατα δεν είδαμε πρόοδο και αυτό δείχνει ότι χρειαζόμαστε παρεμβάσεις σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και νομίζω ότι είναι θετικό το ότι η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Μακρό και ο κύριος Τζόνσον προσπάθησαν να ξεκλειδώσουν τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς, διότι η έλλειψη μιας συμφωνίας θα οδηγήσει σε διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ, Μαρκές. Πρόεδρε, αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει να αντιμετωπίσει δύο τεράστιες προκλήσεις. Η πρώτη ε, είναι η ανέβρεση μιας πολιτικής συμφωνίας ε, ε, όπου να συμφωνούν όλα τα κράτη και να έχουμε και καλή πρόταση ταυτόχρονα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν απαιτητικό. Ζήτησε την αναθεώρηση τη πρόταση για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αμοιβιοποίηση των ευθυνών, ευρωομόλογα, περισσότερε επιδοτήσει και ενισχύσει παρά δάνεια, ε, αύξηση των ιδίων πόρων ω πόρο χρηματοδότηση των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζήτησε πολιτική, ε, ευρωπαϊκή πολιτική αυτές οι αρχέ αρχές είναι στο τμήμα της πρότασης της Κομισιόν. Δεύτερη πρόκληση, ε, η εξέβρεση πολιτικής συμφωνίας για το μέλλον του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μια κακή πρόταση για, το δεύτερο, για τη δεύτερη περίοδο του πλαισίου. Η απόφαση θα είναι ε, καθοριστική. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στομπέ. Ένα λεπτό. Η Ευρώπη πρέπει... Η Ευρώπη πρέπει να συμφωνήσει πάνω σε ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και, και τη δέσμη ανάκαμψης. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό με υπευθυνότητα. Δεν μπορούμε απλά να δώσουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές και γι' αυτό θέλουμε να απαιτήσουμε πολύ πιο αυστηρό ε, πρόγραμμα ε, Επιστροφή των χρημάτων. Δεν μπορεί να ξεκινήσει αυτό το 2028 και να συνεχιστεί για άλλα 30 χρόνια. Θα πρέπει να τηρήσουμε την αρχή του κράτους δικαίου και του πόρου τη Ευρωπαϊκή Ένωσης να τους δαπανούμε με σωστό τρόπο. Και τέλος, άσχετα από το τι συμβασμός θα επιτευχθεί, ε, δεν ενισχύει την ανταγωνιστικότητά μας ε, ένα δάνειο. Ε, θα πρέπει να, να είμαστε καινοτόμοι και να είμαστε πιο παραγωγικοί. Ευχαριστώ, κύριος Βίτανοφ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν οδηγήσει σε πρόοδο οι Βρετανοί έχουν μια μαξιμαλιστική προσέγγιση και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ενιαία αγορά χωρίς να αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση. Δυστυχώς η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δεν θα συνεχιστεί όταν ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος. Υπάρχουν ανησυχίες για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που αυξάνονται διότι κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων το Ηνωμένο Βασίλειο περιορίζει τα δικαιώματα αυτά. Η νομοθεσία αντικατάστασης προχωράει πιο γρήγορα από τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος μη συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιμείνει έτσι ώστε να υπάρξει μια μελλοντική συμφωνία βάσει της αμοιβαιότητας των μη διακρίσεων και λαμβάνοντα βεβαίω πάντα υπόψη τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κ. Σικόρσκι έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, όσο αναπληρωτής ε, πρόεδρος της ε, ομάδας φιλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Βρετανίας και θα ήθελα να επιτευχθεί η συμφωνία, αλλά έχω απογοητευτεί ακαιρεότητα της ενιαίας, της ενιαίας αγοράς. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να δεχτεί συμφωνία που να βάζει την Βρετανία υπό την δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή που περιορίζει το, η Βουλή των Κοινοτήτων ε, κατά καθιονδήποτε τρόπο στο μέλλον να αποφασίζει τι βρετανικέ πολιτικές. Αυτό καθιστά μια συμφωνία δύνατη να βρεθεί, γιατί η φύση μια συνθηκη οποιασδήποτε συμφωνία είναι ότι στο μέλλον θα κάνει αυτό που λέει η συνθήκη και ό,τι σου ε, ε, έρχεται. Ε, άρα λοιπόν δεν φαίνεται να υπάρχουν σημεία ε, που εφάπτονται εκεί. Δηλαδή το να ζητάμε το αδύνατο από τους διαπραγματευτές μας. Καλύτερα να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για αυτό που είναι βέβαια λυπηρό, αλλά φαίνεται να είναι πλέον αναποφευκτό. Δηλαδή ένα πολύ σκληρό Brexit. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γκαρσία Μαρκάλιο. Η αρχή των ευκαιριών, ο, ο αμοιβαίος ανταγωνισμός είναι κάτι το οποίο είχε αναγνωριστεί στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας. Είναι κάτι που επιτρέπει τη συνέχιση ενός φορολογικού καθεστώτος όπου τα ωφέλη ε, τα οποία τα κέρδη τα οποία προκύπτουν εντό του Γιβραλτάρ ε, ε, φορολογούνται και όχι αυτά που είναι εκτός και αυτό βεβαίω οδηγεί σε συγκεκριμένε επιπτώσει. 30.000 επιχειρήσει offshore στο Γιβραλτάρ και 60% ε, του, των, των παιγνίων επιγραμμικά ελέγχονται από το Γιβραλτάρ. Είναι η, το τρίτο κατακεφαλήν εισόδημα στον κόσμο. Ενώ είναι έξι φορές λιγότερο σε υπόλοιπε ε, ε, στις υπόλοιπες περιοχές της Ισπανίας ε, μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι Ηνωμένε Πολιτείε και Μεξικό. Είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει τον κώδικα το φορολογικό του Μόντι και τον κώδικα ε, που διέπει τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Δεν μπορούμε πλέον να το ανεχτούμε αυτό σε Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό σαφώς στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Στις διαπραγματεύσεις αυτές λοιπόν θα πρέπει όλοι ε, να σεβόμαστε τη διεθνή νομιμότητα σε ό,τι αφορά την αποπακιοποίηση, μια και είμαστε μια, ένα κράτο δικαίου, μια ένωση δικαίου, συγγνώμη. Ο κ. Χριστοφόρου έχει τον λόγο, παρακαλώ. Κατόμενο τη ευκαιρία τη παρουσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρισκόμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την ισχυρή δύναμη των λαών τη Ευρώπη, θα ήθελα με όλη τη δύναμη τη ψυχή μου να καταγγείλω για ένα ζήτημα το οποίο είναι αποκλειστικά και μόνο ευρωπαϊκό και θα εξελιχθεί σε ένα τραγικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι οι απειλέ οι εκβιασμοί και οι επεκτατικέ επιθετικέ πολιτικέ τη τουρκία ενάντια σε δύο χώρε μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση την ελλάδα και την κύπρο οι παράνομε οι παραβιάσει τη τουρκία στην κύπρο οι παραβιάσει στην ελλάδα το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο δεν είναι υποθέσει που αφορούν την κύπρο αλλά αφορούν ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση η ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να χρηματοδοτεί αυτήν την παράνομη εκβιαστική χώρα που πλήττει δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από θράσινα την Τουρκία και δεν νοείται την ώρα που βρίσκεται παράνομα στην Κυπριακή ΑΟΣ και παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας και τα θαλάσσια σύνορα να συνεχίζει αυτή η χρηματοδότηση. Κάνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προ τι ισχυρέ χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπιστούν τα θαλάσσια σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ίδιο τρόπο που υπερασπίζονται τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στου παράνομου μετανάστε. Εάν χρειαστεί και τελειώνω, να στείλουν ακόμα και το πολεμικό του ναυτικό να υπερασπιστεί τα θαλάσσια σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριο Σουόρπον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε μια όσο γίνεται πιο στενή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο όσο γίνεται. Είναι εταίρος μας και σύμμαχός μας ε, η ε, γεωγραφική γυτνίαση και η ε, στενές εμπορικές μας ε, σχέσεις καθιστούν αδύνατο το να μην έχουμε μια συμφωνία. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει ισχυρό ανταγωνιστή τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις θέσει απασχόλησης και τις επενδύσεις. Ε, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει πιο υψηλού στόχου ε, για την απασχόληση και την ανάπτυξη και θα πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τις εξαγωγικές μας επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις είναι ατύχες ε, ότι οι διαπραγματεύσεις ε, που ήταν περιορισμένες χρονικά συνέπεσαν ε, με τον κορονοϊό. Επικροτώ όμως το ότι τώρα λαμβάνονται νέα επικοδομητικά μέτρα πριν τις διαπραγματεύσεις του καλοκαιριού. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε ένα τον άλλον να συνεργαστούμε για καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριο Φαντάλη. Ο κύριος Βαντάλεν για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, θέλουμε μια συμφωνία που είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές. Το μόνο Βασίλειο όμως πάει πίσω και αμφισβητεί τη διαπραγμάτευση. Θέλω να ξαναδιαπραγματευτούν τα ίδια πράγματα. Ε, το ερώτημα λοιπόν ε, είναι εάν ε, η Βρετανική κυβέρνηση θέλει μια συμφωνία. Οι Βρετανικές επιχειρήσεις σίγουρα θέλουν. Ο σύνδεσμός τους θεωρούν ότι η εσωτερική αγορά είναι κρίσιμη σημασία για αυτούς ένα σκληρό Brexit ε, θα ήταν εις βάρος ε, και των δύο πλευρών. Είναι κάτι που δεν θα αντέξει η Βρετανική οικονομία. Εγώ λοιπόν θα ήθελα μια συμφωνία με δίκαιη ρύθμιση για την αλληλεία, να μας επιτρέπει να αλλιεύουμε στη Βόρεια Θάλασσα και να επιτρέπει και διατήρηση των αποθεμάτων. Εάν δεν λύσουμε το θέμα της αλληλείας δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια εμπορική συμφωνία. Ευχαριστώ κυρία Σπυράκη ευχαριστώ κυρία πρόεδρε αντιπρόεδρε σεφκοβιτ κυρίε και κύριοι συνάδελφοι οι χαμηλέ προσδοκίε που καλλιεργούνται εν ώψη του ευρωπαϊκού συμβουλίου υπονομεύουν το κλίμα αισιοδοξία και εμπιστοσύνη που έχουν ανάγκη οι πολίτε μα και οι οικονομίε μα. στη χώρα μου την ελλάδα αφού χάσαμε το 25% πέντε του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης είμαστε τώρα αντιμέτωποι με βαθιά ύφεση εάν η ευρωπαϊκή ένωση δεν δράσει άμεσα γι' αυτό και είναι απαραίτητο το ευρωπαϊκό συμβούλιο να δράξει την ευκαιρία και να στείλει στις αγορές ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης να δείξει ότι η ευρωπαϊκή ένωση είναι έτοιμη να εγγυηθεί το μέλλον της γενιάς της. το ταμείο ανάκαμψης σε συνδυασμό με τον κοινοτικό προϋπολογισμό μπορούν να στηρίξουν την υψηλής ποιότητας πρωτογενή παραγωγή τον εξηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές σε συνδυασμό με θέσεις εργασία στην κυκλική οικονομία την ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα και τη διασύνδεσή του με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τώρα δίνουν μάχη να ξανανοίξουν. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τα χρήματα από τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια οφείλουν να δοθούν ώστε οι οικονομίες μας να μετασχηματιστούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τη γενιά μας και για την επόμενη γενιά. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα οι μας. Πρώτα η κυρία Πύρη για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους σε αυτή τη συζήτηση και για την συνεχή υποστήριξη. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω όλου ιδιαίτερω τον συνάδελφο, την εισηγητή, τον κύριο Κρίστοφ Χάνσον και όλου του σχεδόν εισηγητέ που εργάστηκαν επί του φακέλου αυτού. Και βεβαίω δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι ευχαριστίε και προ τον Μισελ Μπαρνιέ και την ομάδα του για την απόλυτη ε, δέσμευσή τους, στη συνεργασία τους μαζί μας. Τους ευχόμαστε πολύ κουράγιο και πολύ χιούμορ το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που χρειαζόμαστε με τη συμφωνία αυτή δεν είναι βραχυπρόθεσμε απαντήσει. Χρειαζόμαστε ένα πιο μακροπρόθεσμο όραμα, διότι είναι τεράστιε οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Εάν η κυβέρνηση του Βασιλείου δεν αλλάξει άμεσα και ριζικά την προσέγγιση τη, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να φτάσουμε σε κάποια εταιρική σχέση πριν το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Και για να είμαι ειλικρινής, υπό τις παρούσες συνθήκες νομίζω ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για μια μη συμφωνία. Τα δεδομένα από το Στατιστικό Γραφείο των, των Βασιλείου της περσμένης εβδομάδας δείχνουν σαφώς τον οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης του κορονοϊού. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει η αφήγηση. Η πανδημία να είναι ο λόγος για την επιτυχία και όχι ε, ο λόγος για την αποτυχία. Αλλιώ θα ήταν τραγικό. Χρειαζόμαστε συμφωνία και μπορούμε να έχουμε συμφωνία που να είναι καλή για όλους. Η μη συμφωνία δεν έχει νόημα και δεν είναι και υπεύθυνο. το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι η στιγμή της αλήθειας. Ήρθε η ώρα για την ευθύνη και το θάρρος. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ασφάλεια, χρειάζονται προβλεψιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παίξει το ρόλο της και ε, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις προσδοκίες της. Και τώρα το λόγο για δύο λεπτά έχει ο κύριος Χάνσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφοι, σα ευχαριστώ όλου για τι συμβολέ σα. Ε, μακάρι να μπορούσα να απαντήσω σε κάθε μια από τι παρατηρήσει σα. Ε, δεδομένων όμω των περιορισμών, θα επανέλθω σε κάποια από τα πιο ουσιαστικά από τι παρατηρήσει που άκουσα για το level playing field, το ισότιμο πεδίο. Ο πατέρα μου δεν μιλά αγγλικά. Με ρωτά πάντα γιατί ε, όταν ε, μιλά στο ραδιόφωνο μιλά για αυτό το level playing field. Τι σημαίνει. Και μετά το έμαθα, επειδή είμαστε και οι δύο, είμαστε πολύ ε, φανατική οπαδή της ποδηλασίας του είπα, φαντάσου εκεί στη γύρω της Γαλλίας να είναι κάποιοι που ε, τρέχουν με τα ποδήλατα ε, τα κανονικά και άλλοι με τα πιο εξελιγμένα τελευταία ε, λέξη τεχνολογία. Ή θα ήταν δίκαιο αυτό, όχι, δεν θα ήταν δίκαιο μου απάντησε. Θα θέλουμε να έχουμε δίκαιο ανταγωνισμό. Ακριβώ περί αυτό πρόκειται. Θέλουμε καλή συνεργασία και στενή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό είναι προ όλων το συμφέρον. Ε, θα δουλέψουμε για ισορροπημένε και δίκαιε συμβιβαστικέ που ελπίζουμε να αναδυθούν τι επόμενε εβδομάδε εδώ στι Βρυξέλλε και στο Λονδίνο. Φυσικά, όπω είπαμε, χρειάζονται και τα δύο μέρη να συνεργαστούν. Όπως είπε πριν και ο Επίτροπος, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ε, και εμείς είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο αυτό χώρο. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, αγαπητέ φίλε, συνάδελφε, ε, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ε, Μισελ Μπαρνιέ. Κάποιες παρατηρήσεις ε, ανέφερε η κυρία Γκαρσία η κυρία ε, Κέλλερ, βεβαίω είναι και η τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το, αυτή την Παρασκευή για το PDP και το Next Generation EU. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τις συζητήσεις μας για τα ευρωπαϊκά και με το κοινό. Δεν χάνουμε ούτε λεπτό, σας διαβεβαιώ, από το χρόνο που τώρα έχουμε πια μπροστά μας, που ελπίζω ότι θα είναι πολύ σημαντική, ε, ιστορική και φιλόδοξη ε, συμφωνία για το Next Generation και το... Ε, ε σχέδιο ανάκαμψης ε, συζητάμε με τους εκπροσώπους ε, των κρατών και μάλιστα εγώ μιλούσα για, με τους εκπροσώπους Εθνικών Κοινοβουλίων μόλις την περασμένη Πέμπτη ε, και τους εξηγούσα για το πώς, ε, ποια είναι η αρχιτεκτονική αυτού του νέου ταμείου. Βεβαίω, η αλληλεγγύη είναι must και πιστεύω πως αυτή δηλαδή, η διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μας επιτρέψει να περιορίσουμε τις διαφορές μας ε, που εξακολουθούν να υπάρχουν και να προετοιμάσουμε καλά το έδαφος ώστε να φτάσουμε σε μια καθοριστική και αποφασιστική κίνηση για συμφωνία τον Ιούλιο. Το δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε από τους υπόλοιπους ε, βουλευτές να σας ενημερώσω για το πώς θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία απόσυρσης. Όπως ξέρετε, εγώ εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κοινή επιτροπή, μειχτή επιτροπή με τον Μάικλ Γκόλ που εκπροσωπεί την Βρετανική κυβέρνηση. Και μιλάμε για τη συμφωνία που εγκρίθηκε και υπογράφηκε και κυρώθηκε από το Κοινοβούλιο και από το Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας. Και ε, μάλιστα έγινε σε δήλωση από το ΜΑΙΚΟ ότι δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω παράταση της μεταβατικής περίοδου. Ακούσαμε ε, από τον κύριο Πύρη, τον κύριο Χάνσεν και από τον κύριο Μακάλιστερ ότι χρειάζεται να επιταχύνουμε τη δουλειά μας και να εξασφαλίσουμε πως η συμφωνία απόσυρση θα εφαρμοστεί σωστά. Εγώ με χαρά ανακοινώνω, αναφέρω ότι η συζήτηση στην Κοινή Επιτροπή ήταν πολύ θετική, για την, έγινε σε πολύ θετική ατμόσφαιρα, ήταν πολύ καλή πρόεδρος στο τομέα των δημοσιονομικών προβλέψεων για το πρωτόκολλο για το Γιουραλτάρ, για τις ε, κυρίαρχες βάσεις ε, του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο και για τα δικαιώματα των πολιτών επίσης, που ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για το Ευρωκοινοβούλιο και τους πολίτες μας ε, και όπου πιστεύω θα μπορέσουμε να λύσουμε λύσουμε αυτές μας τις διαφορές οριστικά πριν το τέλος του χρόνου. Αυτό που είναι το πιο δύσκολο είναι ε, βέβαια η εφαρμογή του πρωτοκόλου για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Και εδώ ήμουν σαφής και ε, το κατέστησα σαφές και στην αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου ότι πρόκειται ε, για μια δύσκολη διαδικασία ε, αλλά για μας είναι σημαντικό να έχουμε ε, απαντήσεις για το συγκεκριμένες για το πώς θα εφαρμόσει το σύστημα ΦΠΑ, τους δασμούς, τους τελωνιακούς και ούτω καθεξής που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία απόσυρσης και η απάντηση του Michael ήταν ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά στη διάρκεια του καλοκαιριού, θα φτιάξουμε και μία ακόμα ειδικευμένη επιτροπή για το Ιρλανδικό πρωτόκολλο θα συγκληθεί τον Ιούλιο και πιστεύω πως θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να το συζητήσουμε μαζί στο Σεπτέμβριο. Ε, πολύ δουλειά λοιπόν, αλλά πιστεύω πως ε, τελικά και οι δύο πλευρές καταλαβαίνουν ότι η σωστή εφαρμογή είναι κλειδί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και για, το, και για αγαστές μελλοντικές σχέσεις ανάμεσα στην Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο και πώς τι εικόνα θα έχουν αυτές οι μελλοντικέ σχέσεις. Θα μου επιτρέπετε, Προέδρε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπαρνία γιατί νυχθημερών διαπραγματεύεται με τους Βρετανούς μας συναδέλφους και μπορεί να σας δώσει καλύτερη εικόνα. Έχετε το λόγο, κύριε Μπαρνία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστώ και τον Μάρος. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Να πω κι εγώ δύο λόγια μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σεύκοβιτς για τη διαπραγμάτευση αυτή που είναι εξαιρετικά περίπλοκη, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά το Κοινοβούλιο, κυρία Πρόεδρε, τις 17 επιτροπές, των εισηγητή. Ε, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά την Κέιτι Πέρι, και τον Κριστόφ Χάνσεν για αυτή την, το δύσκολο έργο σύνθεσης το οποίο επετέλεσαν. Χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα αλλά και επαγρύπνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτή η αποφασιστικότητα είναι που εξέφρασε ο πρόεδρό σα, ο κύριο Σασόλη, στην διάσκεψη ψηλού επίπεδου που οργανώθηκε μαζί με την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τον Σαρλ Μισελ, εσά και τον Μπόρι Τζόνσον. Και βεβαίω, ε, νομίζω το είπε η Ανταλή Λουαζό προηγουμένω, θα έχετε και το τελευταίο λόγο. Ε, όταν θα έχουμε φτάσει, ελπίζω, σε μια συμφωνία με το Μένο Βασίλειο. Ο Μάρο Εύκοβιτ μόλι ε, σημείωσε ότι βεβαίω και λάβαμε γνώση της αρνητικής στάσης του Βασιλείου σε ό,τι αφορά την παράταση της μεταβατικής περίοδου ε, έως τις 30 Ιουνίου. Είναι μια περίοδος διαπραγμάτευσης κανονικά αυτή. Είναι δικαίωμα του Ηνωμένου Βασιλείου να το κάνει αυτό. Είμαστε λοιπόν στα μέσα, τέσσερι μήνε πίσω μα, τέσσερι μήνε μπροστά μα. Η Κέτι Πέρι είπε 204 μέρε νωρίτερα. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα, αλλά γίνεται. Γίνεται. Είναι λίγο ο χρόνο. Ε, Καταλαβαίνομαι και εγώ ότι επήγει να βρούμε μια λύση. Το είπε και ο Τζόνσον αυτό. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε με τον David Frost και την ομάδα του τον ε, συνδιαπραγματευτή μου ε, που ε, φέρεται πολύ επαγγελματικά να αντικοποιήσουμε τις συζητήσεις τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, πιο πολλές συναντήσεις, πιο στοχευμένες, με την υποχρέωση βέβαια για μας, αυτός είναι ο κανόνας για μένα, να υπάρχει διαφάνεια απέναντι στο Κοινοβούλιο, στη συντονιστική ομάδα, στις επιτροπές σας και με 27 κράτη-μέλη βέβαια, ε, στο όνομα των οποίων διαπραγματευόμαστε. Ποια είναι τα επόμενα στάδια τώρα. Ένα είναι σίγουρο, όπω ε, υπενθύμησαν οι τρει πρόεδροι τριών θεσμικών οργάνων όταν συνάντησαν τον Μπόρι Τζόνσον τη Δευτέρα, αυτό που έχει σημασία για μα πριν κάνει τη διαδικασία την ίδια είναι να προχωρήσουμε επί τη ουσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό που θα πρέπει να διαλέξει τι θέλει και αν θέλει συμφωνία. Το είπατε πολύ καλά ε, κυρία Μπρέσνατς προηγουμένως ε, στην αρχή της ε, συνάντησης είναι επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου το αν θέλει ή δεν θέλει συμφωνία διότι οι προϋποθέσεις για τη συμφωνία είναι γνωστές τη συμφωνήσαμε με τον κύριο Τζόνσον το κάθε κόμμα ήταν αντικείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης στην πολιτική δήλωση για να πάμε προς μια βιώσιμη και φιλόδοξη εταιρική σχέση όχι μόνο μια εμπορική συμφωνία χωρί προηγούμενο, μηδέν ποσοστώσει, μηδέν δασμοί για όλα τα αγαθά, δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία στο παρελθόν, αλλά και με συμφωνία ε, στον τομέα τη Αλία, το σύνθημα ο κ. Μπελαμή, και βεβαίω για το ίσο ε, πεδίο ευκαιριών, level playing field, περιβαλλοντικά κοινωνικά δικαιώματα, ε, ίση πρόσβαση στην αγορά κτλ και όπως είπε ο κ. Χάνσεν υπάρχει ένα θέμα οικονομικού και κοινωνικού fair play. Πρέπει να καλύπτει και την ενέργεια, τι μεταφορέ, την ασφάλεια, την άμυνα. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η προσφορά άνευ προηγουμένου και θέλουμε και πρόσβαση ε, στην αγορά μας να διέπεται από δίκαιες συνθήκες. Αυτά, αυτές τις αρχές τις έχουμε ασπαστεί στην εντολή μας και στο σχέδιο συμφωνίας που δημοσίευσαμε στις 18 Μαρτίου. Και βεβαίως αυτό δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγμάτευσης, διαπιστώνουμε, κύριοι βουλευτές, ε, ποια είναι η στρατηγική του Βρετανικού, της Βρετανικής κυβέρνησης. Στην αρχή δεν ήθελε καμία συζήτηση για τα σημαντικά ζητήματα. Άμυνα, ασφάλεια, ανάπτυξη. Εγώ αυτό το είχα ερμηνεύσει ως μια ιδέα του να συγκεντρώσουμε όλη τη συζήτηση μόνο στα οικονομικά θέματα. Μόνο δηλαδή στην υπεράσπιση, στην προάσπιση των δικών τους οικονομικών συμφερόντων. Στη συνέχεια, στα πλαίσια στρατηγική αυτή, το Μένο Βασίλειο θέλει να διαπραγματευτεί σε κάποιου τομεί ένα καθεστώ πολύ πολύ κοντινό ε, στο να είναι κάποιο μέλο τη ενιαία αγορά, τη Σέγγεν, τη Τελωνική Ένωση, χωρί όμω τι υποχρεώσει που ε, προβλέπονται cherry picking για την αμοιβαία αναγνώριση, του κανόνε προέλευση, τι επαγγελματικέ δεξιότητε, τι ροέ δεδομένων, την ανταλλαγή στον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά δεν θα το δεχτούμε εμεί. Δεν μπορεί να διαλέγει το ΗΠΑ Βασίλειο ό,τι θέλει. Το δεύτερο κομμάτι τη στρατηγική των Βρετανών είναι να αρνείται οποιαδήποτε δέσμευση στον τομέα του level playing field, των ίσων ευκαιριών, έτσι ώστε να μπορεί ανα πάσα στιγμή να απομακρυνθεί από του παρόντε κανόνε τη Ένωση και βεβαίω να ε, ανταγωνιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο λόγο ύπαρξη του Brexit, λένε κάποιοι. Και βλέπουμε τη στρατηγική αυτή για τα δεδομένα. Γνωρίζω ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, βέβαια. Για τι οικονομικέ ε, υπηρεσίε, τι κρατικέ ενισχύσει. Ο Πρωτομένο Βασίλειο τώρα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη σε ό,τι αφορά το εθνικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Ε, το βλέπω και για τους, ε, τις προδιαγραφές της, Μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο θέλησε να ξανανοίξει το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται σαφώ όμω στη συμφωνία απόσυρση στην οποία αναφέρθηκε ο Μάρο Εύκοβιτς. Όλα αυτά δεν είναι συμβατά με τι βάσει μια βιώσιμη φιλόδοξή συμφωνία με μια μεγάλη χώρα ε, που θα παραμείνει μια χώρα φίλος και σύμμαχος κατά πάσα πιθανότητα. Είμαι παρόλα αυτά πεπισμένος κύριε και κύριοι ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία. Μια συμφωνία μακροπρόθεσμη όπως είπε η κυρία Χούμπνερ εμείς αυτής της αρχής το επιθυμούμε αυτό, το προσδοκούμε. Εξού και η ιδιωτικοποίηση των γραμματεύσεων. Όμω, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, όπω ε, ε, στο ψήφισμά σα αναφέρεται, δεν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία πάση θυσία. Το είπε ο Μπέντ Λάγκε νωρίτερα. Δεν πρόκειται ε, να ε, θυσιάσουμε, όπω είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν, τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, τα μακροπρόθεσμα των καταναλωτών και των επιχείρησεων τη Ένωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ταυτόχρονα θέλουμε απτά, απτή πρόοδο ό,τι αφορά τη συμφωνία απόσυρσης ε, ε της για τα δικαιώματα των, ε, των, πολιτών και αυτό έχει να κάνει βεβαίω και με την ε, ε, ειρήνη στην Ιρλανδία, με σωστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Εάν θέλουμε λοιπόν ως προτεραιότητα να φτάσουμε σε συμφωνία, ταυτόχρονα, και το είπε ο κ. Αριμών και ο κ. Σέρντεμαρ προηγουμένω, πρέπει να προετοιμαστούμε συλλογικά για όλα τα σενάρια στο τέλο του έτους. Είτε υπάρξει συμφωνία είτε δεν υπάρξει. Εμεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα ετοιμαστούμε. Θα είμαστε έτοιμοι. Σα ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σα, σα ευχαριστώ που εμπιστεύεστε την ε, διαπραγματευτική ομάδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι η δική σα διαπραγματευτική ομάδα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Τις επόμενε εβδομάδε που θα είναι ε, ε, ε, κρίσιμες θα πρέπει να επιδείξουμε κάποια ποιοτικά στοιχεία μου είπε η κυρία Πέρι να επιδείξω χιούμορ. Έχω σημειώσει πρόοδο σιγά σιγά σε επίπεδο Είναι σημαντικό έτσι να προοδεύω ακόμα στην ηλικία μου. Να παραμείνω ψύχρεμο, μου είπε ο κύριο Ντάνιελσον. Να είμαι υπομονετικό. Είναι η υπομονή μου και η, ηρεμία μου είναι ε, ατελείωτη η δική μου. Να είμαστε αποφασιστικοί βεβαίω ταυτόχρονα και να είμαστε ενωμένοι το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλλον για άλλη μια φορά μα το απέδειξε αυτό σήμερα και σα ευχαριστώ. Thank you very much and I hope your reserves... Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαρνιέ. Ε, καλή δύναμη σας εύχομαι στις διαπραγματεύσεις και δίνω ε, το λόγο στην ε, κυρία Υπουργό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, πρώτα λίγα λόγια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το, Ηνωμένο, με το Βασίλειο. Ε, κάτι στο οποίο αναφερθήκατε αρκετοί από εσά. Ε, πιστεύουμε ότι ο διαπραγματευτής μας ε, θα πρέπει να είναι σε καλύτερη θέση ε, για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις με τις παρατηρήσεις σας συμφωνία αποχώρηση θα έπρεπε να συνοδεύει τι διαπραγματεύσει ε, για την ε, συμφωνία εταιρική σχέση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε όσον αφορά καταρχά ε, την διατήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών σε οποιαδήποτε μελλοντική σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά θα πρέπει να επαγρυπνούμε επίσης όσον αφορά τη την μελλοντική εταιρική σχέση θα χρειαστεί σωστή διακυβέρνηση για να προστατεύσουμε την ε, ενιαία αγορά και τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα βασιστούμε ε, στη δική σας υποστήριξη με τις κοινέ μας προσπάθειες και τον κοινό μας στόχο θα παράσχουμε την ε, υποστήριξη που χρειάζεται ε, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχέδιο ανάκαμψης, ε, ε, η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέλει να δώσει στους ηγέτες τη δυνατότητα να συζητήσουν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχέδιο ανάκαμψης και γι' αυτό η συνάντηση του, ε, της Παρασκευής ε, θα είναι μια ευκαιρία να εξηγήσουν οι ηγέτες πώς βλέπουν τις... Ε, πώς βλέπουν τα θέματα αυτά. Ε, με βάση αυτά, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για να ε, προετοιμαστεί για το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων και να πετύχει μια ε, καλή συμβαστική λύση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι απομένουν πολλά να γίνουν για να συμφιλειωθούν ε, διστάμενες ε, απόψεις ε, και συμφέροντα και να υπάρξει συμβιβασμός. Ο τελικός μας στόχος είναι να υπάρξει όσο γίνεται συντομότερα συμφωνία πάνω σε ένα άνευ προηγουμένου οικονομικού πακέτου για να αντιμετωπιστεί και μια άνευ προηγουμένου κρίση. Θα συνεχίσουμε να είμαστε προσιλωμένοι, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, θα διευκολύνουμε κάθε βήμα προς μια τέτοια συμφωνία και θα το κάνουμε αυτό με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις του Κοινοβουλίου, διότι ήταν σαφές ε, με την πανδημία ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση μόνο εάν είμαστε αλληλέγγυοι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Τέλος της κοινή συζήτηση. Ήδη ψηφίσαμε τις τροπολογίες της κυρίας Πύρη και ε, της έκθεσης της κυρίας Πύρη και του κυρίου Χάνσεν. Τελική ψηφοφορία αύριο το πρωί. Πριν ε, κλείσω τη συνεδρία θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω τους διερμηνείς ε, διότι διήρκησε η συζήτηση περισσότερο από όσο είχαμε προβλέψει. Ευχαριστώ ειλικρινά τους διερμηνείς. Διακοπή της συνεδρίασης μέχρι τις 7.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

και Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο τη διάταξη, που είναι δηλώσει ε, του Συμβουλίου και τη Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Θέλω να σα ενημερώσω ότι δεν ε, μπορείτε να στήσετε αυθορμήτω το λόγο, ούτε θα γίνουν δεκτέ μπλε κάρτε στη συζήτηση αυτή. Καταρχάς, θα ήθελα δώσω το λόγο στην Υπουργό Πρινίτσα για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας παρακαλώ. Thank you, President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξανασυζητήσουμε τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Και μάλιστα αυτή η σκέψη είναι σημαντικότερη από ποτέ και η συζήτηση, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε πρωτοφανείς προκλήσεις. Ε, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Ε, έχει αλλάξει μάλλον ριζικά από τον Ιανουάριο που το είχαμε πρώτο συζητήσει στην Ολομέλεια. Γιατί στο μεταξύ η πανδημία COVID-19 άφησε ανεξίτηλα και βαθύτατα ίχνη στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας και έθιξε τους πάντες και τα πάντα, ακόμη και την άποψή μας για την διάσκεψη. Για προφανείς λόγους, τους τελευταίους ε, μήνες και εβδομάδες χρειάστηκε να επικεντρωθούμε στις πιο επίγουσες προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους πολίτες και πρώτα απ' όλα την έκτακτη ανάγκη της υγείας και τις οικονομικές και κοινωνικές της συνέπειες. Πάντως, αν μας έδειξε κάτι η κρίση, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε από κοινού το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου η Προεδρία είναι δεσμευμένη να διευκολύνει η συνένεση στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία με το, Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή, με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμα, το αντικείμενο και τη γενική διοργάνωση τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε το συντομότερο συμφωνία στο Συμβούλιο για το σημαντικό αυτό θέμα. Συνεχίζεται βέβαια το έργο μα και έχει ενταθεί τι τελευταίε εβδομάδε σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσωπιών, υπουργικό και άλλα πολιτικά επίπεδα. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργό τη Κροατία, ο κύριος ε, επισήμενε την σημαντική κοινοβουλευτική διάσκεψη που θα έχει διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και η ανάγκη να λάβουμε υπόψη και το, την άποψη των πολιτών και κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό καθώς και σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 26 Μαΐου η Προεδρία οργάνωσε και μία ε, συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης με στην ε, εξαποστάσεως ε, Υπουργική Διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών. Οπότε το θα πρέπει φυσικά στην οργάνωση της διάσκεψης να λάβουμε υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και γι' αυτό τροποποιούμε τώρα το αναθεωρημένο κείμενο της θέσης του Συμβουλίου ώστε να λάβουμε υπόψη και την πραγματικότητα που δημιουργήθηκε με την πανδημία COVID-19 και φυσικά σημειώνουμε και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διάσκεψη που θα ψηφίσετε σε αυτή την Ολομέλεια και που φυσικά αντικατοπτρίζει τη νέα πραγματικότητα. Πιστεύουμε πάντως ότι η φύση της διάσκεψης και το περιεχόμενό της δεν θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτικών μας μέσω και πρόθεσμα ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ε, όσο περισσότερες απόψεις γίνεται. Τα διδάγματα πάντως της πανδημίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προβληματισμό μας ε, για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί η κρίση έχει καταδείξει πόσο σημαντικές είναι οι ήδη ε, προκαθορισμένες ε, προτεραιότητες της στρατηγικής ατζέντα μας για το 2021 και 2024. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά, να υλοποιήσουμε την περιβαλλοντική μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση και να έχουμε αυτά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Πρώτα απ' όλα πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επικείμενη διάσκεψη θα πρέπει να μην αποκλείει κανέναν, να, να συμπεριλαμβάνει και τα τρία θεσμικά όργανα με σεβασμό της διοργανικής ισορροπίας και των διαφόρων ρόλων των θεσμικών οργάνων. Επίσης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει ισότιμα να εμπλακούν και να αναμειχθούν και με τις, τα εθνικά του κοινοβούλια. Και φυσικά θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε εκτίμα αυτή τη διάσκεψη. Τέλος, για να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητές μας και να καθορίσουμε το μελλοντικό μας όραμα για την Ευρώπη σε ένα δεκαετή, εικοσαετή ορίζοντα, η συνεργασία των θεσμικών οργάνων είναι επιτακτική ανάγκη. Και όπως μας υπενθύμισε και η πανδημία, οι διενέξεις και οι διαφορές, οι διαφωνίες μας αποδυναμώνουν. Εν τη ενός ισχύς, μόνο με κοινή συνεργασία θα, μπορούσα, θα μπορέσουμε ενωρατικά να διαμορφώσουμε το μέλλον μας. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Τώρα Εκ μέρου ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο έχει η Αντιπρόεδρο, η κυρία Ντομπραφκά Σουίτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, την τελευταία φορά που είχα την ευκαιρία να σας μιλήσω όσον αφορά την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ήταν στις 15 πρώτου. Πριν λίγους μήνες. Από τότε άλλαξε πολύ ο κόσμος. Δεν έχουμε ακόμα βρει την έξοδο από την κρίση, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι επιπτώσεις θα έχει η κρίση επί του έργου μας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης τώρα είναι πιο σημαντική από ποτέ άλλοτε. Πρόκειται για ε, μια δοκιμασία, μια δοκιμή για δημοκρατική συμμετοχή. Οι κοινέ αξίε είναι το επίκεντρο ε, και είναι η ανθεκτικότητα τη κοινωνία μα και πάνω σε αυτό θα χτίσουμε την ανάκαμψη από την κρίση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία προς τα εμπρός, φιλόδοξα και με όραμα. Οπότε ε, η δική μας δουλειά είναι να απευθυνθούμε σε όλους. Η πανδημία έδειξε πόσο σημαντική είναι η ελληνική και επίσης το πώς ε, μπορούμε να βγούμε πιο δυνατοί, να ανακάμψουμε να ανασυγκροτηθούμε όπως τα είπε πρόεδρος Φοντερ εδώ σε αυτό το ημικύκλιο και συμφωνώ ότι μόνο από κοινού μπορούμε να χτίσουμε το παρόν και το μέλλον αυτό που αξίζουν οι πολίτες και μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για το μέλλον και για το παρόν υπάρχει αυτό το ξεκάθαρο πλάνο της Κομισιόν για να βρούμε την διέξοδο από την κρίση και επίσης έχουμε έτσι μια βιώσιμη ανάπτυξη, ε, προστασία του περιβάλλοντος, ψηφιακή μεταρρύθμιση όπως ζήτησε το Συμβούλιο και επίσης έχουμε ένα σφαιρικό πακέτο για την ανάκαμψη 1,85 Τρεις είναι η και έτσι ελπίζουμε να ανακάμψει η Ευρώπη και θα υποστηρίξουμε ένα σωρό κλάδους ε, βγαίνοντα από την περίοδο των περιοριστικών μέτρων πρωτοβουλίες όπως το Next Generation EU. Έτσι θα βοηθήσει ο προϋπολογισμός τα πρώτα ε, κρίσιμα χρόνια. Θα βοηθηθεί δημοσιονομικά λοιπόν ο κόσμος ε, για την περίοδο 21 με 27 επίσης θα έχουμε μια κοινωνία δίκαιη χωρίς να αφήνουμε κανένα απ' έξω. Θα βοηθήσουμε τους ε, μειονεκτούντες, αυτούς που έχουν φυγεί περισσότερο από την κρίση. Μαζί θα βρούμε την διέξοδο από την κρίση. Η διάσκεψη αυτή είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο ούτω ώστε να εμπλακούν όλοι οι Ευρωπαίοι. Περιμένω πώς και πώς την κοινή δήλωση, διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συμβούλιο και Κομισιόν. Και κάποια στιγμή αργότερα θα ξεκινήσει αυτή η διάσκεψη. Άλλαξε η πολιτική. Δεν είναι business as usual. Θα πρέπει με θάρρος να προτάξουμε τις πεπιθήσεις μας και να δώσουμε στον κόσμο αυτό που ζητεί. Αυτή είναι η εντολή μας. Πρέπει να δυναμώσουμε περισσότερο την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και να δοθεί η ευκαιρία για μια αναβαθμισμένη συμμετοχική δημοκρατία. Οπότε και εγώ ποντάρω στη δική σας βοήθεια να γίνει η κοινή δήλωση το συντομότερο να συμφωνήσουμε όσον αφορά τη δομή, ε, το, το, το, το πεδίο ε, τα βασικέ αρχέ που θα διέπουν αυτή τη διάσκεψη με, τους, ε, με τα θεσμικά όργανα που, με όλου που θα συμμετάσχουν εκεί. Στο, στην συνάντηση τη Κόζακ τη προάλλε είπαν τα εθνικά κοινοβούλια ότι θέλουν να λάβουν μέρο σε αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει επομένω αυτή η προσέγγιση να εδραιωθεί. Εδώ δεν κάνουμε κόντρα. Εδώ θέλουμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αγγίξουμε και να απευθυνθούμε σε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο και υπολογίζουμε το Συμβούλιο να μπορέσει να συμφωνήσει μια εντολή για να ξεκινήσουμε κι εμείς τις διαπραγματεύσεις. Θα γίνουν εκείνη, εκείνη η δήλωση και έτσι να ξεκινήσει το νωρίτερο η διάσκεψη. Αυτά πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας πω δύο λόγια για τη δημοκρατία και τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ότι ε, τη σήμερα ημέρα ο κόσμος θεωρεί ότι έχει μείνει πίσω, τον έχουμε εγκαταλείψει και πολλές φορές κατηγορεί την δημοκρατία. Ε, αυτό είναι ατυχές. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνει το πόσο σημαντική είναι η δημοκρατία στην καθημερινή ζωή. Ποιο, αυτός που είναι εδώ σήμερα θα μπορούσε να σκεφτεί το πόσο θα έφυγε ε, με διαφορετικούς τρόπους την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα τη χτυπούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ο COVID-19. Περισσότερο από ποτέ τώρα είναι σαφές ότι δημοκρατία και οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι κλειδί, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Οπότε ε, ε, ε, καταλαβαίνουμε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προ τη δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται κάτι το αυτονόητο. Οι πολίτε ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή στη χαρακτήρα τη πολιτική και θα πρέπει και εμεί να του αφουγκραστούμε. Όμω η κοινωνία και οι πολίτε θέλουν να θωρακιστεί η Ευρώπη. Οπότε και εμεί α καινοτομήσουμε με καινοτόμα μέσα να κάνουμε όλα αυτά που θέλει ο κόσμο. Και ξεκινάμε ε, αυτή τη διαδρομή με την διάσκεψη. Και κλείνω υπενθυμίζοντας σας το γιατί γίνεται αυτή η διάσκεψη. Γίνεται για τις σημερινές αλλά και τις επόμενες γενιές Ευρωπαίων. Οπότε πολίτες και θεσμικά οργάνα θα μπορέσουμε να, να βρούμε το πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι να έχει πιο αποτελεσματικό ρόλο ε, και ας ε, πετύχουμε σε αυτό μας το έργο τη διάσκεψη για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ο συνάδελφος ο κύριος Ρανζέλ έχει τώρα το λόγο για δυόμιση λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο του Συμβουλίου και την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχόλιά τους. Το πρώτο ουσιώδες σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι πολύ καλή η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι φιλοευρωπαϊκές παρατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατάφεραν αυτές οι φιλοευρωπαϊκές ομάδες ε, να καταλήξουν σε συμφωνία σε ό,τι αφορά τη θέση τους για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Είμαστε ενωμένοι λοιπόν και έχουμε, έχουμε ένα κοινό όραμα για αυτό που θα πρέπει να αποτελέσει η διάσκεψη και το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει. Σήμερα όπως φαίνεται ότι ανακάλυψε και το Συμβούλιο πρόσφατα, σήμερα η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης έχει πολύ μεγάλη σημασία από ότι, πολύ μεγαλύτερη σημασία από ότι πριν από, ένα πριν από ένα εξάμεινο. Και πριν από ένα εξάμεινο είναι σημαντική, αλλά σήμερα είναι σπουδαιότερη από ποτέ, γιατί η πανδημία δεν δημιούργησε νέα προβλήματα, αλλά ανέδειξε τα υπάρχοντα προβλήματα. Γι' αυτό και σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν οι συμπολίτε μας και εμείς τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από τη μια τους ε, πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους μεγαλεπίβολους και μακρόπνους στόχους, αλλά να βρούμε και τα προβλήματα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τα, τις ελλείψεις που έχουμε στη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών. Και α, ε, οι προτεραιότητες και οι στόχοι που ήταν και αρχικά της διάσκεψης σήμερα είναι πιο σημαντικοί από ποτέ. Το δεύτερο και σημαντικό σημείο είναι ε, σημαντικό να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να ενημερώνουμε τους πολίτες ε, και να προσφέρουμε έργο με αυτή τη διάσκεψη, να έχουν αυτά αποτελέσματα και οι πολίτες από τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Και γι' αυτό ζητώ από το Συμβούλιο να λάβει μία θέση επιτέλους, να καταλήξει απόφαση και να διαμορφώσει τη θέση του απέναντι στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ωραία λόγια ακούμε μονίμως. Πολύ α, ωραία λόγια από την Προεδρία, αλλά καμία πρόεδρο, πρόοδος, καμία δράση και εξακολουθούμε να προσκρούμε στη διστακτικότητα και την απροθυμία του Συμβουλίου. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα προ Ευρωπαίου πολίτε. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για το δημοκρατικό έλλειμμα και να καθυστερούμε συνεχώ και στη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Νομίζω ότι οι πολίτε ε, αξίζουν καλύτερη μεταχείριση και γι' αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να καταλήξει σε απόφαση για τη θέση του και να προωθήσουμε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία που έχουμε ενώπιόν μα. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφο Γκαρθία Πέρεθ από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Οι περισσότερε προκλήσει ε, δεν γνωρίζουν σύνορα. Σύνορα πρόκειται για τι ε, ανισότητε, ψηφιοποίηση, κλιματική αλλαγή. Είναι προκλήσει μεταξύ άλλων που τι αντιμετωπίζουμε χωρί ε, να έχει καμία σημασία το που ζούμε. Πρέπει να επιταχυνθούν οι αλλαγέ και στο σύστημα λήψη αποφάσεων στην Ένωση. Από την ομοφωνία πρέπει να περάσουμε σε ό,τι αφορά σημαντικέ πτυχέ στο σύστημα τη ομοφωνία. Και πριν από την κρίση του COVID-19 είχαμε πει Θέλουμε μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για να ορίσουμε το μέλλον μας, ε, που είναι ακόμα κάτι πιο αναγκαίο σήμερα με την COVID-19 φάνηκαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες της Ένωσης. Πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά, όπως έλλειψη ε, αρμοδιοτήτων και ευθύνη στα υγειονομικά θύμα, ε, θέματα, η έλλειψη αλληλεγγύης, κλείσιμο συνόρων με χαοτικό τρόπο κτλ. Αν δεν υπάρξουν συμφωνίες για το σχέδιο ανάκαμψης, τότε θα αντιμετωπίσουμε κοινωνική και οικονομική κρίση χωρίς προηγούμενο, αν δεν συμφωνήσουν οι ηγέτες των χωρών. Και δυστυχώς καθυστερεί ακόμη, κολυσιεργεί το Συμβούλιο. Από τον Γενάρη είναι έτοιμη η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Η περίπτωση του Συμβούλου διαφορετική. Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει. Θέλουν οι συμπολίτε μα μια πιο ισχυρή Ευρώπη στο μέλλον. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα εδώ ε, στη φυσαλίδα τη Ένωση. Χρειαζόμαστε όλοι να ε, βάλουμε το λιθαράκι μα. Ε, και το Κοινοβούλιο σίγουρα έχει επίγνωση των ευθυνών που τα αναλογούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για τι αλλαγέ και για μια πιο ισχυρή Ευρώπη στο πλευρό των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Φερχόφστατ εκ μέρους ε, τη ομάδα Ρενιού για δύο λεπτά. Παρακαλώ να ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ. Είναι πολύ απλό ο λόγος που έχουμε αυτό το ψήφισμα. Δεν είναι ένα ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή για τους συναδέλφου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Είναι ένα ψήφισμα που ουσιαστικά απευθύνεται στο Συμβούλιο. Και ελπίζω το Συμβούλιο αυτή τη φορά να καταφέρει να φτάσει σε μια συμφωνία ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτήν την ε, διάσκεψη. Γιατί α είμαστε ειλικρινεί. Αυτή η διάσκεψη γίνεται το τέρας του Λόχνες. Ε, δηλαδή κάποτε εμφανίζεται, μετά εξαφανίζεται είναι κάτι σαν ε, αυταπάτη, είναι κάτι σαν αντικατοπτρισμός ε, και συγγνώμη, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Δεν είναι αυτή η διάσκεψη ένα εργαλείο ψηλοασήμαντο για το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό. Είναι ζωτική σημασία σε αυτή η διάσκεψη είναι πραγματικά πολύ σημαντική, είναι κρίσιμη για το μέλλον όλων των Ευρωπαίων. Ας ε, ε, το συνειδητοποιήσουμε, γιατί το είδαμε και με την κρίση της COVID-19 που θα αλλάξει τον κόσμο. Ο κόσμος μετά την ε, COVID-19 θα είναι τελώς διαφορετικός. Δεν νομίζω ότι πλέον θα κυριαρχείται από τις ΗΠΑ που αποχωρούν από το διεθνές προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Αυτό βλέπουμε ίσως κυριαρχείται από την Κίνα ο κόσμος στο μέλλον. Η Κίνα θέλει και είναι ήδη υπερδύναμη παγκόσμια και θέλει ε, να έχει ε, την ε, κυριαρχία αυτή, τη δεσπόζουσα θέση. Και εμεί ε, που βρισκόμαστε, κάπου στη μέση, εγκλωβισμένοι. Αν δεν θέλουμε να είμαστε όμω εγκλωβισμένοι μεταξύ ΙΠΑ και Κίνα και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε στη διάθεσή μα τα εργαλεία για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των πολιτών μα, χρειαζόμαστε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνεται όμως αυτό το σκοπό αυτή η Ένωση όσοι έχει τώρα. Δεν είναι προσαρμοσμένη στο μέλλον. Συμβούλιο το ξέρει, Επιτροπή το ξέρει, Κοινοβούλιο το ξέρει, το ξέρουν και οι συμπολίτε μας. Καιρός πλέον λοιπόν είναι να δρομολογηθεί αυτό το εγχείρημα, διότι δεν είναι μας μένει πολύς χρόνος. Μήπως θα έπρεπε να το πείτε ε, στου συναδέλφους σας ε, στο Συμβουλίο. Έχουμε την ε, κρίση της COVID και αύριο μπορεί να υπάρχουν άλλες προκλήσεις. Παρακαλώ λάβετε μια απόφαση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την κοινή διακήρυξη των τριών θεσμικών οργάνων και το Σεπτέμβρη να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατό το Σεπτέμβρη να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ε, η κυρία ε, από την ομάδα ΙΝΤΕ. Αγαπητοί συναδελφοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τον προβληματισμό για το μέλλον της Ευρώπης. Διάλογος μεταξύ Ένωσης και του κόσμου. Σύμφωνα, είχαμε τη συνθήκη της ε, Ρώμης, αλλά φαίνεται τώρα ότι είναι πάρα πολύ μακριά και νομίζω ότι αυτή η κρίση είναι το κύκνιο άσμα ε, της φεντεραλιστικής Ευρώπης. Είδαμε τα προβλήματα υγειονομικά από την πανδημία και έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα για τη χαλάρωση των μέτρων. Ε, χρειάζεται μια συνένεση στο πρόγραμμα ανάκαμψης, αλλά οι αποτυχίες δεν είναι μόνο για σήμερα και μόνο από σήμερα, οπότε θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και πού θα πάμε. Ο πολιτισμός, ε, η ισχύ της Ευρώπης, οι αρχές της δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο. Ε, ο κόσμος θέλει τη χώρα του, θέλει τους ήρωές του. Ε, ο φεντερελισμός είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Άρα χρειάζεται όλοι μαζί να ξανακερδίσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Ευχαριστώ. Φρόιντ, για 1,5 λεπτό τους πρασίνους, επόμενος ομιλητής. Αγαπητοί, συνάδελφοι, έχω 1,5 λεπτό μόνο σήμερα στη διάθεσή μου. Ακριβώ αυτό το χρόνο αφιέρωσα και το Συμβούλιο για τη συζήτηση της έκβασης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με τους πολίτες. Είχαμε 1.600 διαλόγους των πολιτών. Μιλήσαμε με χιλιάδες συμπολίτες μας και πραγματικά ε, έχω σοκαριστεί με την έκβαση αυτής της διετούς ε, διαβούλευσης που ουσιαστικά κατέληξε σε μια συζήτηση και κλεισμένο το θηρό στο Συμβούλιο. Πώς θα εξηγήσουμε στους πολίτες ότι συζητούμε το μέλλον της Ευρώπης, αλλά δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα και αποκλείουμε την πιθανότητα αναθεώρηση των συνθήκων, μεταρρυθμίση των συνθήκων ευθύ εξ πριν καν την έναρξη τη συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη. Για δεύτερη φορά σε μία δεκαετία φαίνεται ότι διαλυσθάνουμε προ μία από τι χειρότερε οικονομικέ κρίσει. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι χάνουν τι δουλειέ του, κυρίω νέοι, που μόλι ορθοπόδησαν μετά την προηγούμενη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Το θέμα είναι, ε, έχουμε την πολυτέλεια να θυσιάσουμε μία ακόμη δεκαετία. Πότε επιτέλου θα αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές αδυναμίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διέλθουμε από την τρέχουσα κρίση ταχύτερα από, ό,τι, την προηγούμενη. Η διάσκεψη ε, έχει γίνει σαν φάρσα. Ε, έχουμε τονίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών δεν είναι αστείο, δεν είναι πλάκα. Ούτε οι ελάχιστε μεταρρυθμίσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αστείο, δεν είναι πλάκα. Και θα πρέπει να εξέλθουμε από, την, ε, από το εγχείρημα αυτό ισχυρότερη και πιο ενωμένη. Ας αφήσει τα αστεία λοιπόν και τις κοροϊδίες στο Συμβούλιο και ας αρχίσουμε επιτέλους να συζητούμε για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ για το ίσια Κύριος Γκρασνοντές για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Συντηρητική. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μου ομάδα επίσης πιστεύει ότι απαιτείται εις βάθος μεταρρύθμιση της Ένωσης κυρίως υπό το φως των τελευταίων εμπειριών της πανδημίας που μας έδειξε πόσο ανέτοιμοι, πόσο προετοίμαστε και πόσο δύσκολα προσαρμοζόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε απειλές στην ύπαρξή μας. Επίση, συμφωνούμε με την ιδέα τη οργάνωση διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Αρκεί αυτή η διάσκεψη να έχει πραγματικά ανοιχτό χαρακτήρα και να δώσει φωνή ακόμη και σε εκείνου που δεν τηρούν την φεντεραλιστική ορθοδοξία. Βέβαια, δεν έχω και πολλές ελπίδες, βάσιμες ελπίδες ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, επανέλθουμε σε μια ένωση ευρωπαϊκής κοινότητας κυρίαρχων ε, εθνών που θα στηρίζεται σε μια ευρωρεαλιστική άποψη συνομοσπονδιακή Ευρώπη που θα σέβεται το δικαίωμα και την ομοποίηση των κρατών μελών, θα είναι δημοκρατική για τα κράτη-μέλη. Και επίση θα πρέπει να ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε και τα πνευματικά τη θεμέλια και να μάθουμε από την ιστορία του 20ου αιώνα και πόσο επικίνδυνες είναι μερικές φορές οι απόπειρες απόλυτης ανοικοδόμησης των κοινωνιών. Η κυρία Φοντερ Λάιεν είπε ότι η ενότητα στη διαφορετικότητα είναι το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όμως, αντί για διαφορετικότητα, έχουμε όλο και μία μεγαλύτερη ομοιογεωνοποίηση της γνώμης, της κουλτούρας, της συλλογικότητας τα έθνη έχουν την αίσθηση ότι στερούνται όλο και περισσότερο το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα ίδια. Και οι πολίτες πιστεύουν ότι όλο και περισσότερο παρεμβαίνουν στη ζωή τους, περιορίζουν τα δικαιώματά τους. Στο όνομα μιας υποτίθεται ιδεολογικής απελευθέρωσης. Θα πρέπει να δώσουμε στην Ευρώπη το πραγματικό της χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Κύριο Σόλτς για λεπτό για την ομάδα Αγαπητοί Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με προλαλήσαντες. Ε, πραγματικά περιμένουμε τοποθέτηση του, του Συμβουλίου. Ε, οχτώ μήνες έχουν περάσει από τότε που η πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το υποσχέθηκε. Υποσχέθηκε στους πολίτες αυτή την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη και ήδη ξεκίνησε το Κοινοβούλιο εντατική εργασία για αυτή τη διάσκεψη. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν ε, τη θεσμική οργάνωση, ε, την συντακτική και σταματική εντολή αυτής της διάσκεψης. Αυτά δεν τα έχουμε διευκρινίσει ακόμα, αλλά μας πιέζει ο χρόνος αν θέλουμε να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν αυτή τη συζήτηση. Γιατί αλλιώ γινόμαστε πραγματικά ε, αστεί, ε, γελοί και από την χάνη η προσπάθειά μας και χάνεται η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία στην δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει το μέλλον. Ε, υπάρχουν σίγουρα ε, προβλήματα, η ευρωπαϊκή ε, κρίση του ευρώ, η κρίση της μετανάστευσης, το έλλειμμα κράτους δικαίου. Υπάρχουν δηλαδή ελλείψεις, τις είδαμε την τελευταία δεκαετία και επίσης μετά το Brexit θα αντιμετωπίσει Ένωση σίγουρα και άλλες κρίσεις. Υπάρχουν διαφορετικές σίγουρα απόψεις ό,τι αφορά το ΠΔΠ, την ΕΚΤ και την πανδημία. Όμως χρειάζεται μαζί με τους πολίτες μας ε, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις αδυναμίες ε, της δομής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενδυναμώσουμε την Ένωση μαζί με τους πολίτες. Θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία του αναστοχασμού. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να συνεργαστούμε και με τους πολίτες, να δείξουμε τι μπορούμε να πετύχουμε, τι έχουμε πετύχει και ποιοι είναι οι λόγοι για τις αδυναμίες και τις αποτυχίες. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά ελπίζω και περιμένω από το Συμβούλιο να κάνει ένα βήμα ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η διάσκεψη, κάτι το οποίο είναι απόλυτα αναγκαίο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Καστάλτο για ένα λεπτό, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροπε συναδελφοί. Αυτή η κρίση είναι κοινωνική, οικονομική από την πανδημία και έτσι απογυμνώθηκε, έτσι φάνηκε το πόσο χρειάζεται να ξανακερδίσουμε τον ε, κόσμο. Είδατε τι έγινε με αυτά τα γκάλωπ, ότι 57% από τον κόσμο δεν είναι ικανοποιημένοι από την αλληλεγγύη των ε, προς τα κράτη-μέλη κατά την κατάσταση ανάγκης. Συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση και θα πρέπει αυτή η δυσκολία να γίνει ευκαιρία, θα πρέπει άπαξ και διαπαντός να παρακάμψουμε όλα αυτά τα, τα εμπόδια, τα νομικίστικα, όπως ε, ε, τις διάφορες ρήτρε, όπως την ενισχυμένη πλειοψηφία, τόσο ώστε κάτι να κάνουμε για την υγεία, για τις ανισότητες, για να υπεραμεινθούμε όλων αυτών των δικαιωμάτων και όσων καίνε τους πολίτες και αυτό να γίνει από τη βάση ακόμα και αλλάζοντας τις συνθήκες χωρίς να φυστούμε μέσον θα πρέπει να αλλάξουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές εδώ στο Κοινοβούλιο για τις αξίες μας, για το όραμά μας και επίσης και το Συμβούλιο θα πρέπει να ξυπνήσει μη χάνεται άλλο χρόνο από το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ε, γιατί αλλιώς θα ξυπνήσουμε πολύ άσχημα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χίμπνερ τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. President... Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ με όλους σας ότι συζητούμε για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης τόσο καιρό που επιτέλους είναι και η ώρα να τις δώσουμε σάρκα και ωστά. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το καθήκον να δείξει πολιτικό θάρρος και τόλμη και μας εξέλεξαν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και εμείς πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και πόσο προσιλωμένοι και αφοσιωμένοι είναι οι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο ενδιαφέρονται να είναι ανοιχτοί στον κόσμο. Βέβαια υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των προσδοκιών ε, των ε, πολιτών από την Ευρώπη και τι πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει για αυτούς σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κενά ε, που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν οι αντιευρωπαίοι και οι λαϊκιστές. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να κήρυξουμε τα εγγένεια της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, που είναι μεγάλη ευκαιρία να έχουμε πιο νομιμοποιημένη και δημοκρατική Ευρώπη και να καταστήσουμε και πιο αποτελεσματική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι κρίμα και ντροπή η διάσκεψη να μην μας θωρακίσει στο μέλλον, να μην μας επιτρέψει να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες για να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Νομίζω ήρθε το πλοίο της, ιστορία, της ιστορίας στις ακτές μας. Δεν μπορούμε να το χάσουμε. Αυτό μου λένε οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ρουίς Ντεβέσα για ένα λεπτό είναι επόμενος. Για ένα λεπτό κύριος Ρουίς Ντεβέσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε την ευκαιρία αλλά και ταυτόχρονα το καθήκον και την υποχρέωση, αγαπητοί συνάδελφοι, να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο δημοκρατική, πιο διαφανή, πιο αποτελεσματική και πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Πριν από 20 χρόνια, θα το θυμάται ο κύριο Φερχόφστατ, με τη διακήρυξη του Λάκεν, ξεκινήσαμε το τελευταίο επίσημο εγχείρημα για το μέλλον της Ευρώπης, την επίσημη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Οι συνάδελφοι απαρίθμησαν ε, τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και η πανδημία είναι η τελευταία πρόκληση μόνο. Κυρία εκπρόσωπε του Συμβουλίου, είδατε την ξεκάθαρη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συντριπτική πλειοψηφία είναι ενωμένη. Ακόμη και ο κύριος Καστάλντο από τους μη μας στηρίζει. Τι περιμένουν λοιπόν οι κύριοι του Συμβουλίου, τι περιμένετε. Η θέση μας είναι διαμορφωμένη ήδη από τον Ιανουάριο. Έχει περάσει ένα εξάμενο. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο είναι πιο αργό ε, θέλει χρόνο. Αλλά επιτέλους θα πρέπει να διαμορφώσει και το Συμβούλιο τη θέση του και το Σεπτέμβριο να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε αυτή τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Χωρίς αποκλεισμού, όπως είπε και η κυρία Χιούμπνερ. Και ίσως θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε και στη συζήτηση και το θέμα της μεταρρύθμισης των συνθήκων. Ευχαριστώ. Επόμενο είναι ο κύριο ε, Γκούναρ Μπέκα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στο Στρασβούργο είχα μιλήσει για τον ε, Ζίγμουντ Φρόιντ και την ε, φυγή των ευρωσικών προ την νόσο, διότι η νόσο απελευθερώνει από την ταλαιπωρία τη ίαση και ουσιαστικά επαγγέλλεται την διακοπή από την πραγματικότητα. Τι προφητικά λόγια ήταν αυτά, διότι βλέπουμε τώρα με την κρίση του κορονοϊού μια τελευταία πιο πρόσφατη ψαναρρύθμιτε κρίση Ευρωπαϊκή Ένωση, για τι οποίε είμαστε μόνοι μα υπέτη και τώρα πάλι κλαίγονται οι πολιτικοί και δεν ξέρουν πώ θα προχωρήσουν. Το μόνο που ξέρουν ότι χρειάζονται περισσότερη Ευρώπη και το προσκήνιο, η ε, σκηνή τώρα είναι αυτή η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αποτελεσματική, δημοκρατική, κοντά στον πολίτη, αλλά τελικά αυτό το οποίο προβλέπεται δεν είναι οι αποφάσει ε, που θα λαμβάνονται από του πολίτε, αλλά ένα ε, δομημένος διάλογο των πολιτών που όμω θα είναι υπό την καθοδήγηση των φιλοευρωπαϊκών ε, ΜΚΟ και της Ένωσης. Ε, και τελικά πρόκειται ε, για μεγαλύτερο χρέος, για πατρονάρισμα και για ανακατανομή των ε, του πλούτου. Το αποτέλεσμα τελικά δεν είναι δηλαδή η ίαση, αλλά το αντίθετο. Είναι μια φυγή προ τα κάτω, γι' αυτό η Γερμανία και η Ένωση χρειάζονται να καθίσουν, να ξαπλώσουν στο διβάνι του. Ευχαριστώ, just... Πρόεδρε. Μισό αυτό να βγάλω τη μάσκα μου. Θέλω να πω στον κύριο Μπέκο, δεν θα διαβάσατε το σημείωμα. Όχι, δεν είναι ενορχιστρωμένοι οι διάλογοι με του πολίτε, Είναι διάλογο των πολιτών. Τίποτα δεν ενορχιστρώνουμε και ούτε θέλουμε και είπαμε ξεκάθαρα στο Συμβούλιο ότι αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Δεν μπορεί να αποφασίσει το Συμβούλιο. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε με του πολίτε γιατί πρόκειται για το μέλλον. Κανεί δεν είχε προγνωστικά για την πανδημία, αλλά είδατε ποιο ήταν ο αντίκτυπο και πώ δουλεύουμε και εμεί τώρα στι οικογένειε. Γιατί να μην τα συζητήσουμε ανοιχτά. Και ε, Όλο λέει το συντομότερο δυνατόν το Συμβούλιο. Όχι, δεν υπάρχει συντομότερο. Εγώ λέω τώρα, όχι σε ένα χρόνο, τώρα, σήμερα. Οπότε ακούστε τι πρεσβεύουμε όλοι, όλοι αυτό από έναν δύο. Θέλουμε να κάνουμε βήματα προ τα εμπρό. καθίστε με το Κοινοβούλιο, τα ε, Εθνικά Κοινοβούλια, με του πολίτε για μια καλύτερη Ευρώπη. Δεν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, θέλουμε καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπίσοφ, έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ακούσατε, έχουμε εδώ ένα κοινοβούλιο το οποίο εκπλήσεται και διαρωτάτε γιατί ένα μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να κάνει καν το πρώτο βήμα. Δεν μπορεί να αποφασίσει εδώ δεν μιλάμε για αλλαγή της ε, συνθήκης, δεν είναι πολύπλοκη εντολή. Πρέπει απλά να συμφωνήσουμε, θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ε, για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η διάσκεψη. Και ούτε αυτό δεν γίνεται από το Συμβούλιο. Εξού και χρησιμοποιούμε αυτή την ολομέλεια για να στείλουμε ε, ένα σαφές μήνυμα. Έξι μήνες μέχρι τον Ιούνιο, από, τον Γενάριο, από τον Ιανουάριο ψάχνουμε πλέον αυτή την εντολή. Γιατί δεν προχωράει το Συμβούλιο γιατί υπάρχει αυτή, αυτό το αδιέξοδο. Ε, πώς θα προχωρήσουμε αν δεν μπορούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Αν δεν μπορεί το Συμβούλιο να κάνει το πρώτο βήμα. Δεν θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε έτσι σταθεροποίηση της Ευρώπης. Ε, το ακούσατε και το επαναλαμβάνουμε δεν επιτρέπουμε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια ακόμη αποτυχία. Δεν ε, θέλουμε ε, να παραμένει σε ακινησία το Συμβούλιο και γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση και στη Γερμανική Πρόεδρε που θα αναλάβει από τον Ιούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Κόφτ για ένα λεπτό. Um Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα είναι απλώς μία από τα ίδια περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερες δαπάνες. Ε, τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Ε, πριν έρθω στο κοινοβούλιο ε, ήμουν επιφυλακτικός, τώρα είμαι κατά, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα τι θα γίνει, το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να αδειάζουμε τις τσέπες μας και να δίνουμε επιδόματα, τέρμα η γραφειοκρατία, τέρματα τα ανοιχτά σύνορα της Ευρώπης. Δεν θέλω να μας δυναμητίζει την αγορά εργασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινωνικές μας πολιτικές. Θέλω πίσω τη χώρα μου, τη Δανία. Με πείσατε αυτό το σύστημα δεν μπορεί ούτε να βελτιωθεί ούτε να διασωθεί. είναι καταδικασμένο για το χροντούλο από της ιστορίας. Οπότε θέλω η Δανία να φύγει από την Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία του Πρόεδρου Σουίτσα έχει το λόγο ακόμη μια φορά και μέρος της Κομισιόν. President. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θερμά ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να συζητήσουμε και πάλι τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Τα σχόλιά σας είναι πολύ σημαντικά και τροφοδούν την περαιτέρω συζήτηση. Εκτιμώ ιδιαίτερω ε, τις απόψεις σας, την συμμετοχή σας και την επιθυμία σας να δώσετε σάρκα και οστά στην διάσκεψη αυτή για το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όταν υιοθετήθηκε στις 22 Ιανουαρίου ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση της διάσκεψης Ήμασταν ήδη στην 7η ε, χρονιά ανάκαμψης και μάλιστα οι προβλέψεις έδινα, έδειχναν ε, περαιτέρω μεγέθυνση για την επόμενη περίοδο. Και τώρα αργά εκατομμύρια πολίτε βγαίνουν σιγά σιγά από τα περιοριστικά μέτρα και οι προπτικές έχουν αλλάξει ριζικά. Παρ' όλα αυτά, η αποφασιστικότητά μας να συνομιλήσουμε με τους πολίτες και να τους αφουγκραστούμε και να εισακούσουμε την φωνή τους, αυτό δεν έχει αλλάξει. Και το βασικό μήνυμα σήμερα είναι ότι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης έχει κρίσιμη σημασία. Θα έλεγα μάλιστα ότι ακριβώς λόγω της πανδημίας είναι ακόμη πιο σημαντικό σπουδαιότερο από ποτέ να έχουν περισσότερο λόγο οι Ευρωπαίοι πολίτες στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι λειτουργεί σε αυτή. Θα πρέπει να απαντήσουμε σε δύσκολα ερωτήματα και έτσι θα σώσουμε ζωές. Θα ήθελα να τονίσω ότι θέλουμε η διάσκεψη να είναι ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανής και να έχει μια συγκροτημένη, διαρθρωμένη συζήτηση. Και όπως λέμε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διάσκεψη, οι αρχές ε, που προδιαγράψαμε εκεί ισχύουν. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι πολίτης θεωρεί σημαντικό. Ε, θα έχουμε φυσικά και πολιτικές προτεραιότητες και το στρατηγικό θεματολόγιο του Συμβουλίου που δίνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είχαμε ήδη πολυάριθμους διαλόγους με τους Ευρωπαίους πολίτες και θεωρώ ότι θέματα όπως ε, η υγεία και η αντιμετώπιση της ε, υγειονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία τώρα. Οπότε, παρά τις δύσκολες συνθήκες, θα, θα θέλαμε το συντομότερο δυνατό Ακόμη και τώρα, αν γίνεται, να εγκαινιάσουμε τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Και από τη στιγμή που θα καθορίσει το Συμβούλιο την εντολή του, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή διακήρυξη. Και έχουμε δεσμευθεί να εφαρμόσουμε ό,τι θα αποφασιστεί στη διάσκεψη. Γιατί αυτό θα είναι το μέτρο τη επιτυχία μα. Της επιτυχίας μας και είμαι προσιλωμένη σε αυτό. Πριν την πανδημία, ε, είχα προγραμματίσει να επισκεφτώ και τις 27 χώρες μέλη. Τελικά πρόλαβα μέσα σε ένα εξάμεινο μόνο 10 να επισκεφτώ και στην εντολή και την αποστολή μου επικεντρώθηκα σε τοπικά και περιφερειακά παραδείγματα, γιατί εκεί συμμετέχουν διαρθρωτικά οι πολίτες στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Γιατί θα πρέπει να έχουμε feedback από τους πολίτες. Αυτό θα έχει κέρια σημασία στην επιτυχία της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει να έχουμε συνεχώς τροφοδοσία από τους πολίτες σε αντίθεση με τις προηγούμενες διαβουλεύσεις. Επίσης, οι ιδέες που θα προκύψουν σε τοπικές συζητήσεις θα πρέπει να συζητηθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όπως ε, είπαν και οι ευρωβουλευτές σήμερα, Επιμένω η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης να είναι αντιπροσωπευτική και από γεωγραφική άποψη, από άποψη φύλου, ε, ηλικίας, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και μορφωτικού επίπεδου των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και μειονοτικούς πληθυσμούς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Όπω είπα και προηγουμένω, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να προκαθορίσουμε ή να προδικάσουμε την έκβαση, το αποτέλεσμα τη διάσκεψη. Αυτό το είχαμε συμφωνήσει ήδη από την αρχή. Δεν θα πρέπει να προεξοφλούμε το αποτέλεσμα τη διάσκεψη, ούτε να περιορίσουμε τα θέματα προ συζήτηση είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μας. Έχουμε το, τη δυνατότητα να χαράξουμε το δρόμο για νέου είδους πολιτικής, για μια νέα δυναμική, για να συμπληρώσουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και μόνο από κοινού μπορούμε να το επιτύχουμε. Μπορούμε να ενισχύσουμε από κοινού τη, το δεσμό μεταξύ της δια, διαδικασίας λήψης αποφάσεων και πολιτικών και της αυξανόμενης ε, εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η αύξηση της εμπιστοσύνης αυξάνει και την νομιμοποίηση. Α συνεργαστούμε λοιπόν για να κάνουμε τη διάσκεψη τη Ευρώπη πραγματική επιτυχία για του Ευρωπαίου πολίτε. Και περιμένω με αδειμονία την απόφαση του Συμβουλίου επί τη κοινή διακήρυξη. Ελπίζω ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι και θα καταφέρουμε να κηρύξουμε την έναρξη της διάσκεψης. Σας ευχαριστώ και τώρα ο λόγος ε, στην Υπουργό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα κατακλείδη να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη χρήσιμη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις απόψεις για το σημαντικό αυτό θέμα και τις σημείωσα λεπτομεριακά. Η Προεδρία είναι πλήρως προσιλωμένη στην αναζήτηση λύσης και απόφαση του Συμβουλίου. Και εγώ προσωπικά λυπούμε ειλικρινά που δεν καταφέραμε στο Συμβούλιο ε, να ε, καταλήξουμε σε απόφαση και να κηρύξουμε την έναρξη τη διάσκεψη κατά τη διάρκεια τη Κροατική Προεδρία και από την έναρξη τη πανδημία, δεν εφίστημα προσπαθειών για να διευκολύνουμε τη συμφωνία στο Συμβούλιο και συνεχίζουμε τι προσπάθειέ μα. Θα ήθελα να σα καθησυχάσω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με φιλοδοξία και πυγμή προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι ένα νέο σχέδιο αυτή η διάσκεψη και μάλιστα μερικοί εμπλεκόμενοι φορείς έχουν μεγάλες φιλοδοξίε από το εγχείρημα αυτό. Αναμένεται ε, τα κράτη-μέλη να την προσεγγίσουν με διαφορετικές ιδέες, εμπειρίε εμπειρίες και προτεραιότητες. Πάντως το ζητούμενο είναι η συνένεση και μια και είναι μια πολύ σημαντική και συναισθηματικά φορτισμένη συζήτηση για την Προεδρία και αυτή θα είναι και η τελευταία μου ολομέλεια ως εκπροσώπου της Προεδρίας, θα ήθελα να πω και λίγα λόγια στη μητρική μου γλώσσα, τα κροατικά. Κατά την πρώτη Κροατική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίσαμε μια πρωτοφανή στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκληση. Είμαι υπερήφανη για την άμεση κοινή μας αντίδραση ε, χάρη στην προσήλωση όλων των συναδέλφων και είμαι υπερήφανη που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την ε, συνέχιση των, ε, της λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο και να έχουμε και συνεχή επικοινωνία με τους υπουργού στα διάφορα υπουργικά συμβούλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ευρωβουλευτές άνδρες και γυναίκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέχισαν την στενή συνεργασία με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή στο απόγειο της κρίσης και έτσι καταφέραμε να εθετήσουμε τις πρώτες τη δέσμη μέτρων για να αντιμετωπίσουμε ε, τα προβλήματα για την ευρωπαϊκή υγεία, την οικονομία, την κοινωνία που δημιούργησε η πανδημία COVID-19. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με επιτυχία και για το σχέδιο ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που υποστηρίξατε ενθουσιοδό το κροατικό πρόγραμμα και τι προτεραιότητε τη κροατική Προεδρία. Ήταν ανεκτήμητη η συνεργασία σα στο τελευταίο αυτό εξάμεινο. Επίση, θα ήθελα να εκφράσω την ακράδαντη πεποίθηση ότι πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη του μήνα θα καταλήξουμε στην άποψη του Συμβουλίου για τη θέση του ως προς τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Μια υγιής, ανθεκτική, υπεύθυνη, ισχυρή και ασφαλής Ευρώπη στα μέτρα των πολιτών μας θα πρέπει να αποτελέσει την πρωταρχική μας προτεραιότητα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην συνέχεια ε, προς όφελος και προς την, για χάρη της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα που εκπροσώπησα την Κροατική Προεδρία σε αυτή την πρώτη φορά που η Κροατία ανέλαβε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ σίγουρα. Ε, κάνατε πάρα πολλέ προσπάθειες αυτό το εξάμεινο και θέλω να σα ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία. Εδώ ολοκληρώθηκε λοιπόν σήμερα θα ε, ολοκληρωθεί η προθεσμία την κατάσταση απολογιών και αύριο θα ψηφίσουμε. Έχω να σας ε, κάνω και μια ανακοίνωση ότι αφορά ε, τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας. Θα τα ακούσει στις 8 και 8 και 4 και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της διάταξη, διάταξης που είναι οι δηλώσει της επιτροπή και του Συμβουλίου για την προστασία ευρωπαϊκών στρατηγικών κλάδων από εξαγορές μετά τον COVID, την κρίση COVID. Δεν μπορείτε να ζητήσετε το λόγο φορμήτως ούτε θα γίνει χρήση μπλε καρτών. Περιμένουμε να γίνει απολύμανση και να, ε, λάβουν, αλλάξουν σκητάλι οι ομιλητές μας όταν όλοι θα έχουν ε, καθίσει στις θέσεις τους. να ξαναδώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της κρατικής προεδρίας. Thank you again. President, honorable member. Και πάλι ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Τα μέλη του Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου σε κοινή δήλωση τόνισαν ότι η πανδημία είναι ένα πρόβλημα χωρίς προηγούμενο, μια πρόκληση για Ευρώπη για όλο τον κόσμο, οπότε χρειάζεται αποφασιστική δράση σε κάθε επίπεδο, ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό και δεσμευτήκαμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται να προστατεύσουμε τον κόσμο και να βρούμε τη διέξοδο από την ε, κρίση ε, και να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και επίσης το Συμβούλιο θεώρησε πάρα πολύ θετικά τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτές τις επενδύσεις από το εξωτερικό. Να προστατεύσουμε του στρατηγικούς μας κλάδους, την τεχνολογία από τέτοιες επενδύσεις που μπορεί να αντιβαίνουν στους στόχους μας και οι ηγέτες. Είπαν ότι έτσι ε, συμβάλλουμε στην στρατηγική αυτονομία της Ένωσης κατά την κρίση και μετά και είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να βγει από την κρίση κλείνοντας τις πόρτες στο διεθνές συμπόριο και επενδύσεις. Πάρα πολλέ ευρωπαϊκές εταιρείε ανήκουν στην παγκόσμια ε, αλυσίδα ε, προσφοράς και ε, επίσης γι' αυτό και υπάρχουν όλες αυτές οι επενδύσει, το διεθνέ εμπόριο, πολύ σημαντικό την ανάκαμψη τη οικονομία μα. Οπότε θα πρέπει εμεί να έχουμε μια ποικιλία σε αυτέ τι αλυσίδε προσφορά και θα πρέπει να έχουμε ε, βελτίωση των υπηρεσιών μα, να προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση. Αλλά επίση θα πρέπει να επαγρυπνήσουμε, να εξασφαλιστεί ότι θα προστατεύσουμε του ε, τομεί μα που είναι σημαντικοί για την ε, ασφάλεια και είναι η σημαντική στήλη τη οικονομία σε αυτό άμεσα έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα ανακάμψουμε. Η οικονομική κρίση που είναι απόρρια της πανδημίας έχει αδυνατήσει πάρα πολλές εταιρείε. Ε, πέσανε οι μετοχές τους και υπάρχει ο κίνδυνος των εξαγρών από αλλοδαπές εταιρείε ιδίως από τις χώρες ε, όπου οι επενδυτές βοηθούνται από το κράτος. Οπότε θα πρέπει να ξεσορροπήσουμε τις επενδύσεις ε, να τις παρακολουθήσουν με τα κατάλληλα εργαλεία, να υπάρχει ένα πλαίσιο αυτό που ήδη έχουμε για την προστασία αυτών των θεμητών μας ε, συμφέροντων. Οπότε θα πρέπει οι αρμόδιοι για την εσωτερική αγορά, οι υπουργοί να τα συζητούν ε, και τα συζητούν σε τακτά διαστήματα όσον αφορά το τι γίνεται με την αγορά και με την βιομηχανία για το πώς θα ενδυναμώσουμε στρατηγικά και οικονομικά τους σχετικούς κλάδους, την αλυσίδα αξιών και επίσης να υπάρξει προστασία από αυτές τις αλλοδαπές Εξάγορε. Θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ θετική η νέα βιομηχανική πολιτική της Κομισιόν. Παρουσιάστηκε τον Μάρτιο. Είμαστε υπέρ των δράσεων που εξήγηλε η Κομισιόν για τις ψηφιακές ε, υποδομές, συνέργεια. Ε, επίσης να δούμε τι θα γίνει με την βιομηχανία, την αμυντική, τη φαρμακοβιομηχανία ε, να δούμε πώς θα έχουμε περισσότερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Και αυτά μόνο ενδεικτικά τα αναφέρουμε και την Παρασκευή κάναμε μία τηλεσυνεδρίαση ε, και οι αρμόδιοι υπουργοί για την εσωτερική αγορά επίση συζήτησαν την ανακοίνωση τη Κομισιόν για τη δέσμη μέτρων τη 27η Μαου για την ανάκαμψη. Επίση, θεωρήσαν θετικά τα μέτρα τη Επιτροπή, ούτω ώστε να υπάρχει περισσότερη ανθεκτικότητα, στρατηγική αυτονομία με στρατηγικέ τεχνολογίε και αλυσίδε αξιών και ε, έτσι βέβαια να ισχύουν και αρχέ τη ανοιχτή αγορά, τη ελεύθερη αγορά. Έχουμε το Invest EU, ε, έτσι θα έχουν περισσότερη ανθεκτικότητα και καλύτερες ε, επενδύσεις ε, στην βιομηχανία και αυτό θα έχει σχέση και με την μετάβαση την ψηφιακή και την περιβαλλοντική. Λάβαμε υπόψη το θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των ε, επενδύσεων. Έτσι θα προστατεύσουμε ε, την, την περιουσία μας, της στρατηγικούς τομείς. Οπότε να μπορούμε να αποκρούσουμε τις επιθετικές, απειλητικές ε, εξαγορές στο εξωτερικό. Αυτό ήδη στο παρελθόν αυτό το μέσον του screening, αυτό του ελέγχου των επενδύσεων και εξαγορών υπήρχε και όλα αυτά οι συνομοθέτες τα βλέπουν με ενιαία άποψη. Τώρα είμαστε ικανοί περισσότερο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα έρθουν. Και όλο ένα και περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ένα τέτοιο μηχανισμό ελέγχου των επενδύσεων και πολλά άλλα κράτη επιταχύνουν το πώς θα υπάρχουν σημεία επαφής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ανταλλαγή με την Κομισιόν για τέτοιες ε, εξαγορές, γιατί αλλιώς απειλείται η ασφαλειά μας, όλο ένα και περισσότερο. Οπότε η Κομισιόν τα αναλύει, αναλύει τις τάσεις. Έχει μια ομάδα από εμπειρογνώμονες, υπάρχει σχετικός κανονισμός και υπάρχει και η λευκή βίβλος όσον αφορά τις ξένες ενισχύσεις, επιδοτήσεις, ούτως ώστε να ξέρουμε τι γίνεται με αυτές τις κρατικές επιδοτήσεις που θίγουν τον θεμητό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Σας είπα κάποια παραδείγματα και βλέπετε ότι έχει βελτιωθεί η θεσμική συνεργασία. Και αυτό προς στον των εταιριών μας και παραλαμβάνω ότι Συμβούλιο και κράτη-μέλη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, να προστατεύσουν τους στρατηγικούς μας ε, τομείς και εταιρείε, ούτω ώστε να μπορούμε να πετύχουμε τους ε, στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Πριν ε, προχωρήσουμε θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν στο τηλέφωνο να βγουν από την αίθουσα λόγω της ακουστικής που έχει η αίθουσα. Ο θόρυβος είναι πάρα πολύ ενοχλητικός. Να δώσω τώρα το λόγο στην αντιπρόεδρο κυρία Φεστάγκη, αντιπρόεδρο τη Κομισιόν. Ναι, σας ευχαριστώ κιόλας γιατί πραγματικά ήταν κάτι το οποίο μας ε, ε, αποσπίσε την προσοχή. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ επικυρή αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προστασία των ευρωπαϊκών στρατηγικών κλάδων, δηλαδή από ξένες εξαγορές στη μετά τον κορονοϊό εποχή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο και το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ίσως να είναι και το πλέον δύσκολο που είχαμε να ε, βιώσουμε ε, τον τελευταίο καιρό. αντιμετωπίζουν προκλήσεις ε, οι αγορές και η παγκοσμιαμπορική τάξη. Παρουσιάζουμε λοιπόν αυτή τη λευκή βιβλό για να ξεκινήσουν δημόσιες διαβουλεύσεις. Ιδέες για τους μελλοντικούς κανόνες ξένες ε, επενδύσεις στο μέλλον δεν θα υπονομεύσουν το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκές αγορές. αυτή τη στιγμή ξεκινούμε την ανοικοδόμηση ε, της ζημιάς που έχει προκληθεί από την COVID-19. Χρειαζόμαστε επενδύσει. Ξένε επενδύσει σίγουρα είναι σημαντική πηγή θέσεων εργασία και απασχόλησης. Είναι κάτι καλοδεχούμενο, ευπρόσδεκτο στην Ευρώπη. Οι ξένε κυβερνήσει όμω επιδοτούν ε, και στηρίζουν επενδύσει και ε, συναλλαγέ ε, στην ιστορική αγορά που μπορεί να επηρεάσει το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού με διάφορου τρόπου. Να σα δώσω μερικά παραδείγματα. Αν επιδοτούνται επιχειρήσεις που είναι στην Ευρώπη, αν βοηθούνται ε, κάποιες επιχειρήσεις με επιδοτήσεις να εξαγοράσουν ευρωπαϊκές ή ε, σε δημόσιους διαγωνισμούς ε, κάποιες επιδοτούμενες επιχειρήσεις μπορούν να, να αποκτήσουν προβάδισμα ε, σε άλλες, ε, από άλλες επιχειρήσεις και τα λοιπά. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχάς έχουμε ένα μέσο ελέγχου της αγοράς για να μπορούμε να δούμε όλες τις περιπτώσεις όπου θα είχαμε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς από τις ξένες επενδύσεις, ε, κοινή συναρμοδιότητα δηλαδή με το κράτο μέλος και την Επιτροπή και αν μια επένδυση φανεί ότι επηρεάζει πράγματα και στρεβλώνει την εσωτερική αγορά μπορούν να ληφθούν μέτρα. Αλλά αν είναι θετικό το ε, μέτρο και δεν οδεί σε στρέβλωση του ε, ανταγωνισμού, δεν θα, ε, το, δεν θα λαμβάνει μέτρα η Κομισιόν. Δηλαδή θα ελέγχουμε ακριβώς ποιο είναι το συμφέρον και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Επίσης θα έχουμε το ρόλο της Κομισιόνας εποπτική αρχής για κάποιες συναλλαγές. Θα πρέπει να κάνει την αναθεώρηση κάθε συναλλαγής και μετά θα κλείνει και θα επιτρέπει την εξαγορά θα έχουμε ακριβώς το λεγόμενο interest test, τον έλεγχο των ε, συμφερόντων και σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να υπάρξουν κάποια ζητήματα που προκύπτουν στις ε, δημόσιους διαγωνισμούς και θα πρέπει ε, οι προσφέροντες να δίνουν πληροφορίες, θα εκτιμώνται αυτές από τις αρμόδιες αρχές για να δουν κατά πόσο υπάρχει κάποια ξένη επένδυση που καθιστά θέμητη την όλη διαδικασία και τότε προσφέρον θα αποκλείεται από τη συγκεκριμένη από το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Επίσης, ε, προτείνουμε πρόσβαση σε ενωσιακή χρηματοδότηση, να δούμε αν υπάρχει εφαρμογή από τα κρατημέλη ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα. Σίγουρα όλα αυτά που λέω είναι πολύπλοκα πράγματα, γι' αυτό ξεκινάμε αυτή τη δημόσια διαβούλευση για 14 ε, εβδομάδες μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε ε, να έχουμε πολλές συμμετοχές, να λάβουμε πολλές ε, απόψεις, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, πολύ καλά ε, αυτή την διαβούλευση ερχόμενη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας παρουσιάσουμε αυτά τα θέματα και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου, τον Φιλ Χόγκαν. Έχετε το λόγο κύριε Χόγκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και η εκτελεστική αντιπρόεδρος η κυρία Βερστάγκερ, ε, η συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ επίκαιρη. Ε, ε, αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα και μια παγκόσμια υγειονομική πρόκληση που έχει σοβαρές συνέπειες και στην οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Και η έκτακτη ανάγκη του COVID ανέδειξε τα τρωτά μας σημεία. Και επίση ανθεκτικότητα των στρατηγικών μα επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στι ζωτικέ ανάγκε των συμπολιτών και οι επενδύσει ε, φυσικά θα παίξουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη των κρατών μελών. Και οι άμεσε ξένε επενδύσει ε, θα συμβάλλουν στο να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ των, ε, των τωρινών μας οικονομικών και των μελλοντικών μας προτεραιοτήτων, όπω είναι οι περιβαλλοντικέ και οι ψηφιακέ προκλήσει. Και σίγουρα θα ενισχύσουν και την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Γιατί η Γερμανία και η Ισπανία έχουν περισσότερες τέτοιε επενδύσει, μεταξύ 30 και 50% στην, Πολωνία, στην Πορτογαλία και στη Σουηδία και πάνω από 50% Βέλγιο, Αυστρία και Ιρλανδία ε, είναι οι εξωτερικές, οι ξένες μου συγγνώμη, επενδύσεις. Βέβαια αυτέ οι ξένες επενδύσεις δεν θα πρέπει να θίγουν την εθνική μας ασφάλεια και γι' αυτό και ο σχετικός κανονισμός για την παρακολούθηση αυτών των επενδύσεων ε, θα ε, συμβάλλει στην ε, αναγνώριση των προβλημάτων που ίσως δημιουργούν στην ασφάλεια αυτές οι ξένες επενδύσεις. Και μάλιστα στα τέλη Μαρτίου, όπως είπε και η Προεδρία, έχουμε, εκδώσαμε ειδικέ κατευθυντήρες γραμμές προς τα κράτη-μέλη για την προάσπιση των ε, στρατηγικών μας περιουσιακών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον κανονισμό για το screening. Φυσικά λόγω της μεγάλης εξάρτησης της οικονομίας ε, χρειάστηκε να ζητήσουν ε, συμβουλές στα κράτη-μέλη για το πού μπορεί οι εξωτερικές επενδύσεις να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην ασφάλεια. Και τα κράτη-μέλη που έχουν τέτοιους μηχανισμούς ήδη ελέγχου θα πρέπει να τους αξιοποιήσουν και να τους χρησιμοποιήσουν. Και τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη τέτοιους μηχανισμούς θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να τους θεσπίσουν. Η Ευρώπη έχει ένα αυστηρό και μοναδικό σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Υπάρχει όμως αυξανόμενη ανησυχία ότι κάποιες τρίτες χώρες ε, δεν διστάζουν ε, να βεβαίνουν σε αγορές με τεράστιες κρατικές ενισχύσεις. Και φυσικά κάτι τέτοιο θα διαστρέβλωνε την εσωτερική ε, ενιαία αγορά. Οπότε οι επενδυτές που λαμβάνουν κάποιες κρατικές ενισχύσεις θα μπορούσαν να προσβλέπουν σε εξαγορά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραγωνίζοντας ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις. Όπως είπε η κυρία Φερστάγκερ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σήμερα μια λευκή βίβλο ε, ξεκινώντας τεράστιες δημόσιες διαβουλεύσεις, ώστε οι επιδοτήσεις στο μέλλον να μην ε, αλλοιώνουν και να μην στρεβλώνουν τον ίσο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένω με ανυπομονησία τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και κυρία Επίτροπε για τις αγωγές αυτές της παρατήρησης πριν να προχωρήσουμε με τη συζήτηση και δώσω το λόγο στον κύριο Χάνσεν θα ήθελα να σας δώσω τα αποτελέσματα τον πρώτου γύρου ψηφοφορίας και ζητώ συγγνώμη που διακόπτω. Η δεύτερη ψηφοφορία ε, αρχίζει αυτή τη στιγμή επίσης. Τα αποτελέσματα λοιπόν της πρώτης ε, ψηφοφορίας, του πρώτου γύρου, είναι στις οθόνες σας τα βλέπετε σε ό,τι αφορά την άρση ε, ασύλειας του κυρίου Μπέκ εγκρίνεται η τροπολογία σε ό,τι αφορά ε, την άρση ασύλειας του κυρίου Φερχόφστατ ε, εγκρίνεται η τροπολογία σε ό,τι αφορά ε, τις για τις, το Ισραήλ απορρίπτονται για τα κατεμπήγοντα σε ό,τι αφορά την τεχνική συνεργασία και τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας εγκρίνονται για την ειδική υποστήριξη της ΕΛΑ μετά την ε, κρίση του κορονοϊού και εδώ εγκρίνονται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επίσης. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, Μεγάλη Βρετανία και Βόρειο Ιρλανδία, η 1 απορρίπτεται, η 20 απορρίπτεται, παράγραφος 4, παράγραφος ε, πρώτο τμήμα εγκρίνεται, Παράγραφος 4, δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 8, σημείο 2 ή εγκρίνεται. Οι 2 απορρίπτεται, 25 εγκρίνεται, 27 εγκρίνεται, 21 απορρίπτεται, 22 απορρίπτεται, 23 απορρίπτεται, 24 απορρίπτεται, η 3 απορρίπτεται, η 12 απορρίπτεται, η 14 απορρίπτεται, 15 απορρίπτεται, παράγραφο 41 πρώτο τμήμα δεκτό, 41 παράγραφος δεύτερο τμήμα δεκτό, παράγραφο 45 τμήμα 1 εγκρίνεται, παράγραφο 45 τμήμα δεύτερο απορρίπτεται. Τροπολογία 16 εγκρίνεται, 17 απορρίπτεται, 18 απορρίπτεται, παράγραφος δεκτή, παράγραφος 91 πρώτο τμήμα εγκρίνεται, παράγραφος 99 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται, παράγραφος 133. τροπολογία εγκρίνεται, 148 παράγραφος τέταρτο τμήμα απορρίπτεται, το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται, η 5 απορρίπτεται, η 6 απορρίπτεται, στην 153 d απορρίπτεται, ε, 156 8 απορρίπτεται, 158 9D απορρίπτεται, 10 τροπολογία απορρίπτεται, το 159 ε, το 11D απορρίπτεται, το recital ε, ε δεκτό, το 19 ε, ε, η τροπολογία 19 στο F απορρίπτεται 27 εγκρίνεται στο Result J Σε ό,τι αφορά στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άτομα με αναπηρία έχουμε τα εξαποτελέσματα 1 ε, του 3 γίνεται δεκτό 2 του 3 δεκτό 1 του 5 δεκτό 2 του 5 δεκτό. Η τροπολογία 2 απορρίπτεται. Παράγραφος 8, το πρώτο τμήμα εγκρίνεται, όπως και το δεύτερο τμήμα. Στην τροπολογία 3, εδώ είχαμε αρνητικό αποτέλεσμα. Στην παράγραφο 16, το πρώτο τμήμα γίνεται δεκτό, το δεύτερο δεκτό και το τρίτο δεκτό. Μετά την παράγραφο 21, τροπολογία 4 απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 29 το 6 εγκρίνεται. Παράγραφος 32 ε, πρώτο τμήμα δεκτό, δεύτερο τμήμα της 32 δεκτό. Παράγραφος 34 γίνεται δεκτή, παράγραφος 36 πρώτο τμήμα δεκτό, παράγραφος 36 δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Παράγραφος 38 γίνεται δεκτή, παράγραφος 46 πρώτο τμήμα δεκτό, Παράγραφος 46, δεύτερο τμήμα, δεκτό. Παράγραφος 46, ε, το τρίτο τμήμα δεκτό, 53-1 δεκτό, 53-2 δεκτό. Παράγραφος 60 δεκτή, η παράγραφος 63, πρώτο τμήμα δεκτό, το δεύτερο δεκτό μετά το recital α έχουμε τροπολογία 1 που απορρίπτεται, το G δεκτό, το L απορρίπτεται, το P δεκτό, το U γίνεται δεκτό το πρώτο τμήμα, γίνεται δεκτό και το δεύτερο τμήμα και μετά το Y έχουμε τροπολογία 5 που γίνεται δεκτή. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ψηφοφοριών και πριν ξεκινήσουμε ε, μάλλον όπως είπα ανακήρυξα και, κήρυξα και την έναρξη του δεύτερου γύρου ψηφοφορίας και τώρα δίνω το στο στον κύριο ε, Χάνσεν ε, ζητώντας του συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αγαπητοί κύριε Υπουργέ, συναδελφοί, η Κίνα δεν είναι ο μόνος ε, που προξενεί το πρόβλημα. Απλώς είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν αναφέρει κανένας. Να, τι θα πει ε, ρεαλισμός. Είδατε τι κάνει ο Τραμπ, ο οποίος είναι τάβρος ενιαλοπολείο και όλες αυτές οι κρατικές ενισχύσεις ε, έχουν πολλές εναλλακτικέ, αλλά έχουν σημασία οι πράξεις και όχι τα λόγια. Ε, Είδατε, έχουμε γεμίσει με προϊόντα ε, τα οποία πουλούνται σε όλο τον κόσμο, φτιάχνονται στην ε, Κίνα ε, και οπότε θα πρέπει ενιαία να αντιμετωπίσουμε την Κίνα, να ακουστεί η φωνή μας. Θα πρέπει αυτό το μέσο ελέγχων να αναβαθμιστεί και επίσης να προωθηθεί η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Έτσι θα πρέπει να είναι η εμπορική μας πολιτική και να έχουμε και δίκαιο αν θεμητό ανταγωνισμό. Ανιές Γιονγκέριος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όχι, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η πανδημία για να κερδίζουν κάποιοι από τις εταιρείες που έχουν χτυπηθεί. Δεν θα πρέπει να είμαστε στο έλεος των ξένων επενδυτών και εταιριών. Είδατε τι γίνεται σε πολλές χώρες. Ε, αναθεωρούνται οι νόμοι ακριβώς για αυτό το πρόβλημα. Άρα χρειάζεται να δοθεί ένας ορισμός του τι είναι στρατηγική εταιρεία. Είναι μόνο οι φαρμακοβιομηχανίες ή πρέπει να προστατεύσουμε και άλλους κλάδους που έχουν στρατηγική σημασία. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς κάποιοι, κάποιες επιχειρήσεις ε, κερδίζουν ενώ λαμβάνουν χρήματα από τον ε, δημόσιο κορβανά. Ευχαριστώ κυρία Ιόν Κοχτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Εκτελεστική Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, στο Δεκέμβριο του 2019 η πρόεδρος Ursula von der ανήγγειλε ότι η επιτροπή στην οποία θα προεδρεύσει θα ε, διαδραματίσει ένα ισχυρό γεωπολιτικό ρόλο. Η Λευκή Βίβλος που παρουσιάζεται σήμερα για τις ε, ξένες επιδοτήσεις σίγουρα είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και το χαιρετίζω. Πολλό δε μάλλον που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται εντατικά για τη διαχείριση τη κρίση μέσω και τη προσωρινή πλαισίωση των κρατικών ενισχύσεων. Στην ετήσια έκθεση για την ε, πολιτική ανταγωνισμού, στην οποία είμαι εισηγήτρια και θα ψηφιστεί αύριο, Απευθύνουμε έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με του συναδέλφου για να ενισχύσει την πολιτική ανταγωνισμού στα πλαίσια τη παγκοσμιοποίηση και να εξασφαλίσει αμοιβαιότητα με τι τρίτε χώρε σε θέματα δημοσίων προμηθειών και κρατικών ενισχύσεων έχουμε μια αδιαφυσβήτη διαπίστωση. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τους κανόνες μας στην παρούσα κατάσταση για να αντιμετωπίσουμε κάποια νομικά κενά. Καταρχήν, οι ε, κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει που έχουν, δεν εφαρμόζονται στου ξένους παρόχους, παρόλα αυτά έχουν πρόσβαση στις, στην αγορά μα, και ούτε οι αντιμονοπολιακοί κανόνε ούτε ο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν λαμβάνουν υπόψη τι ε, ξένε επιδοτήσει. Φανταστείτε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα όπου η φιλοξενούμενη ομάδα υπακούει σε πολύ πιο επίκει κανόνε από ότι η ομάδα που παίζει ε, στην έδρα τη. Δεν χρειάζεται καν να παρακολουθήσουμε τον αγώνα. Δεν χρειάζεται να είμαστε medium για να γνωρίζουμε ποιο θα βγει νικητή. Θα είναι παρόλα αυτά άδικο το αποτέλεσμα. Η κρίση του COVID-19 μα ε, χτύπησε το συναγερμό ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τι στρατηγικέ μα επιχειρήσει για να επιτύχουμε μια θεκτική Ευρώπη γιατί δεν θα πρέπει οι επιθετικές εξαγορές να γίνουν κάτι καθημερινό και τετριμένο επειδή δεν θα καταφέρουμε να τις αποτρέψουμε. Χαίρομαι λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει και θα αποτρέψει τέτοιου είδου ε, αρπακτικές συμπεριφορές. Βέβαια έχουμε πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας και ελπίζω ότι η δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσει θα απαντήσει στις εξή ερωτήσεις. Ποια θα είναι η κατανομή των εξουσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Τι ελευθερία θα έχουν τα κράτη-μέλη που τώρα δέχονται ευχαρίστω τι ξένες επενδύσει ε, ή τι εξαγορές ε, των ε, εθνικών του εμβληματικών επιχειρήσεων από ξένες επιχειρήσεις που θα επιδοτούνται δαψιλώς, θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Αλλιώ οι εμπορικοί μας εταίροι θα εκμεταλλευτούν τις διαφορές μας και όχι την ενότητά μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Βανσπάρεντακ. Σας ευχαριστώ. Ε, το ενδιαφέρον του Τραμπ ε, να αγοράσει μια γερμανική εταιρεία ε, μας άνοιξε πραγματικά τα μάτια. Για, χαίρομαι για την πρώτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να αποτραπούν τέτοιες ε, επιθετικές εξαγορές ιδιαίτερα επιχειρήσεων του υγειονομικού τομέα. Νομίζω ότι είναι βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Ο τομέας της υγείας και η φαρμακευτική βιομηχανία είναι κρίσιμη για τη δημόσια υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα η δημόσια υγεία υπερέχει και υπερτερεί των συμφερόντων των μετόχων. Θέλουμε λοιπόν σαφείς κατευθυντήρε γραμμές. Θα πρέπει να αλλάξει και το μοντέλο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τη φαρμακοβιομηχανία, να στηρίζεται στην ανοιχτή επιστήμη και σε διαφανή κόστη αλλά για στη φαρμακοβιομηχανία προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό θα είναι πολύ πιο δύσκολο ε, αν οι φαρμακοβιομηχανίες μας πέσουν σε ξένα χέρια. Γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύσουμε κυρίως τη φαρμακοβιομηχανία μας από επιθετικές εξαγορές, κυρίως ε, από χώρες που έχουν ιδιαίτερα εθνικιστικά συμφέροντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φανόβαρτφελτ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 Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί ε, στην προστασία των ευρωπαϊκών στρατικών κλάδων από εξαγορέ, ιδίως από κρατικούς κινέζικους ομίλους ε, που παίρνουν κρατικές ενισχύσεις, είναι κάτι αξιέπαινο, γιατί η Κίνα δεν τηρεί ε, τους διεθνού εμπορικούς κανόνες. Οι ξένοι επενδυτές ουσιαστικά ε, υποβαθμίζονται και είναι σε μειονεκτική θέση γιατί υπάρχει κρατική ενίσχυση και ε, υπάρχει ε, και έντονη εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Άρα καλή είναι η προστασία των ευρωπαϊκών στρατηγικών κλάδων. Νομίζω ότι δύο κανόνες εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς γιατί χωρίς την εσωτερική αγορά δεν θα μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις μας ε, στην παγκόσμια αγορά και το δεύτερο είναι η δημιουργία ε, της εσωτερικής ε, αγοράς για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Κύριος Μορέλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πόσο χα... πολύ χαμένος χρόνος. Έφτασε το 2020 να έχουμε μια τέτοια κρίση τεράστιων διαστάσεων για να κουνηθεί ε, το Συμβούλιο και, η Επιτροπή και να ε, δυσαρεστηθούν από τις αθέμητες ξένες ε, εμπορικές πρακτικές και να μιλήσουμε για τις ξένες εξαγορές. Το 2020 ε, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ΠΟΕ ή στον ΠΟΕ μάλλον η Κίνα ή η δεν είναι και τόσο υπέρμαχοι της αμοιβαιότητας. Ήμασταν ε, αφελείς, ε, κύριε Βεστάγκερ. Καλό είναι που το αναγνωρίζουμε και καιρό είναι να δράσουμε τώρα σε ό,τι αφορά τη Λευκή Βίβλο. Είναι πολύπλοκη καταρχάς Τρία επίπεδα έρευνας έχετε και πάρα πολλά έντυπα. Ε, πρέπει να είμαστε όμως απλοί ρεαλιστές, να πάμε στην ουσία. Όχι όπως κάνετε πολύ συχνά ε, να θέλετε να έχουμε την τέλεια αγορά. Μα δεν υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ας πάμε στην ουσία λοιπόν. Αυτό πρέπει να προστατεύσουμε. Είναι επιχειρήσει, εχνογνωσία, θέσει εργασία. Ε, χρειαζόμαστε χρηματοδότηση και σε ό,τι αφορά τι ξένε επιχειρήσει θα πρέπει να υποστηρίζονται οι Ευρωπαίοι ευρωπαίες επιχειρήσεις, ευρωπαίοι μισθωτοί και όχι ξένες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το δικαίωμα στην αλήθεια είναι από τα θεμελιώδη δικαιώματα τη ανθρωπότητα. Για να μπορούμε να λάβουμε τεκμηριωμένε και δίκαιε αποφάσει, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά. το 2020 σας είχα ζητήσει να μην κλείσουμε τις πόρτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μείνουμε εδώ και να μάθουμε την αλήθεια για τον ιό και να δούμε ποιες είναι οι διαστάσεις του ιού και ε, της, ε, του COVID-19. Αντί για την έκκληση μου αυτή όμως κλείσαμε τα εισπύλες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι δώσαμε την ευκαιρία και σε άλλους να κλείσουν τις εθνικές βουλές, να ε, κλείσουν την οικονομία τους. Ουσιαστικά κινητοποιήθηκε η οικονομία. Και τι συνέβη, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, μια ανήκουστη και πρωτοφανή οικονομική καταστροφή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά, να καλέσουμε τους, τους πιο κορυφαίους επιδημιολόγους και ιολόγους, να τους θέσουμε ε, ερωτήσεις και να δούμε πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε το 10 τον ε, Οκτώβριο, ας πούμε, στο μέλλον. Θέλω να σας πω. Αγαπητοί ποτέ δεν έκλεισε τις πόρτες του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε η μόνη διεθνής ε, πολύγλωση οργάνωση που συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με πολλές γλώσσες χωρίς να σταματήσουμε καθόλου. Η κυρία Λίντια Περέρα είναι επόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει ολέθριες ε, συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία με τις ε, ε, ευρωπαϊκές εξαγωγές να κινδυνεύουν να μειωθούν μέχρι τα τέλη του έτους κατά 470 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ρευστότητα των αγορών αφήνει τις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες ευάλωτες απέναντι στις ε, εξωτερικές επιθέσεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για να τις προστατεύσουμε κυρίως από εταιρείε ε, ε, που είναι κρατικές ή στι οποίες το κρατικό μερίδιο είναι μεγάλο. Και το παλιό δόγμα ότι το κεφάλαιο δεν έχει εθνικότητα ισχύει μόνο όταν κίνητρο του κεφαλαίου είναι η κερδοφορία. Όταν όμως γίνεται ε, πολιτιστικό ε, εργαλείο, τότε αυτό το δόγμα δεν ισχύει. Και είναι μεγαλύτερη η απειλή όταν βάλετε κατά στρατηγικών κλάδων, ε, υποδομών ή κρίσιμων τεχνολογιών. Θέλουμε λοιπόν μια ρεαλιστική, οικονομικά ελκυστική οικονομική πρόταση για να μπορούμε να προβλέπουμε την πηγή του ξένου κεφαλαίου σε όλη τη διαδικασία της εξαγοράς ή της συγχώνευσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκλουξμαν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λιμάνι του Πειραιά, το αεροδρόμιο της Τουλούζης, Άλστομ, μέχρι στιγμής όλα σε εμά ήταν προς πώληση, προς εκποίηση. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε με την Λευκή Βίβλο και το φιλτράρισμα των ξένων επενδύσεων έχει ζωτική σημασία, αλλά δεν επαρκεί. Θα σας διηγηθώ την ιστορία ενός γαλλικού εργοστασίου, τη Ζέρζατ, που είναι, ε, ήταν το τελευταίο εργοστάσιο που μπορούσε να παράγει φιάλες οξυγόνο για τα νοσοκομεία και την πυροσβεστική. Πριν από ένα ε, χρόνο η Αμερικανική Διεύθυνση του Lux Fair αποφάσισε να κλείσει το εργοστάσιο παρόλο που είχε κέρδη 55%. Ε, και έτσι χάνουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία και εξαρτώμαστε από χώρες όπως η Τουρκία και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Έχουμε ένα ε, πραγματικά βραχίωνα οπλισμένο με 2-3 εκατομμύρια ευρώ για τις ε, ε, παραγγελίες του δημοσίου. Θέλουμε ένα πραγματικά αγοράστε ευρωπαϊκά νόμο. Δεν θα μας ε, το συγχωρήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αν αντί να τις προστατεύσουμε, γονατίσουμε. Ευχαριστώ. Κύριος κύριε Πρόεδρε, Επιτροπή. Θέλουμε να προστατεύσουμε στρατηγικούς κλάδους. Δεν υπάρχει όμως μία και μόνη θαυματουργή λύση. Χρειαζόμαστε μία εργαλειοθήκη. Γι' αυτό και χαιρετίζω τη Λευκή Βίβλο που ουσιαστικά ε, θα δώσει τις επιδοτήσεις αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε και τη διαλογή και το screening των επενδύσεων. Εάν αποφύγουμε επιθετικές εξαγορές σίγουρα η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου μειώθηκε πρόσφατα. Ο αριθμό των επενδύσεων όμως έχει αυξηθεί, κάτι που σημαίνει ότι οι επενδύσεις από την Κίνα ε, απευθύνονται σε μικρότερες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να έχουν στρατηγικό ρόλο. Εκεί ε, έχουν ε, στοχεύσει. Πρέπει νομίζω τους μηχανισμούς ελέγχου των επενδύσεων που θα τεθούν σε τον οποίο θα ήταν καλό να τους μελετήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την προστασία των στρατηγικών κλάδων, κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε είναι και η αλυσίδα εφοδιασμού και θα ήθελα να δω τι γίνεται στην Ιαπωνία. Επενδύουν στην μετεκατάσταση για να προστατεύσουν τα λυσίδα εφοδιασμού από κοινού με τις χώρες Ασεάννα. Μήπως θα έπρεπε να το κάνουμε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και άλλους εταίρους και εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Τόμ Μπέρεντσεν. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι θα είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη περίοδος για να δούμε πώς ε, θα ε, διαμορφώσουμε το μέλλον τη Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς. Χρειαζόμαστε κονδύλια για να προστατεύσουμε τους στρατηγικού κλάδου μας. Σίγουρα όμως πρέπει να τηρούνται οι κανόνε και οι κανόνε θα πρέπει να ε, εξυπηρετούν ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ε, πραγματικά δεν είναι κάτι προ το συμφέρον μας μια εταιρεία παραγωγή εμβολίων ουσιαστικά να τα διαθέσει τα εμβόλια της κατά αποκλειστικότητα στη ΣΥΠΑ πρέπει εμείς τα δικά μας συμφέροντα να προστατεύσουμε. Στις αγορές μας επίσης πρέπει να εφαρμόζονται τα δικά μας πρότυπα, οι δικές μας αρχές και αξίες. Έτσι θα διατηρήσουμε τις αγορές μας ε, την απασχόληση και θα παραμείνουν εδώ οι θέσεις εργασίας και στο μέλλον. Πευθύνομαι στην Κομισιόν, ε, θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να εφαρμόσετε τα σχέδιά σας στην πράξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ο Επίτροπος Φιλ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση για το σημαντικό θέμα και έχω να σας πω και επί συμπερασματικές παρατηρήσεις επιμένω ότι είμαστε μια ανοιχτή αγορά και ότι είναι καλοδεχούμενες οι επενδύσεις και οι ξένες επενδύσεις που φυσικά και θα πρέπει να φιλτρέρονται και συμφωνώ με ε, τον κύριο Γλουξμαν τον κύριο Μπουτικόφερ και τον κύριο Χάνσεν που είπαν ότι ακριβώς θα πρέπει να έχουμε πιο στεγανά μέτρα αλλά έτσι τα θέλησαν οι συνομοθέτες. Μηχανισμό συλλογή δεδομένων, τον θέλανε όπως τον θέλανε, οπότε, ε, βέβαια, σίγουρα έχετε δίκιο και είναι δυνατόν να έχουμε καλύτερο φιλτράρισμα. Οπότε αυτός ο μηχανισμός θα αρχίσει να τρέχει τον Οκτώβριο και θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Επίσης έχουμε δύο θέματα που θέλω να με βοηθήσετε. Πρώτα πρώτα μια ανταπόκριση αποφασιστική ε, σε σχέση με την Λευκή Βίβλο που σας τα εξήγησε η κυρία Βέσταγερ. Ε, να δούμε πώς θα κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις και όσον αφορά το θεμητό ανταγωνισμό για τις εταιρείε μας. Επίσης, η πολιτική σας υποστήριξη είναι καλοδεχούμενη όσον αφορά ε, τους διεθνείς διαγωνισμούς που ακόμη ε, χρειάζεται ένα μικρό σπρόξιμο από τα θεσμικά όργανα. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε για να περάσει αυτή η νομοθεσία και να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπος Βεστάγκερ. Well, thank you. Ευχαριστώ πολύ, λέει κύριε Βεστάγκερ να συμφωνήσω με όσα είπε ο συνάδελφος αλλά και ο κύριος Μπουτικόφερ το είπε πρώτος χρειάζεται αυτό που λέμε εργαλειοθήκη μαγικές, ξαφνικές α, ακαρίες λύσεις δεν υπάρχουν άρα λύσεις όμως ναι μπορούν να εξευρεθούν οπότε θέλω να σας πω ότι δεν θέλουμε ε, να θυσιάσουμε τον θεμητό ανταγωνισμό γιατί μας βοηθάει, βοηθάει τις εταιρείε μας φέρνει καλές τιμές και καινοτομία. Φυσικά, από την άλλη μεριά, δεν θα απεμπολίσουμε αυτό το πιστεύω στην, στον, ε, στον αθέμητο ανταγωνισμό για τις εταιρείε μας και οπότε θα δούμε τι γίνεται με τις εξαγορές, με τις κρατικές επιδοτήσεις ε, και ε, ακριβώς το, να υποστηρίζεται κάποιες εταιρείες το λειτουργικό κόστος, αυτό είναι η επιδότηση. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα ενθαρρυνθούν οι συνομοθήτες. Και εσείς θα ενθαρρύνετε το Συμβουλίο. Χρειαζόμαστε αμοιβιότητα και χρειαζόμαστε επίσης και τα σχετικά μέσα. Καλύτεροι κανόνες για τους διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός είναι διαγωνισμός και άρα να είμαστε αυτοί που να αφήνουν να κερδίσει όχι αυτός που έχει την επιδότηση στη τσέπη αλλά αυτός που είναι πιο αποτελεσματικός κάνουν ό,τι μπορούν τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ε, κλείσουν τις πληγές ε, της ε, πανδημίας αλλά όμως εμείς είμαστε κάποιοι που έχουν διαφάνεια έτσι θέλουμε να γίνει η ανάκαμψη και να ξανακερδίσουμε τις χαμένες θέσεις εργασίας όμως στις ξένες επενδύσεις δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει έλεγχος. Ε, για αυτό και συζητάμε το θέμα και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και περιμένω επίσης την βοήθεια σας και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Η κυρία ε, Μπρίνιας έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτές, πολύ χρήσιμη συζήτηση για όλους μας και σας ευχαριστώ γιατί είσαστε συνεχώς στρατευμένοι σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ για όσα είπατε. Θα τα μεταφέρω στους συναδέλφους στο Συμβούλιο και όπως είπαμε προηγουμένως η οικονομική κρίση κατόπιν της πανδημίας ε, έφερε πολλές εταιρείε σε θέση ευάλωτη σε σχέση με αυτές τι επιθετικές εξαγορές. Εμείς θα εξασφαλίσουμε το ότι θα προστατευτούν οι εταιρείε, οι κλάδοι που έχουν στρατηγική σημασία και στη συνέχεια με την ανάκαμψη νέα νομοθεσία θέλουμε για να υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό για αυτό το φιλτράρισμα των μεδίσεων. Αυτό που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 19 από Συμβουλίο και Κοινοβούλιο. Τώρα αυτό το νομοθέτημα έχει τεθεί σε ισχύ ε, και θα τεθεί σε ισχύ οριστικά στις 11 Δεκάτου του 20. Επαναλαμβάνω, τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να προστατεύσουν τις εταιρείε. εταιρείες, τεχνολογία από τέτοιες ξένες επενδύσεις που θέτουν εν κινδύνο τους ε, στόχους των πολιτικών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτού προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης. Έχουμε το δεύτερο γύρο ε, ψηφοφοριών σε σχέση ε, με τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν από τις 20 και 23 έως τις 45 έχετε χρόνο για να ψηφίσετε ακριβώ με την ίδια διαδικασία που τη γνωρίζετε πλέον. Είναι ονομαστικές όλες οι ψηφοφορίες και μπορείτε να ψηφίσετε και θα βρείτε και ε, τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα. Άρα τώρα κηρύσω την έναρξη την ε, σε δεύτερης ψηφοφορίας μέχρι τις 21.45 και αύριο στις 9 το πρωί στην έναρξη δηλαδή της πρωινής ε, συνόδου, της πρωινής συνεδρίας Ολομέλειας θα δημοσιοποιηθούν, θα ανακοινωθούν και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο ε, θέμα της ε, ημερήσιας ε, διάταξης για τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά. Και να επαναλάβω για τελευταία φορά για σήμερα ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπλε κάρτα ούτε να προσεκίσετε την προσοχή του για να λάβετε το λόγο αυθορμήτως. Ε, το λόγο έχει η Επίτροπος. Παρακαλώ, κυρία Βαλέα. Well. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση αυτή. θα συζητήσουμε κάτι που μας απασχολεί όλους σήμερα. Ποιο είναι το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκαμψη του τουρισμού και των μεταφορών. Ε, γιατί πέστησαν τρομερές συνέπειες με την πανδημία COVID-19. Χαίρομαι που ξαναβλεπόμαστε. Ε, εν ώψη των θερινών διακοπών θα πρέπει να συζητήσουμε από κοινού τον τουρισμό και τις μεταφορές για να δούμε ε, γιατί πώς θα πάμε διακοπές αν δεν έχουμε απρόσκαπτη ε, μετακίνηση των μέσων μεταφοράς. Ε, και επίσης ε, για να κινηθεί και ο κόσμος χρειάζεται συντονισμός και εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, αποφυγή των διακρίσεων και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Σίγουρα ο τουρισμό και οι μεταφορές ήταν από τους, ε, από που δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία, κυρίως η μεταφορά επιβατών. Ε, μειώθηκαν κατά 80% οι μεταφορές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι μεταφορές ε, είναι σημαντικός κλάδος που κινητοποιεί και άλλου τομεί όπως τον τουρισμό και άλλου, που είναι σημαντικά Μεταφορέ της οικονομίας. Ε, οι μεταφορές είναι ρεχοκοκαλιά της οικονομίας. Η αποκατάσταση των μεταφορών λοιπόν και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιταχυνθεί, έχοντα φυσικά υπόψη και κάποια υγειονομικά κριτήρια. Στις 13 Μαΐου στις κατευθυντήριες γραμμές μας θέτουμε ένα πλαίσιο για σταδιακή και ε, ε, ασφαλή επιστροφή της συνδεσιμότητας των μεταφορών και σε όλες τις υπηρεσίες μεταφορών και έχουμε και ειδικέ συστάσεις για κάθε μέσο μεταφοράς. Προτείναμε κατευθυντήρες γραμμές και για την ασφαλή συνέχιση των τουριστικών υπηρεσιών στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια και στα ταξιδιωτικά πρακτορία. Επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές προτάθηκαν για την αποκατάσταση της ελεύθερης διακίνησης και για την έκδοση πιο ελκυστικών κουπονιών. Όλα αυτά τα μέσα θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη αυτών των σημαντικών κλάδων της οικονομίας. Γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία αυτό το καλοκαίρι του 2020. Φυσικά καμία δράση δεν είναι απόλυτα κίνδυνη. Έχουμε όμως αναπτύξει κάποια πρωτόκολλα και στη συνεργασία με τους οργανισμούς. Έχουμε κάποια ε, πρωτόκολλα και μέτρα για τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να μειώσουμε τους κινδύνους και να διευκολύνουμε την ε, επαναφορά των, των συγκοινωνιών και της μετακίνησης. Θέλουμε φυσικά και καλή ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε κάθε πολίτη να μπορεί τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα να κάνει τι αποφάσει του για να περιορίσει τον υγειονομικό κίνδυνο κατά τα ταξίδια του. Τα μέτρα που θα επιβληθούν στι μεταφορέ θα πρέπει να είναι αναλογικά και να βασίζονται στον κίνδυνο. Και επίση τα κράτη-μέλη από αυτή την εβδομάδα θα άρουν τα περιοριστικά μέτρα για τις μεταφορές και τους περιορισμούς στα εσωτερικά σύνορα. Θα καταργηθούν πια αυτά τα μέτρα και θα υιοθετηθούν πιο στοχευμένα μέτρα. Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, καλύτερος καθαρισμός, προτεραιότητα στα ηλεκτρονικά εισιτήρια και αποφυγή του συνοστισμού στους κόμβου. Επιπλέον, αυτά τα στοχευμένα μέτρα θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη που χρειάζεται ο κόσμος για να ξαναρχίσει τα ταξίδια και τι μετα... μετακινήσεις. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της αεροπορίας ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Πολιτική Αεροπορία και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη των Νόσων έχουν εκδώσει συμπληρωματικέ ε, ε λειτουργικέ κατευθυντήριε γραμμέ με βάση κατευθυντήριε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων. Επίση, ε, προβλέπονται κάποια ειδικά φίλτρα που θα περιληφθούν στα αεροπλάνα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σε αποδεκτά επίπεδα στις αεροπορικές μεταφορές. Θα πρέπει να συνεργαστούμε γιατί οι μεταφορές είναι διασυνοριακή και διαπεριφερειακή δραστηριότητα. Είναι αυτονόητο ότι οι ιστορικοί σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι συντονισμένοι και ό,τι μέτρα εφαρμόζονται στα σημεία αύξησης και ε, προορισμού να είναι αμοιβαίω αποδεκτοί. Αλλιώς ε, οι μεταφορές θα γίνουν ε, επικίνδυνα βεβαρημένες και αποτρεπτικά δαπανηρές. Τέτοιο φυσικά προποθέτει την ε, συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των σημείων επαφή για τι μεταφορέ που θεσπίστηκαν κατά την έναρξη τη πανδημία, με βάση κατευθυντήριε γραμμέ για τι πράσινε λωρίδε. Η ασφάλεια βέβαια δεν είναι το μόνο που χρειαζόμαστε για να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στηρίζεται και σε προηγούμενα. Και το προηγούμενο που θέλαμε να προσπίσουμε είναι να προστατεύσουμε του καταναλωτέ μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανα πάσα στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σαφής καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης ότι το δικαίωμα των επιβατών για επιστροφή των χρημάτων δεν θα περιοριστεί. Οι καταναλωστές και κυρίως όσοι έχουν πληγεί οικονομικά από την κρίση θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν για αναψυχή και τουρισμό αν είναι σίγουροι ότι θα επιστραφούν τα χρήματα των εισιτηρίων και των πακέτων που έχουν αγοράσει σε περίπτωση που ακυρωθούν τα ταξίδια. Επίσης, Θέλουμε συνέχιση ε, των δραστηριοτήτων για όλους τους τομείς. Γι' αυτό και η δημόσια στήριξη των ε, επιχειρήσεων για να κρατηθούν ζωντανές οι επενδύσεις είναι σημαντικά προαπαιτούμενα για να ανακτήσουμε τη διασυνδεσιμότητα και να έχουμε μεταφορές που θα αντέξουν και στο μέλλον. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα εύρωστο και περιεκτικό πακέτο για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και μπορεί κάποιοι οικονομικοί τομεί να μην έχουν συγκεκριμένη επιδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης, από το σχέδιο ανάκαμψη, κάποιοι σημαντικοί τομεί όπω ο τουρισμό και οι μεταφορέ θα υποφεληθούν από πολλέ χρηματοδοτικέ δυνατότητε. Για να εξασφαλίσουμε υποστήριξη για το πακέτο αυτό, θέλουμε τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πραγματικά θα δώσουμε χρηματοδοτικέ. Ε, ευκαιρίες ε, στις μεταφορές, στον τουρισμό, αεροναυπηγική, ναυπηγική και όλους τους τομείς που χρειάζονται για να έχουμε συνδεσιμότητα στις μεταφορές σε προσιτές τιμές για το 2020 και επέκεινα. Ελπίζω να χρησιμοποιηθούν όλα τα κοινοτικά μέσα για να εξασφαλιστεί η ρευστότητα ε, των επιχειρήσεων και να επιστρέψουν στον δρόμο της ανάκαμψης. Μάλιστα, Έχουμε προτείνει και το σχέδιο ανάκαμψης με πολλές ε, δυνατότητες ε, για τον τουρισμό. 1,1 δις 1,13 ε, μάλλον για το σχέδιο ανάπτυξη και πάνω από 500 δις για τις μεταφορές. Επίσης, έχουμε ένα νέο ενισχυμένο κανονισμό ε, για το σύνδετο στην Ευρώπη με 1,5 επιπλέον δισεκατομμύρια για την ενίσχυση των υποδομών. Θα επιταχυνθεί και η ολοκλήρωση των, ε, του κεντρικού δικτύου του διευρωπαϊκών δικτύων ε, μεταφορών και θα δώσουμε ναύσματα για την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση προκειμένου να ε, υιοθετήσουμε πιο φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες και θα ενισχύσουμε και τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων με βάση το θεματολόγιο για την Πράσινη Συμφωνία. Επίσης έχουμε αυξανόμενο InvestEU ε, με 1,3 δις με νέο, νέα επενδυτική πρωτοβουλία για να στηρίξουμε κρίσιμες υποδομές και την ανάπτυξη ανθεκτικών αξιακών αλυσίδων και ε, επίσης νέες τεχνολογίες που χρειάζονται για τις μεταφορές και επίσης ένα, ε, μια νέα θηρίδα βιώσιμων επενδύσεων που είναι διπλάσια θα έχει εγγυήσεις 20 δις εκατομμυρίων για να προσελκύσει και ιδιωτικές επενδύσεις για τις υποδομές των μεταφορών. Οπότε με 560 δισεκατομμύρια η χρηματοδοτική αυτή δυνατότητα θα ευνοήσει όλους τους ε, κλάδους των μεταφορών. Τα κράτη-μέλη μπορούν να υποβάλουν τα σχέδια ανάκαμψης και θεκτικότητας μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο για να λάβουν δάνεια οι επιδοτήσεις και είμαι βέβαια ότι οι επενδύσεις σε βιώσιμα συστήματα μεταφορών θα είναι πολλές και θα δοθεί προτεραιότητα στα κράτη-μέλη όπως φαίνεται σε όλες τις εκθέσεις αναχώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στις οποίες ε, θα στηρίζεται το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων με 26 δις κονδύλιο που επίσης μπορεί να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις για να στηριχθούν ε, επιλέξιμες επιχειρήσεις στους τομείς που έχουν πληγεί κυρίως από την πανδημία. Με όλα αυτά τα μέσα θα προωθούμε τις προτεραιότητες της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης και στην επικείμενη μας στρατηγική για τις μεταφορές ε, και στη σχετική ανακοίνωση ε, θα επικεντρωθούμε σε όλα αυτά. Γιατί η πανδημία άλλαξε πολλά, αλλά όχι την ανάγκη για έξυπνη κινητικότητα. 80% του συνολικού προπολογισμού ε, έχει αφιερωθεί στην περιβαλλοντική δράση και ο συνολικός μας στόχος είναι 25% ε, του, της συνεκτίμησης του κλίματος ε, για τους τομείς γενικώ για, το, για τις μεταφορές θα είναι υψηλότερο το ποσοστό. Χαίρομαι για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισημαίνει πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Όσο προχωρούμε θα αντλούμε διδάγματα και από την πρόσφατη εμπειρία μας γιατί η κατάσταση όντως ήταν πρωτοφανής και θα τολμούσα να πω ότι είμαστε τώρα καλύτερα προετοιμασμένοι και σοφότεροι. Ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλιά σας. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Βαλεάν για τη δήλωση αυτή και τώρα ξεκινάει η συζήτηση η κυρία Στάρα Φεραγκού, την πρώτη ομιλήτρια Ρώσα. Ευχαριστώ πολύ. Ο τουριστικός κλάδος και οι μεταφορές σίγουρα είναι οι πλέον πληγέντες από την πανδημία ένα τρίτο της ανθρωπότητας ε, σε εγκλισμό, κάτω από 90%, ε, περισσότερο από 90% των μεταφορών έχει σταματήσει και γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τον τουρισμό είναι ο πρώτος προορισμός. Μιλάμε για τη συνοχή, για την αλληλεγγύη, για τον πολιτισμό, για τη διάρθρωση, για το μέλλον. Όλα αυτά είναι ο τουρισμός. Χρειάζεται ευρωπαϊκή ανταπόκριση. Ε, θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή και από την Ισπανία και ζητούμε πρώτα απ' όλα κατά προτεραιότητα στο σχέδιο ανάκτηση ε, να ασχοληθούμε με τον τουρισμό. Θέλουμε έναν οδικό χάρτη, θέλουμε σαφή στοιχεία, θέλουμε συντονισμό, θέλουμε ασφάλεια ασφάλεια στα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και στα πρωτόκολλα πρέπει να είναι κοινά. Τα ευρωπαϊκά μέτρα πρέπει να αναγνωρίζουν ε, τα μεν, τα δε και να λαμβάνουν υπόψη μα και τι ΜΜΕ που είναι ο παραγωγικό ιστό ε, του τουρισμού κατά 1%. Θέλουμε συνδεσιμότητα για τι Βαλεαρίδε, ε, για τα Κανάρια, για τι απόκεντρε περιφέρειε και επίση χρειαζόμαστε μια στρατηγική για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού. Απευθύνουμε έκκληση για ανάληψη δράση. Ούτε ένα λεπτό δεν πρέπει να χάσουμε, γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι το μέλλον της Ευρώπης. Χωρίς αλληλεγγύη η Ευρώπη δεν υπάρχει. Ούτε όμως και χωρίς τουρισμό θα μπορέσει να υπάρξει Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Συνάλφος Γιουέλη. Ιστβαν Γιουέλη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως σοσιαλδημοκράτης, ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να πω ότι εκπροσωπώ 27 εκατομμύρια εργαζομένους και Ούγγρους εργαζομένους ρεσεψιονίστε, εινολόγους ή ε, αεροσυνοδούς. Όλοι μας ρωτούν τι κάνετε για να μας βοηθήσετε διότι οι κυβερνήσει θεωρούσαν μέχρι τώρα τον τουρισμό ως κάτι, ε, ως μία κότα που γεννάει τα χρυσά αυγά, ε, αλλά δεν χρειάζεται να την ταΐσεις. Ε. πάντα θα φέρνει έσοδα. Τώρα όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι και τόσο δεδομένο. Γι' αυτό λοιπόν οι σοσιαλδημοκράτες ζητούμε άμεση ανάληψη δράσης και ένα σχέδιο ανάκαμψης για την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας. Θέλουμε ένα σχέδιο διαχείρισης της κρίσης. Ένα σύστημα εγγύησης για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες. Θέλουμε να υπάρχει βιωσιμότητα και στο μέλλον. Άρα νέα ευφύ στρατηγική. Αυτό είναι που χρειάζεται. Αυτή είναι η πρότασή μας. Πρέπει να στηριχθεί αυτός ο κλάδος για να μπορέσει να επιβιώσει. Και έπειτα χρειάζεται και ένα ευφυές σχέδιο για να μπορεί και στο μέλλον να είναι βιώσιμος ο τουρισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριος Μπαουθά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εδώ και μήνες ακούμε δεδομένα, στοιχεία και αφηρημένες ιδέες, μα είναι στρατηγικός τομέας αυτός. Η Κομισιόν ακριβώς ασχολήθηκε με αυτό αλλά δεν είναι εδώ να αρκέσουν τόσο έχουν μέχρι τώρα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες συστάσεις για το ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια στη βοήθεια προς τα Γιατί στις 13 Μαΐου είπε η Κομισιόν ότι θα σταμάτησαν οι καραντίνες, όμως κάποιες χώρες είχαν καραντίνα όπως η Ισπανία. Γιατί άνοιξαν τα σύνορα χωρίς συντονισμό μα ήταν χώρες που είχαν τα ίδια επιδημιουργία χαρακτηριστικά αλλά δεν, δεν άνοιξαν μαζί τα σύνορά τους γιατί ε, βλέπουμε ότι ο ένας κοντράρει τον άλλο στην γιατί έχουμε το, το, 12% των εργαζομένων που δεν πήραν ούτε μία δεκάρα ε, όσον αφορά τον τουρισμό που δουλεύουν εκεί γιατί τον έχει βάλει σε δεύτερη κατηγορία τον τουρισμό η Κομισιόν. Το έχουμε πει πολλέ σε πολλές φορές και συνεχίζουμε και το ακούμε αυτό γιατί είπαμε ότι πτώχευσε η Τόμας και οπότε αυτό έδειξε ότι χρειάζεται μια στρατηγική κοινή και έτσι να μπορέσουμε να μην ενεργούμε στο γόνατο αλλά είμαστε προνοητικοί. Κι όμως μετά την Thomas Κουκ ήρθε η κατάσταση με την κρίση. Και ε, Αδάνος ε, ως εκπρόσωπος των Βαλιαρίδων ε, προέρχομαι από κάπου που ο τουρισμό είναι πολύ σημαντικό και μα χρειάζεται να έχουμε τρεις καινούριου πυλώνες, άνοιγμα των συνόρων, κοινά πρότυπα ασφάλειας και επίσης να υπάρξει διαφήμιση της Ευρώπης ως προορισμού τουριστικού. Εμεί είμαστε στο πλάι σας. Πρέπει η Ευρώπη να γίνει πρωταγωνίστρια. Είμαστε συνεχώς ε, στο πλάι σας για τον τουρισμό, για την Ευρώπη, για τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Αδελφό ε, Ρόμαν Χάντερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ ε, έχει πληγεί πάρα πολύ ε, βαριά, ίσω βαρύτερα από οποιοδήποτε άλλο κλάδο, το μέσο του τουρισμού. Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαντελάιεν όμω σήμερα δεν είπε τίποτα για τον τουρισμό. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για τον πάρα πολύ σημαντικό νευραλγικό τουριστικό κλάδο αλλά και για τις μεταφορές στην Ευρώπη είναι ε, από την αρχή, ε, μάλλον καταρχάς μη γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις, οι και επίσης ε, θα πρέπει ε, να δούμε τι θα γίνει και με την πράσινη συμφωνία και αυτούς τους στόχους ε, που υπάρχουν για τον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού. Αυτό ε, θα είναι πραγματικά κάτι που θα δημιουργήσει μεγάλους περιορισμούς αυτή τη στιγμή εάν επιμείνουμε σε αυτούς τους στόχους όταν προσπαθούν οι κλάδοι αυτοί να ορθοποδήσουν. Θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, η απαραίτητη ενίσχυση και τα ταυτόχρονα ε, τα κίνητρα ώστε να μπορέσουν να φιλοπεριβαλλοντικοί αυτοί οι τομεί. Κυρία Τίλιμέτς, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, μετά τα μέτρα εγκλισμού και απομόνωσης για την COVID-19 χρειάζεται συντονισμένη και συντεταγμένη ε, επανέναρξη της δραστηριότητας τουριστικής ε, και των μεταφορών. Θα πρέπει να δούμε προς το μέλλον, προς τα εμπρός και θέλουμε να προ προωθήσουμε έναν τουρισμό ε, μεταφορές που επιθυμούμε για το μέλλον δεν ε, ε, θα πάψει ε, να υπάρχει τουρισμός, δεν θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν μεταφορές και μετά την κρίση. Σίγουρα υπάρχει το οικολογικό αποτύπωμα το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη. Ξέρουμε ότι μετά από την επιδημία άλλαξαν σημαντικά οι συνήθειες πολλών συμπολιτών μας. Περισσότερο περισσότεροι στο σπίτι, δεν μπορούσαν να βγουν καν για ένα περίπατο, δεν μπορούσαν φυσικά να ταξιδέψουν. Πρέπει τώρα να διαμορφώσουμε εκ νέου με βιώσιμο τρόπο τον τουρισμό, ε, ιδίω ε, ε, τις σιδηροδρόμους. Πρέπει να ενισχύσουμε τις υποδομές. Επίσης, θέλουμε να προωθήσουμε την οικολογική γεωργία, να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ήπαθρο, να προωθήσουμε τον αγροτουρισμό. Θέλουμε έναν βιώσιμο τουρισμό στην Ευρώπη για να έχουμε μια κατάσταση όπου όλοι θα είναι κερδισμένοι, θα έχουμε έσοδα, θα έχουμε έχουμε υγιές περιβάλλον, ε, θα έχουμε ε, ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς και πολύ ωραίες εμπειρίες και έσοδα για τον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ Κύριο Ζλωτόφσκι. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Επίτροπε, λίγοι ήταν οι κλάδοι που υπέστησαν τόσο τεράστιες ζημιές από την πανδημία όπως ο, οι μεταφορές και ο τουρισμός. Μέρα με τη μέρα επιχειρήσεις του κλάδου χρειάστηκε να βάλουν λουκέτο. Η ανάκτηση του δυναμικού της θα τους πάρει χρόνια και θα απαιτήσει τεράστια οργανωτική και οικονομική προσπάθεια που αυτή τη στιγμή την επομίζονται τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και απλές κατευθυντήρες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκούν. Χρειάζεται ουσιαστική υποστήριξη που δεν θα επιβαρύνεται με ανέφικτους κλιματικούς στόχους. Η θέσπιση νέων διατάξεων, όπως το πολυδάπανο και επιζήμιο πακέτο κινητοποίησης, θα πρέπει να ανασταλούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια επανεξέταση των διατάξεων που σε αυτού του έκτακτου καιρού μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον επιβαρύνσει. Τη σωστή κατεύθυνση έδωσαν 15 κράτη-μέλη που απέθυναν έκκληση για τα κουπόνια στις αεροπορικές μεταφορές. Κρίμα που στο θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε κάποια λογικά επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Um Ευχαριστώ κυρία Κουντουρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ο τουρισμός είναι ισχυρός επιταχυντής της ανάπτυξης και ο οικονομικός κλάδος που χτυπήθηκε περισσότερο από την υγειονομική κρίση. Κινδυνεύουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας με υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων, με οριζόντιες μειώσεις μισθών και εισοδημάτων ο τουρισμός είναι οι άνθρωποι της φιλοξενίας και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτούς. οφείλουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασφικτιούν από έλλειψη ρευστότητας για να επιβιώσουν στην κρίσιμη αυτή περίοδο να αποτρέψουμε χρεοκοπίες εξαγορές τους από ισχυρού και σοβαρές στρεβλώσεις στις τιμές που θα πλήξουν τον υγιή ανταγωνισμό την αγορά και τους ίδιους τους καταναλωτές. σήμερα λοιπόν ζητάμε την ασφαλή επανεκκίνηση των ταξιδιών με μαζικά τεστ χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών την άμεση στήριξη της εργασίας και των επιχειρήσεων για να παραμείνουν ανταγωνιστικές την επόμενη μέρα και ουσιαστικά εργαλεία για το μέλλον προϋπολογισμό για τον τουρισμό ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων που να περιλαμβάνει προστασία και αποζημίωση των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτωχεύσεων και μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ντορίν Ροκμάκερ. Εσείς παρακαλώ το λόγο. Βρισκόμαστε στην κρίση προβλήματα στις μεταφορές, αλλά οι μεταφορές είναι και η λύση. Γιατί να Θέλουμε ένα τέτοιο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, ένα τρένο που να συνδέει τις βασικές πόλεις και όλα αυτά εν μέσω της κρίσης. Διότι οι δημόσιες δαπάνες σώζουν από την κρίση. Είναι λογικό αυτό. Επενδύοντας σε ένα πρόγραμμα πράσινο περιβαλλοντικό έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Κάτι καλό για όλους. Αυτό είναι κάτι το λογικό και οι επενδύσεις στις υποδομές χρειάζονται για να έρθει η οικονομική ανάπτυξη. Οι γενιές στο μέλλον θα πρέπει να ξέρουν πού πήγαν τα χρήματα που δαπανούμε σήμερα. Ε, για αυτό και χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, πρακτικό, με την κατάλληλη προοικοδότηση. Ε, για αυτό και θα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο τρένο, ένα τέτοιο τρένο ψηλής ταχύτητας και ένα τέτοιο δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας. Ευχαριστώ κύριος Μασιμιλιάνο Σαλίνη. Ο κύριος Σαλίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση που μας δίνει την δυνατότητα να επεξεργαστούμε αυτό το κείμενο το οποίο όπως είπε ένας συνάδελφος και το επαναλάβαμε έναν στρατηγικό τομέα όπου οι επιπτώσεις της ε, κρίσης συνολικά τον χτύπησαν, τον, τον έφεραν σε ευάλωτη θέση γιατί πρόκειται για έναν ε, κλάδο πάρα πολύ σημαντικό. Έχει οριζόντιο χαρακτήρα ο τουρισμός, ε, έχει σχέση με μεταφορές, με πολιτισμό, με οικονομική ανάπτυξη και υπάρχει και κάτι, υπάρχει κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να προσεχθεί και να πλαισιωθεί και δημιουργικά. Πρόκειται για το πώς θα πλαισιώσουμε ε, την επαγγελματικότητα όλων ε, αυτών, όλων αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πασχίζοντας τόσα χρόνια ε, φτιάξανε αυτοί που έχουν αυτές τις εταιρείες ένα πάρα πολύ ικανό προσωπικό. Τώρα αυτοί όλοι θα χαθούν. Μιλάμε για εστιατόρια, για ξενοδοχεία που τώρα αυτοί θα χαθούν ως δυναμικό. Οπότε και οι επιπτώσει κοινωνικέ θα είναι πολύ σοβαρέ και όλοι θα πληρώσουμε την νύφη. Είναι και θέμα και πολιτιστικό. Σα ευχαριστούμε. Γιώχαν Ντάνιλσον. Γιώχαν Ντάνιλσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, είναι θέμα επίκαιρο. Γιατί αυτή τη βδομάδα άνοιξαν τα περισσότερα σύνορα και πάλι. Να, τώρα έχουμε τις θερινές διακοπές. Πολύ σημαντικό αυτό για τον τουρισμό και τα ταξίδια στην Ευρώπη. Μπορούμε να ξανακάνουμε επομένως τουρισμό, αλλά πάντως πρόκειται σίγουρα για έναν κλάδο πολύ σημαντικό, ε, φέρνει πάρα πολύ εισόδημα, οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχουν ασφάλεια αυτοί που θα κάνουν τουρισμό, να είναι ασφαλείς στα ξενοδοχεία, στα μέσα μεταφοράς, αλλά να είναι ασφαλείς και όλοι όσοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, τον τουριστικό, να αισθάνονται ασφαλείς όταν πάνε να δουλέψουν. Οπότε όταν ανοίξει η οικονομία σιγά σιγά να εξασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια α, όλων αυτών είναι επομένω πάρα πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να είναι ασφαλείς και να έχουν υγεία. Ο κύριος Μάρκο Καμπομενόζη. Θα σας τα πω στα Ιταλικά, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βαλιάν που ήρθατε με αυτή η ευκαιρία της ανταλλαγής απόψεων και με εσά και με την άλλη μεριά βέβαια είχαμε τον κύριο Λεμπρετών ε, που μας τα είπε διαφορετικά όσον αφορά τις επιπτώσεις σε τουρισμό, και σε μεταφορές ε, ε, από την κρίση και απόψε. Όμως θέλω να μιλήσω για τον τουρισμό, διότι όπως είπαν οι συνάδελφοι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο και για την Ιταλία, τη χώρα μου, είναι το 13% του ΑΕΠ και είπαμε πολλά για το τι μπορούμε να κάνουμε ως οικονομική δημιουργική παρέμβαση ε, φυσικά θα πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, να βοηθήσουμε και νομοθετικά και από τις Βρυξέλλες να γίνει αυτή η προσπάθεια και μιλώ για την οδηγία για τις υπηρεσίες και μας τα είπε ο κύριος Μπρετών ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το πεδίο εφαρμογή, τι θα γίνει με το ότι έχουν μπλοκαριστεί οι επενδύσεις στα, στους, στους χώρους παραθερισμού και το 2020 θα πρέπει κάτι φέτος να γίνει για να δοθούν αυτές οι αγαπητές παρεκκλήσεις. Ευχαριστώ κύριος Λούγκριν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τη γνώμη ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να ανακατευτεί στον τουρισμό. Ο τουρισμός θα πρέπει να είναι τοπικό, περιφερειακό και εθνικό ζήτημα γιατί το να έχουμε μία υπέρτατη αρχή δεν θα μας εξασφαλίσει ένα τουρισμό φέτος το καλοκαίρι. Στη Σουηδία είχαμε τόσο κακή διαχείριση της πανδημίας COVID που οι Σουηδοί δεν μπορούν καν να ταξιδέψουν σε ορισμένες χώρες. Οπότε θα χρειαστεί σίγουρα χρόνος για να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα και να έχουμε ένα τουρισμό όπως τον θυμόμαστε. Θα χρειαστεί χρόνος για να ξεπεράσουμε την πανδημία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όμως τον τουρισμό και πιστεύω ότι θα το κάνουμε καλύτερα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Δεν χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χώνει τη μύτη της παντού, ακόμη και εκεί που τα κράτη-μέλη θα είναι πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ κύριο Σισμάιλ Ερτούκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Πιστεύω ότι η κρίση του κορονοϊού μας έδειξε πολύ καλά τα όρια μας. Μας έδειξε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν είναι ακόμα η Ένωση την οποία επιθυμούμε. Αυτό σημαίνει όμως ότι μπορούμε να δουλέψουμε ώστε να γίνει καλύτερη αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 27 εκατομμύρια ανθρώπους ε, οι οποίοι εργάζονται στα τουριστικά επαγγέλματα, 10,3%. Κυρία Επίτροπε γνωρίζετε αυτά τα νούμερα, 10,3% του ΑΕΠ και σε ό,τι αφορά ε, το, τα δισεκατομμύρια ευρώ ε, τζίρο ε, των τουριστικών επιχειρήσεων που χάνεται, εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος στις μικρές επιχειρήσεις, στα ταξιδιωτικά γραφεία. Προβλήματα ρευστότητας είναι πάρα πολύ μεγάλα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης 5 με 7 δις θα κοστίσει αυτό αυτή πρόταση σε σχέση με 32 και κάτι ε, που έχουν διαθέσει για τη διάσωση των αεροπορικών επιχειρήσεων είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό και νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η δημιουργία αυτού του ταμείου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα θα πάρει το λόγο η κυρία Βαλεάν για να κλείσει με τις καταληκτικές παρατήσεις αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι όλοι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Αναγνωρίζουμε όλοι τη σημασία του τουριστικού κλάδου και του κλάδου των μεταφορών για τις οικονομίες των χωρών μας και όλοι ανησυχούμε. Ποια θα είναι η εξέλιξη, πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον και πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Πώς είπα και στην αρχή όταν έδωσα νομίζω κάποια στοιχεία Ξέρετε τι σκέφτομαι και φαντάζομαι ότι και εσείς, πολλοί από εσάς, το ίδιο πιστεύετε. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο εκτάκτης ανάγκης, ώστε την επόμενη φορά που, μακάρι να μην συμβεί βέβαια, έχουμε κάτι ανάλογο, να είμαστε προετοιμασμένοι. Παραδείγματο χάρη, να έχουμε ένα δεύτερο κύμα ε, της επιδημίας. Πρέπει να διδαχθούμε τα μαθήματα αυτά τα οποία πήραμε, να τα αφομοιώσουμε, να μάθουμε από αυτή την κρίση. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Το είπε και ο κύριος Σερτούγκ. Γιατί πράγματι μας έδειξε τα όρια μας η πανδημία. Πράγματι έχει πληγεί πάρα πολύ ο τουριστικός κλάδος και σίγουρα είναι μια μακρά συζήτηση αυτή για την επικουρικότητα και τι πρέπει να κάνουν τα κρατημέλη, τι πρέπει να κάνει η Κομισιόν, ε, σε ποιο βαθμό πρέπει να παρεμβαίνει κτλ. Φυσικά όποτε υπάρχει ένα πρόβλημα όλοι στρέφουν το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μακάρι, μακάρι να είχαμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε επαρκώς τον κλάδο. Δεν είχαμε όμως τα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ρευστότητας. Περάσαμε λοιπόν ε, σε αυτό το ευέλικτο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για να βοηθήσει με τη ρευστότητα τα κρατημέλη. Πρέπει να προστατεύσουμε πίσω του καταναλωτέ. Να βοηθήσουμε και τι επιχειρήσει. Υπάρχει η ιδέα αυτή που ακούγεται, γιατί είναι ένα μάθημα που έχουμε πάρει, τι γίνεται με τα θέματα της ρευστότητα. Ε? Τι γίνεται με τις ακυρώσεις ε? και τα τεράστια ποσά αποζημιώσεων αυτή δεν Ευρωπαϊκού Ταμείου. Καλή είναι, αλλά πού θα βρεθεί ο προπολογισμό. Αυτό είναι το θέμα. Αν θέλουν να βάλουν ε, σε ένα κοινό κορβανά για κάτι τέτοιο τα κράτη-μέλη, καλό είναι αυτό. Αλλά αν έχετε υπόψη όλε αυτέ τι πολύπλοκε συζητήσει που είχαμε για το ΠΙΔΕΛΤΑΠ και τα λοιπά, δεν βλέπω ότι να υπάρχει όρεξη να δημιουργηθεί κάτι νέο ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρέπει να παραδεχθούμε το γεγονό ότι σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλά σχήματα που ε, θα μπορούσαν να εγγυηθούν τέτοιου είδους πακέτα, τέτοιου είδους δέσμες μέτρων. Παναλαμβάνω, πρέπει να αφομοιώσουμε τα μαθήματα που έχουμε πάρει και ένα από αυτά είναι ότι θα πρέπει σίγουρα ε, να υπάρχει ε, ένα ταμείο εγγύησεων. Αλλά θα δούμε πώς θα πρέπει αυτό να γίνει. Σίγουρα για να λύσουμε το πρόβλημα της ρευστότητας πρέπει να κάνουμε κάτι ε, πολύ σημαντικό. Με τις κρατικές ενισχύσεις σίγουρα μπορούν να δημιουργηθούν ανισορροπίες ε, στην αγορά εργασίας, να διατραχθεί ισορροπία γιατί κάποιες χώρες θα έχουν πολύ μεγαλύτερη δημοσιονομική ικανότητα και μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο τις εταιρείε τους και άλλες χώρες λιγότερο. Επίσης ε, αυτό θα οδηγήσει και σε μελλοντική ανισορροπία. το μέσο solvency, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Θα μπορούσε να παρέμβει με αγορά ε, μετοχών, να βοηθήσει τις εταιρείε που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και χρειάζονται βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν πήραν τέτοια βοήθεια σε εθνικό επίπεδο. Να, ε, να το μελετήσουμε και αυτό. Μαζί με τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να κάνουμε μια χαρτογράφηση όλων αυτών των εργαλείων που έχουμε και είναι μακρύ ο κατάλογο, διεξοδικό ο κατάλογο, να δούμε πώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα εργαλεία. Αλλά ο στόχο μα είναι να στηρίξουμε αυτού οι οποίοι δεν έχουν βοηθηθεί. Και μιλάμε για εταιρείε που μπορούν να βγουν αλόβητε από αυτή την κρίση, μπορούν να επιβιώσουν. Οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών επίση ε, είναι πάρα πολύ σημαντικοί και ήδη από τι πρώτε κατευθυντήριε γραμμέ που δημοσιοποιήσαμε, τονίσαμε την ανάγκη να του αντιμετωπίσουμε σημαντικούς και όχι να υπάρχει αυτή η απομόνωση η καραντίνα όταν θα δέρχονταν τα σύνορα. Για κάθε τρόπο μεταφορά. ε, θέλαμε να υπάρχουν αυτά τα μέτρα προστασίας και επιμείναμε ιδίω για του εργαζόμενου στον τομέα των μεταφορών. Το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και για τον τουρισμό για τα νοσοκομεία. Μα, συγγνώμη, για, την, ε, για τους ε, δομές φιλοξενίας. Πρέπει να είναι ασφαλείς οι εργαζόμενοι στα τουριστικά επαγγέλματα ώστε να μπορέσουν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Σίγουρα. Το υποστηρίζω αυτό. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάρα πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν εργαλεία και μηχανισμοί από τους συνάδελφους μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα SURE, ένα εργαλείο για να στηρίξει ιδιαίτερα την απασχόληση της εργασίας. 100 δις σε δάνεια για το SURE ιδίω για κάποια βραχυπρόθεσμα ε, στου μηχανισμού και προγράμματα εργασίας ε, να προστατεύσουμε τους αυτοαπασχολουμένους ε, και να μην υπάρξουν απολύσεις και απόλυση οδήματο. Δεν ξέρω κατά πόσο αναρκεί αυτό. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε και είναι μια συνεχή διαδικασία όλες αυτές τι διαδικασίε και τους μηχανισμούς που εφαρμόσαμε. Επίση το Next Generation EU. Αυτό το ταμείο ουσιαστικά έχει ως στόχο την ανάκαμψη, γι' αυτό έχει προβλεφθεί. Θέλουμε εμπροστοβαρή ε, διάθεση ήδη και για του χρόνου των κεφαλαίων αυτών που ουσιαστικά θα δημιουργήσουν κέρδη και θα δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας σε πληγέντες κλάσης οικονομίας. Αυτή είναι η απάντηση μπορώ να δώσω στα διάφορα θέματα που αναφέρατε. Μιλήσατε για προστευμένες διαδικασίες. Ε, θα καταγράψω και αυτό και τα άλλα μηνύματα τα οποία ε, μου ε, μεταφέρατε στους συναδέλφους μου ώστε να μπορέσουμε να σκεφτούμε ακόμη πιο αναλυτικά για το μέλλον τώρα. Τη στρατηγική μας θα τη δείτε. Θέλουμε να υπάρξει και διαβούλευση. Θα έχετε πάρει τη στρατηγική μας για τις ε, βιώσιμες μεταφορές που θέλουμε να είναι και ανθεκτικές. Και αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δούμε το μέλλον που πρέπει να είναι ευφυές και πρέπει να είναι βιώσιμο. Θέλουμε λοιπόν ευφυείς βιώσιμες μεταφορές και όσον αφορά τον τουρισμό πρέπει να έχει βιώσιμο μέλλον και αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Υπάρχουν και πολλά περιφερειακά προγράμματα για τον τουρισμό. Το έδειξε η κρίση. Αφήνει περιφερειακό αποτύπωμα η κρίση. Και υπάρχουν αναγκαιότητες και προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη και διαφέρουν αυτές από μια περιοχή στην άλλη. Ξέρω λοιπόν ότι με τα περιφερειακά ταμεία εξασφαλίστηκε χρηματοδότης. Και τέλος, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια υγειονομική κρίση. Ο ιός, η επιδημιολογική κατάσταση ε, δεν είναι ίδια από μια χώρα στην άλλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν εμπιστοσύνη. Όσο δεν υπάρχει ε, μια αποτελεσματική θεραπεία ή ένα εμβόλιο, ο κίνδυνος ε, ελοχεύει. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Δυστυχώς, έτσι έχει κατάσταση. Και πρέπει να προσαρμοστούμε, να προσπαθήσουμε να μένουμε ασφαλείς και ταυτόχρονα να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τη δυνατότητα σύνδεσης ε, των χωρών μας και των περιοχών μας μέσω του τουρισμού και μέσω των μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. που απαντήσατε και στα σχόλια ε, των συναδέλφων με αναλυτικό τρόπο. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση. 9 το πρωί, όπως σας είπα, θα ανακοινώσω τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου ψηφοφοριών. Την Παρασκευή θα γίνει η τελική ψηφοφορία. Σας εύχομαι καλό βράδυ.